Καλημέρα σας. I have your attention, about to get started. Θα ξεκινήσουμε όπου να είναι και σήμερα οι εργασίες της Επιτροπής μας είναι ουσιαστικά ένα είδος ε, σεμιναρίου εργασία Έχουμε διοργανώσει μια ακρόαση επί δύο προτάσεων τη Κομισιόν στον τομέα τη νόμιμη μετανάστευση, Στο πλαίσιο του πακέτου για τη μετανάστευση όπως ε, το αποκαλούμε και σήμερα το πρωί θα δούμε την πρόταση για του ε, εποχιακούς εργαζομένους. Η συγητή είναι ο συνάδελφο Κλοντ Μωράε. Το μεσημέρι τώρα οι εργασίες μας θα έχουν ως αντικείμενο την πρόταση των διατερικών αποσπάσεων. Ενδιατερικών αποσπάσεων. Ο κύριος Γιακολίνο είναι ο εισηγητής. Είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους οι δύο προτάσεις σε ό,τι αφορά το επίκεντρο. Η δεύτερη πρόταση για τις ε, μεταφορές ουσιαστικά θέλει να διευκολύνει την προσωρινή μετανάστευση επαγγελματιών ε, με υψηλή δίκευση. Ενώ η πρόταση του παγικού εργαζομένου θέλει να θεσπίσει κοινά κριτήρια και διαδικασίες για μετανάστες με χαμηλή δίκευση. Έχουν όμως ένα κοινό σημείο και οι δύο προτάσεις είναι οι πρώτε προτάσει από νομική πλευράς που αφορούν την μετανάστευση, δηλαδή την νόμιμη πτυχή της μετανάστευσης μετά τη θέση και τις συνθήκες της Λισαβόνας, που πλέον συναποφασίζει βάσει αυτής το Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο για αυτές τις πολύ σημαντικές πολιτικές στον τομέα, στο, χώρο μάλλον της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ασφάλειας. Έχουμε λοιπόν την μεταναστευτική πολιτική. Εξού και η Επιτροπή μας αποφάσισε να διοργανώσει αυτή την ε, ακρόαση σήμερα για να συζητήσουμε τις δύο προτάσεις αυτές της Κομισιόν βάσει των, εργα... των εγγράφων εργασίας των εισηγητών μας παρόντες θα είναι και η Κομισιόν και το Συμβούλιο αλλά και διεθνείς οργανισμοί, κοινωνικοί εταίροι, εκπρόσωποι των κλάδων, μη κυβερνητικών οργανώσεων από το πρίσμα των νέων αρμοδιοτήτων που έχει πλέον στη θέση το Κοινοβούλιο βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας. Άρα εκπροσωπούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Και επίσης ε, εδώ θα Έχουμε συνεργασία με την Επιτροπή απασχόληση σύμφωνα με το άρθρο 50 του ιστορικού κανονισμού. Έχουμε λοιπόν προσκαλέσει ορισμένα μέλη της Επιτροπής απασχόληση και χαίρομαι που έχουν έρθει ορισμένοι εξ αυτών. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την πρωινή μας σύνοδο της εποχιακούς εργαζομένους ε, και θα δώσω το λόγο κατευθείαν στον εισηγητή μας για το θέμα αυτό, τον κύριο Κλοντ Μωράης, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το έγγραφο εργασίας του και εν συνεχεία θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν, στο Συμβούλιο, στους εισηγητής ε, από την Επιτροπή Απασχόλησης και από την Επιτροπή των Γυναικών, εφόσον θελήσουν να κάνουν κάποια σχόλια και μετά θα έχουμε ένα γύρο απόψε ανταλλαγών, συζήτηση δηλαδή. Άρα πρώτα Κλοντ Μωράης, Μάρτα Σίγκαν, την οποία θέλω και να καλωσορίσω, τη Διευθύντρια Μετανάστευσης και Ασύλου της Γενικής Διεύθυνσης Ιστορικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή θα είναι η δεύτερη ομιλήτρια. Εκεί η τρίτη ομιλήτρια, την οποία επίση καλωσορίζω, είναι η κυρία Βίβιαν Βαντάση, που είναι σύμβουλο τη ε, Μονάδα Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων τη μόνιμη αντιπροσωπεία τη Ουγγαρία, που όπω γνωρίζουμε ασκεί την Προεδρία για αυτό το εξάμεινο. Εν συνεχεία θα μιλήσει ο κύριος Σέρτζο Κοφεράτη, συγητής από την Επιτροπή Απασχόλησης και η κυρία Αντιγόνη Παπαδοπούλου, η συγγήτρια, συνάδελφός μας, η συγγήτρια για την Επιτροπή Γυναικών. Πρώτος ο κύριος Μωράης. έχετε το λόγο. Thank you, And, um, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους ε, συναδέλφους ε, που ήρθαν σήμερα εδώ. Ε, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και συναδέλφους από διάφορες οργανώσεις που θα μας παρουσιάσουν την άποψή τους οι προτάσει που έχουν κατευθεί είναι πολύ ενδιαφέρουσες μερικές φορές και αντιφατικές. Σήμερα λοιπόν έχουμε, ερχόμαστε αντιμέτωποι με διάφορα νομοθετήματα τα οποία δοκιμάζουν τις φιλοδοξίες μας ε, που είναι καταρχήν να έχουμε μια κοινή μεταναστευτική ε, πολιτική. όλη αυτή η διαδρομή μέχρι σήμερα όπου συζητάμε για την οδηγία περί εποχιακών ε, εργαζομένων σε σχέση με τους ανειδίκευτους και τους εξειδικευμένους εργαζόμενους. Όλη αυτή η διαδρομή ήταν ε, ιδιαίτερα μακριά. Το 99 τα κράτη-μέλη, ε, όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε η Επιτροπή, αλλά τα ίδια τα κράτη-μέλη ζήτησαν τη δέσμευση, αυστηρή δέσμευση, να καταρτήσουν μια κοινή μεταναστευτική πολιτική. Και με αυτόν τον τρόπο τα κράτη-μέλη θέλησαν να προβάλλουν και τα επιχειρήματα για να στηρίξουν ε, την ε, μεταναστευτική πολιτική. Γιατί προέβλεπαν ότι θα φτάναμε σε μια φάση όπου θα μιλάγαμε για τη νόμιμη μετανάστευση, όχι μόνο για τους ιδιαίτερα προσοντούχους, αλλά και για τους ανειδίκευτους εργάτες. Τα κράτη-μέλη λοιπόν κατά κάποιον τρόπο υποτίμησαν ε, τι ακριβώς εννοούμε όταν μιλάμε για κοινή μεταναστευτική πολιτική και έπρεπε να περάσουν 10-12 χρόνια μέχρι να κατατεθούν πραγματικά σοβαρές προτάσεις. Το 2005 η ανακοίνωση της ε, Κομισιόν, το σχέδιο για την ε, νόμιμη μετανάστευση κατέστησε περισσότερο σαφές τι ακριβώς έπρεπε να είναι η δουλειά μας. Εγώ λοιπόν καταθέτω σήμερα την πρότασή μου για τους εποχιακούς μετανάστες μέσα σε αυτό το πλαίσιο όλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι τη στιγμή που μιλάμε για τη νόμιμη μετανάστευση ή όταν θα φτάσουμε να μιλάμε για νόμιμη μετανάστευση, κατ' ουσία μιλάμε για πολύ ευαίσθητα θέματα που έχουν σχέση με την απασχόληση, τη ζήτηση μεταναστών εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημογραφικά επιχειρήματα, εκπαίδευση και βεβαίω ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που έχουν σχέση με την πρόταση είναι να διασφαλίσουμε ότι εκατοντάδες χιλιάδων εποχιακών εργαζομένων που αυτή τη στιγμή απασχολούνται στα κράτη-μέλη, αυτοί πρέπει να αποφύγουν την στιγμή εκμετάλλευση της οποίας είναι θύματα. Επιθυμούμε λοιπόν να ρυθμίσουμε την αγορά των εποχιακών εργαζομένων γιατί γνωρίζουμε ότι αυτή η αγορά είναι ένα κομμάτι της ευρύτερη ε, αγοράς μας. Έρχονται λοιπόν εδώ οι εργαζόμενοι, στέλνουν τα εμβάσματά τους ε, στη χώρα προέλευσης είναι άνθρωποι τους οποίους χρειαζόμαστε στις οικονομίες μας. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό, πώς μπορούμε να τους προστατεύσουμε και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε την πρόταση για τους εποχιακούς εργαζόμενους γιατί αυτή η πρόταση είναι άμεσα συνδεμένη με τον τουρισμό, τη γεωργία, με ε, ανειδίκευτους εργάτες ε, που δεν είναι κατ' ουσίαν ανειδικευτοί αλλά η δουλειά που κάνουν είναι για ανειδίκευτους εργαζόμενους. Αυτό λοιπόν είναι το υπόβαθρο. Ε, ο ΣΑ κατέθεσε την εξής, εξέφρασε την εξή άποψη ότι χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετανάστες εργαζόμενους και εποχιακά απασχολούμενους πραγματική βάση της ε, πρότασης ε, είναι επίμαχη, διότι όταν ασχολούμεθα με το θέμα της ε, μετανάστευσης, ασχολούμεθα και με θέματα απασχόλησης. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς εγκρίναμε το άρθρο 50 που προβλέπει να έχουμε συνεισηγητές από την ΛΥΜΠΕ, που είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή, και από την Επιτροπή Απασχόλησης. Παρότι λοιπόν, ε, κατά την άποψή μου, η νομική βάση είναι η σωστή, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών είναι, όπως σας είπα, η κύρια, η καθήλη αρμόδια Επιτροπή. Πρέπει λοιπόν να αναλάβει το ρόλο του συνεισηγητή και να ε, συμβάλλει και αυτή ιδιαίτερα για το άρθρο 16 που ασχολείται με την ε, μεταχείριση των εργαζομένων. Και για αυτόν τον λόγο εγώ συνεργάστηκα στενά με τον συνεισηγητή κύριο Κοφεράτη, ο οποίος θα είναι συνεισηγητής από την Επιτροπή Απασχόλησης. Συνεργάστηκα στενά και με την κυρία Αντιγόνη Παπαδοπούλου, η οποία κατέθεσε τη γνωμοδότηση εκ μέρους της Επιτροπής Γυναικών. Όμως, ε, όπως ε, σας είπα, συνεργαστήκαμε στενά όλες αυτές οι επιτροπές για να διασφαλίσουμε ότι η ουσία του θέματος, οι εποχιακοί εργαζόμενοι που έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί πρέπει να ε, βρίσκονται σε μια αγορά εργασίας όπου βεβαίως δεν υφαρπάζουν την δουλειά άλλων, αλλά και οι ίδιοι δεν καθίστανται θύματα εκμετάλλευσης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνο λοιπόν που επιθυμώ να σας ε, παρουσιάσω σήμερα, ε, έχω μόνο 10 λεπτά για να μιλήσω, δεν θα παρουσιάσω όλες τις πτυχές του θέματος, θα παρουσιάσω ορισμένα βασικά στοιχεία της έκθεσης αυτής. Πρώτον, όσον αφορά την επικουρικότητα, η διαδικασία της κίτρινης κάρτας δεν αναφέρεται στην πρόταση αυτή, αλλά υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που ανέφεραν ότι το θέμα της επικουρικότητας είναι σημαντικό. Ότι το θέμα των εποχιακών εργαζομένων είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να εξετάζεται αποκλειστικά σε επίπεδο κρατών μελών. Εξετάζοντας λοιπόν την πρόταση αυτή, αυτό το στοιχείο το λαμβάνω ιδιαίτερα υπόψη μου. Γιατί το στοιχείο αυτό αναφέρεται στο διαρκέ θέμα της μετανάστευση, το οποίο είναι πράγματι ευαίσθητο θέμα. Ε, τα κρατημέλη που επιθυμούν, υπάρχουν κρατημέλη που επιθυμούν να το αντιμετωπίσουν μόνα τους ε, και άλλα που γνωρίζουν ότι η μετανάστευση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι θα αποκτήσει υπεραξία. Η πρόταση θέλει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου οι εποχιακά εργαζόμενοι θα έρχονται εδώ, θα κάνουν τη δουλειά τους, ε, ε, θα εκτελούν ε, τα χρέη της κυκλικής μετανάστευσης, δηλαδή εδώ και μετά πίσω στην πατρίδα τους. Όμως εργάζονται ικανοποιητικά, με ικανοποιητική αμοιβή, στέγαση και μπορούν να παραμένουν εδώ μέχρι έξι μήνες. Η πρόταση ε, που μερικές φορές αποκλήθηκε και φιλόδοξη δεν είναι και τόσο φιλόδοξη με την έννοια να προσποιείται ότι οι εποχιακά εργαζόμενοι είναι κάτι που δεν είναι. Οι εποχιακά εργαζόμενοι απασχολούνται στη γεωργία, στον τουρισμό που ενέχουν αυτό το εποχιακό στοιχείο. Οφείλουμε λοιπόν να γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι, πρέπει να ασχοληθούμε με τους τομείς που πραγματικά παίζουν ρόλο και όχι εκείνους που ενδέχεται να αποκλειστούν γιατί δεν ενέχουν αυτό το στοιχείο της εποχικότητας. Ασχολούμεθα λοιπόν με ένα σημαντικό στοιχείο του πακέτου της νόμιμης μετανάστευσης και δεν προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν προβλεπόταν ε, στην πρόταση. Επιθυμούμε λοιπόν ισχυρότερη προστασία για ε, εποχιακά εργαζόμενες που είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης, τα κριτήρια εισόδου τους, ε, αυτά ε, θα είναι συνάρτηση του συμβολέου που υπογράφουν. Όσον αφορά τη στέγαση, στην πρότασή μας ο εργοδότης υποχρεούται να ε, αποδείξει ότι ο εποχιακά εργαζόμενος θα έχει σωστή στέγαση κατά τη διάρκεια της παραμονής του. Επίσης υπάρχουν, υπάρχει και κάποιος μηχανισμός κυρώσεων. Τίθεται και το θέμα της ίσης μεταχείρισης. Η πρόταση προβλέπει μεταχείριση με τους εθνικούς ε, εργαζόμενους. Ε, αναφέρομαι στο άρθρο 16. Βεβαίως εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι ο ορισμός του άρθρου 16 δεν είναι ικανοποιητικός, αρκετά ισχυρός ε, για να υπάρχει ίση μεταχείριση. Και αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο της πρότασης, ότι συζητήσαμε με τους συναδέλφους μας από την Επιτροπή Απασχόλησης ε, και πολλοί από εσάς ε, εδώ εκπροσωπούν την οργανωμένη απασχόληση και γνωρίζουν ότι η ίση ε, μεταχείριση είναι εκείνη που διασφαλίζει την αρμονία στην αγορά εργασίας και δεν καταλήγουμε σε μια κατάσταση όπου ο ένας εργαζόμενος να υφαρπάζει την δουλειά ε, του άλλου. Ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπάρχει αρκετή νομολογία σε σχέση με την ε, οδηγία που έχει θεσπιστεί. Οι εποχιακά εργαζόμενοι ορίζονται λοιπόν στην πρόταση αυτή. Αν έχω άλλα πέντε λεπτά θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ και σε πολλές άλλες προτάσεις. Βέβαια δεν σημαίνει αυτό ότι θέλω να μπω σε λεπτομέρειες στη δική μου την πρόταση. Απλά μου είπατε ότι πρέπει να κρατήσω τα δέκα λεπτά. Παρακαλώ λοιπόν ε, να σημειώσετε ε, ότι, ερωτήσεις έχετε και κατά τη να τις θέσετε. Ο ορισμό του εποχιακά εργαζόμενου, αυτό είναι κοινή αρμοδιότητα τη επιτροπή επασχόληση και τη επιτροπή ε, Πολιτικών Ελευθεριών. Ε, εάν δεν υπάρχει ορισμό, δεν υπάρχουν και αποφάσει και επιθυμούμε να οριστεί σαφέστερα τι ακριβώ είναι ο εποχιακά εργαζόμενο. Και εδώ φτάνω στην παρατήρηση που έκανα σχετικά με του τομεί ε, που πλήττονται και το πώ ακριβώ καλείται να λειτουργεί ο εποχιακά εργαζόμενο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τομεί που ενδέχεται να αποκλειστούν γιατί το συζητάμε αυτό στο έγγραφο εργασίας, παραδείγματος χάρη ο τομέας των κατασκευών ε, και άλλοι τομείς που δεν είναι εποχιακοί, αυτά αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της έκθεσης που, την οποία ήδη συζητάμε με εκπροσώπους αυτών των κλάδων. Όσον αφορά το θέμα της κυκλικής μετανάστευσης ε, όταν κατατέθηκαν οι προτάσεις του Τάμπερη, η ιδέα ότι οι νόμιμοι εργαζόμενοι, εξειδικευμένοι ή ανειδίκευτοι, έρχονται εδώ ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απορροφώνται από την κοινωνία, αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχει συζητηθεί πολύ συχνά. Η συμβολή των ε, εποχιακά εργαζόμενων με την έννοια ότι αυτοί στέλνουν εμβάσματα στις ε, χώρες προαλήψης τους που είναι πολύ συχνά αναπτυσσόμενες και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Υπάρχουν ΜΚΟ που επιθυμούν να εξεταστεί το θέμα αυτό και να εξεταστεί η συμβολή των εργαζομένων, να εξεταστούν επίσης και οι συνθήκες διαβίωσής τους. Το επόμενο θέμα, πολύ σημαντικό στην πρόταση, είναι τα κριτήρια εισόδου αυτών των εργαζομένων. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θα εξτάσει κατά κύριο λόγο το θέμα. Θα εξετάσουμε ε, τα συμβόλαια, ε, τις, τους όρους διαβίωσης, ε, τα έγγραφα που πρέπει να έχουν εργαζόμενοι, ε, την ασφάλεια ασθενείας τους, ε, χρήματα που ε, πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι όταν μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον όγκο, τον αριθμό εργαζομένων που θα δεχτούμε και αυτό είναι σημαντικό. Η δυνατότητα του εργαζομένου να αλλάξει εργοδότη και να μην γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευση, να μπορεί να διαμαρτυρηθεί. Οι εποχιακά εργαζόμενοι πολύ συχνά ζουν κάτω από ιδιαίτερα αντίξωε, ακραίε συνθήκε, όπω είδαμε στην Ιταλία, στο Λοζάρνο, όπου οι άνθρωποι αυτοί κατ' ουσίαν ζουν στα δάση. Ε, φτάνουμε σε καταστάσεις όπου εποχιακά εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται βέβαια και με καλύτερο τρόπο. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις περιπτώσεις της στιγμής εκμετάλλευσης, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα κατώτατο όριο που ισχύει για όλους αυτούς τους εργαζόμενους. Θα δούμε τις άδειέ τους, τα κράτη-μέλη καλούνται ε, να δίνουν τις ε, πληροφορίες ε, για τον τόπο διαμονής τους. Θα εξετάσουμε όλο το θέμα της διαβίωσής τους, τα ικανοποιητικά κριτήρια διαβίωσης για τους εποχιακά εργαζόμενους και τέλος όσον αφορά τις κυρώσεις και τις ε, διαμαρτυρίες όπως σας είπα πολύ εύκολα μπορεί κανείς να πει ότι ένας εποχιακά εργαζόμενος μπορεί να διαμαρτυρηθεί όμως αν δεν είναι συνδικαλισμένος και αν αισθάνεται ότι είναι αντικείμενο εκμετάλλευση είναι πολύ δύσκολο να διαμαρτυρηθεί γιατί ε, αν μπορεί να μην βρει εργασία. Πολλές φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι με σκληρές καταστάσεις. Βεβαίως αυτό αφορά του εποχιακά εργαζόμενου. και επιθυμούμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου θα υπάρχει ένα, ε, υπάρχουν τα βασικά, ε, οι βασικές προδιαγραφές. Θέλουμε λοιπόν να εξετάσουμε ε, και το λόγο των μεσαζόντων και των πρακτορείων προσφορά εργασία. Θα καταλήξω στο εξή οι εποχιακά εργαζόμενη η οδηγία η σχετική ε, είναι επίμαχη όπως σας είπα, απλά και μόνο γιατί οφείλουμε να κατανοήσουμε το κύριο και κέριο θέμα της ίσης μεταχείρισης. Πρέπει επίσης να κατανοήσουμε την θέση των κρατών μελών, ευαισθησίες που υπάρχουν σχετικά με την αγορά εργασίας για μετανάστες. Αλλά τελικά πρέπει να γνωρίζουμε ότι αν τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που ζήτησαν την κοινή μεταναστευτική πολιτική, γιατί εκείνα το ζήτησαν, ε, βέβαια υπάρχουν κράτη-μέλη με τελείω διαφορετική πολιτική προσέγγιση, αλλά δέχτηκαν όλοι ότι η μετανάστευση είναι ένας μεγάλος πόρος ε, προσφοράς, ε, μια πηγή προσφοράς για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θεωρούμε ότι εδώ είμαστε σε μια κοινότητα αξιών, τότε ο τρόπος με τον οποίο μεταχειριζόμαστε τους εργαζόμενους αυτούς και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν εκείνοι στην αγορά είναι καθοριστική σημασία. Είναι λοιπόν ένα χρήσιμο βήμα προς τα εμπρός στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης και ελπίζω ότι όλοι σας θα έχετε μία θετική ε, προσέγγιση όσον αφορά στις ε, τροπολογίες ε, και κυρίως όσον αφορά στις λεπτομέρειες που σας παρουσίασα. Ευχαριστούμε πολύ, Κλόντ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή που παρουσίασε το θέμα. Έχει περισσότερο χρόνο, 10 με 20 λεπτά ο εισηγητής, αλλά προτείνω από εδώ και στο εξής να προσπαθήσουμε να αρκεστούμε σε 7 με 8 λεπτά για τις υπόλοιπες ομιλίες, ώστε να υπάρξει χρόνος και για συζήτηση. Και να περάσουμε και στο επόμενο σημείο μας, που είναι ουσιαστικά η εποχιακοί εργαζόμενοι. Τώρα δίνω το λόγο στην Μάρτα Σίγκαν, που είναι η Διευθύντρια Μετανάστευσης και Ασύλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την οργάνωση αυτής της δημόσιας ακρόασης για δύο πολύ σημαντικές προτάσεις που εφαρμόζουν και συμπληρώνουν την εφαρμογή του Σχεδίου Πολιτικής για την Νόμιμη Μετανάστευση του 2005. Όπως υπόθηκε, θα συζητήσουμε σήμερα τους εποχιακούς εργαζομένους και, τους, και τις ενδοεπηρεσιακές ε, μεταθέσεις, όπως υπόθηκε και στα εισαγωγικά σχόλια του Προέδρου. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά. Είναι οι πρώτες προτάσεις που εγκρίνονται μετά την έναρξη ισχύω της συνθήκης της ε, Λισαβόνας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που παρίσταμε σε μια συνεδρία σαν τη σημερινή, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, όλων των εταίρων και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για μας να καταλάβουμε ποιες είναι οι ανησυχίες, οι απόψεις, οι αμφιβολίες, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε και εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτά που θα ακούσουμε για να προωθήσουμε την διαδικασία λήψης αποφάσεών μας. Μία σκέψη για τη μετανάστευση Γνωρίζουμε ότι είναι ένα γεγονός. Κάθε μέρα λαμβάνει χώρα. Συμβαίνουν ε, πολύ έκτακτα περιστατικά σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης και του κόσμου. Κάθε μέρα, σε κάθε στιγμή, ερχόμαστε αντιμέτωποι με το ζήτημα της μετανάστευσης. Νομίζω λοιπόν ότι η καλή διαχείριση, η ολοκληρωμένη διαχείριση της μετανάστευσης ε, είναι μια επιταγή για τις εργασίες μας και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε μια καλή και ολοκληρωμένη διαχείριση του φαινομένου της μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις σχέσεις μας με τις τρίτες χώρες. Δεν, είναι πάντοτε, δεν αφορά μόνο τις περίοδους κρίσης. Προσπαθούμε να σκεφτούμε και πιο μακροπρόθεσμα για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια βιώσιμη προσέγγιση για το θέμα της μετανάστευσης. Θα αναφερθώ αμέσως ε, στην οδηγία για, τα, για τους εργαζομένους, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο. Τα βασικά στοιχεία τα παρουσίασε ο εισηγητής, αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πολύ σύντομα το ιστορικό της πρότασης. Ο βασικός στόχος της πρότασης αυτής είναι να μας βοηθήσει σε μια απλή σε ένα απλό, ομαλό και ελκυστικό ε, πλαίσιο για την κατηγορία των εργαζομένων ε, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι θέλουμε να εξασφαλίσουμε το πλαίσιο αυτό ώστε να μπορούν ε, να εργαστούν σε προσωρινή βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ παράλληλα διασφαλίζουμε ότι η κατηγορία αυτή προστατεύεται ε, επαρκώς ε, ενάντια στην εκμετάλλευση. Είναι η πρώτη πρόταση που αφορά τους εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης ε, μετά από το πακέτο που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την νόμιμη μετανάστευση και μετά από την οδηγία για τους εργαζομένους της ειδίκευσης. Τώρα, για ποιο λόγο θεωρήσαμε απαραίτητη την παρουσίαση της πρότασης αυτής. Υπάρχει πολύ μεγάλο, μεγάλη ανάγκη για ε, εποχιακά εργαζομένους τρίτων χωρών. Ε, χρειαζόμαστε χώρες, ε, εργαζομένους από τις τρίτες χώρες, στην δασοκομεία, στη γεωργία, σε τέτοιου είδους τομείς και όλο και λιγότεροι εργαζόμενοι είναι διαθέσιμοι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τέτοιου είδους εργασίες. Βλέπουμε λοιπόν από την πείρα μας ότι οι άνθρωποι αυτοί θα χρειαστούν κάποια προστασία μερικές φορές ε, έχουν, ε, έρχονται αντιμέτωποι με συνθήκες εκμετάλλευσης και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να καταπολεμήσουμε. Τα πρόσφατα γεγονότα στη Μεσόγειο δείχνουν επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρεμποδίσουμε την ε, λαθρέα μετανάστευση, ανοίγοντας διόδους για νόμιμη μετανάστευση. Και αυτή είναι μία από τις καλύτερες μεθόδους για να μπορέσουμε να μειώσουμε την παράνομη μετανάστευση. Ποια είναι τα βασικά ωφέλη τώρα της ε, πρότασης που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρότασή μας βασίζεται στην εδραίωση μιας γρήγορης ομαλής διαδικασίας για την εισδοχή ε, των ε, εποχιακών εργαζομένων, ώστε να μπορούν να είναι διαθέσιμοι πολύ πιο γρήγορα στις ευρωπαϊκές οικονομίες όταν τις χρειάζονται. Αυτό έχει προβλεφθεί στο σχέδιο νομοθετήσματός μας, δηλαδή ότι τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για τον ορισμό του αριθμού των εργαζομένων που ε, θα δεχθούν. Αυτό αναφέρεται στο κείμενό μας, δηλαδή η αυτονομία του κράτους μέλους, η ελευθερία του να ε, αποφασίσει τον αριθμό των εργαζομένων που θα ε, δεχθεί, αναφέρεται ευθαρσός. Επίσης θέλουμε να εδραιώσουμε μια γρήγορη διαδικασία, μια ταχεία διαδικασία, ισότιμη σε όλα τα κράτη-μέλη και θα δώσει τη δυνατότητα ε, μια καλή, μιας καλύτερης διαδικασίας ε, σε όλα τα κράτη-μέλη, ισότιμης διαδικασίας, ε, πρόσληψης εποχιακών εργαζομένων. Προτείνουμε απλούς κανόνες εισδοχής, που θα έχει ως αποτέλεσμα νόμιμα εργαζομένους ε, εποχιακούς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχει μια πολύ σαφή σχέση εδώ με την ε, οδηγία επιβολής κυρώσεων στους εργοδότες Ελπίζω ότι την, διαδικασ... Ε, προθεσμία μεταγραφής της οδηγίας που είναι ο Ιούλιος του τρέχοντος ε, θα τη σεβαστούν τα κράτη-μέλη γιατί θα είναι πάρα πολύ σημαντική για να παρακολουθήσουμε πώς εφαρμόζονται τα νομοθετήματα αυτά στα κράτη-μέλη. Τώρα, το στοιχείο σταθεροποίησης ε, και νομιμοποίησης της κατάστασης των εργαζομένων Πρώτα απ' όλα έχουμε τις νομικές διατάξεις ε, που εφαρμόζονται για τις συνθήκες εργασίας. Αναφέρονται σαφώς. Οι εργοδότες ε, πρέπει να αποδείξουν ότι οι εποχικά εργαζόμενοι θα έχουν την κατάλληλη στέγαση κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στη χώρα. Οι εποχιακοί εργαζόμενοι επίσης ε, θα έχουν στη διάθεσή τους ένα μηχανισμό καταγγελίας ο οποίος έχει σχεδιαστεί για την καλύτερη ε, εφαρμογή της νομοθεσίας. Και όπως υπόθηκε και από τον εισηγητή, η, εφαρμογή, η παρακολούθηση της εφαρμογής ε, του μηχανισμού αυτού είναι πάρα πολύ σημαντική. Τώρα, για την ίδια την οδηγία και την πρόταση το πώς δηλαδή οι εποχιακά εργαζόμενοι θα στεγάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και αυτό μια συμβολή στην ενίσχυση της κυκλικής μετανάστευσης που είναι μια πάρα πολύ σημαντική έννοια και την προωθούμε στο πακέτο της ε, πολιτικής μετανάστευσης. Η κυκλική μετανάστευση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και άλλων χωρών ε, θα παρεμποδίσει την παραπάνω διαμονή των εποχιακά εργαζομένων, ε, αλλά θα ε, έχει τη δυνατότητα μεταφοράς ε, δεξιοτήτων και γνώσεων προς τις τρίτες χώρες. Τώρα, τι θέλουμε να κάνουμε για να προχωρήσει όλη η διαδικασία. Ελπίζουμε να προοδεύσουμε για αυτό το ζήτημα σύντομα όλες οι συζητήσεις που είχαμε με τους εταίρους και όλη η διαδικασία την οποία θα παρουσιάσει ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου σε λίγο. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ καλέ οι συζητήσεις μας για να μπορέσουμε να επισπεύσουμε την έγκριση της συγκεκριμένη πρότασης. Ελπίζω να μπορέσουμε να ακούσουμε σήμερα τα σχόλιά σας, τα ερωτήματά σας, ε, να ε, τα ενστερνιστούμε για να μπορέσουμε να επισπεύσουμε τη διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι θέλει να πράξει. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω, όπως είπε και ο εισηγητής, για το θέμα της επικουρικότητας. Το οποίο ήταν ιδιαίτερος ε, αισθητό κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Είχαμε διαφορετικές απόψεις από τα εθνικά κοινοβούλια. Κάποια ε, σχόλια ήταν αρνητικά, κάποια ήταν θετικά και ήταν επίσης μια πάρα πολύ σημαντική εμπειρία για την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων η έγκριση της συγκεκριμένης πρότασης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πολύ χαρά θα ακούσω τα σχόλιά σας και θα απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σίγκαν. Η κυρία Βίβιεν Βαντάση από τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ουγγρικής Προεδρίας της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν κάποιοι χρονικοί περιορισμοί γιατί έχουμε ακόμη δύο παρεμβάσει και χρειαζόμαστε και χρόνο για τη συζήτηση. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και που μου δίνετε το λόγο. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. μέρους της Ουκρικής Προεδρίας θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για την ακρόαση που έχει διοργανώσει. Η Ουγγρική Προεδρία με τη σειρά τη προσδίδει και αυτή πολύ μεγάλη σημασία σε ευρείε διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους φορείς και βέβαια και στην στενή συνεργασία με τους συνομοθέτε, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ουγγρική Προεδρία και ελπίζουμε να μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε αυτή τη συζήτηση στο πλαίσιο του Συμβουλίου σε σχέση με αυτά τα δύο στοιχεία του πακέτου μέτρων για την νόμιμη μετανάστευση. Σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη πρόταση για τους εποχιακούς εργαζομένους, ο στόχος είναι να υπάρξει ένα απλό και κατά το δυνατόν ομαλό σύστημα το οποίο θα μπορεί να εφαρμοστεί ε, στα κράτη-μέλη να εφαρμοστεί πρακτικά, να είναι ένα ευέλικτο σύστημα το οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών. Φυσικά πρέπει να έχουμε υπόψη βέβαια και τα δικαιώματα των εποχιακών εργαζομένων που πρέπει να γίνουν σεβαστά. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έγγραφο εργασία του και ελπίζω πραγματικά η συζήτηση να δώσει τροφή για ε, συζήτηση και για προβληματισμό. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω πώς έχει η κατάσταση στο Συμβούλιο και θα μου επιτρέψετε να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα, τα ουγγρικά. Στη διάρκεια της ε, Ουγγρικής Προεδρίας είχαμε εντατικές συζητήσεις ε, σε σχέση με το έργο που ξεκίνησε η Βελγική Προεδρία Έχουμε λοιπόν αυτές τις διαπραγματεύσεις με όλους ε, τους ειδικού και σημειώσαμε πρόοδο σε κάποια ζητήματα. Νομίζω ότι η θέση των κρατών μελών ε, πλέον είναι πιο ξεκάθαρη, έχει αποκρισταλωθεί κατά κάποιο τρόπο. Ο κύριος Μωράης αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφεραν ότι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων ε, συνεχώς ακουγόταν η έννοια και η αρχή της επικουρικότητας από τα κράτη-μέλη. Και αυτό πραγματικά είναι ένα θέμα για εμάς. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο της πρότασης. Υπάρχουν πολύπλοκα ζητήματα που σχετίζονται και με τον κοινωνικό τομέα και με τα εργασιακά δικαιώματα. Η ομάδα εργασίας κυρίως των κοινωνικών υποθέσεων είναι αρμόδια για αυτά τα θέματα και στο πλαίσιο αυτής της ομάδας εργασίας ήδη έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις και η Επιτροπή θα υποβάλει γνωμοδότηση στην καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή δηλαδή την ομάδα εργασίας ε, του Συμβουλίου για θέματα μετανάστευσης. Υποθέτω ότι η διαδικασία που ακολουθείτε σε εμά είναι παρόμοια με αυτή του Κοινοβουλίου, δηλαδή Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και Επιτροπή Απασχόλησης που συνεργάζονται για το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά ζητήματα, μπορώ να σας πω ότι ήταν έντονες και εντατικές οι συζητήσεις, ε, θα συνεχιστούν για κάποιο ακόμη χρονικό διάστημα. Και μπορώ να σας πω επίσης ότι αυτό το οποίο πρώτα απ' όλα εξετάζουμε είναι η άδεια διαμονή που δεν πρέπει να υπερβαίνει του ε, τρει μήνε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και σε σχέση με αυτό θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι είχαμε συζητήσει με του εμπειρογνώμονε μα για θέματα θεώρηση ε, και η βασική πρόκληση είναι αυτή η οποία αφορά διαμένοντε είτε για μικρό χρονικό διάστημα είτε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διότι διαφέρουν οι κανονισμοί στα κράτη-μέλη και θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να του εναρμονίσουμε. Έχουμε έχουμε βέβαια θέσει κάποιου στόχου. Η Ουγγρική Προεδρία, λαμβάνοντα υπόψη του στόχου αυτού, θεωρεί ότι σε ό,τι αφορά του εποχιακού εργαζομένου θα πρέπει να του ε, ε, αναγνωρίζουμε τα ίδια ακριβώ δικαιώματα ανεξαρτήτω του διαστήματο παραμονή του. Και βάσει αυτή τη αρχή προσπαθούμε να εργαστούμε και να επιτύχουμε μια ικανοποιητική ισορροπία. Θα ήθελα επίση ε, να σα ενημερώσω για κάτι άλλο πολύ σημαντικό ε, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Είναι ο ορισμός του εποχιακού εργαζομένου. Ο κύριος Μωράης αναφέρθηκε στον ορισμό όπως και ο πρόεδρος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και υπάρχει και το ζήτημα του προσδιορισμού της περίοδου εργασίας ενός εποχιακού εργαζομένου. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στο Συμβούλιο, αποκλίνουν η μία από την άλλη γιατί διαφέρουν και εθνικές ε, συνθήκες από τη μια χώρα στην άλλη ή υπάρχουν ίσως διαφορετικά συστήματα από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Και σε ό,τι αφορά το πώς ορίζουμε την εποχή και τον εποχιακό εργαζόμενο υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Επίσης, διαφορές διαπιστώνουμε και σε ό,τι αφορά τον τομέα που απασχολεί εποχιακούς εργαζομένους στο ένα κράτος μέλος ή στο άλλο. Γίνεται λόγος ε, για διαμονή έξι μηνών στο έγγραφο. Κάποια κράτη-μέλη θεωρούν ότι είναι πολύ μεγάλο αυτό το χρονικό διάστημα, κάποια άλλα κράτη-μέλη θεωρούν ότι είναι πολύ μικρό. Άρα πρέπει να εξεύρουμε τη σωστή ισορροπία. Και πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη τις εθνικές πρακτικές που ισχύουν. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της μετανάστευσης μπορώ να σας πω ότι συζητείται και ένα άλλο θέμα και συγκεκριμένα κατά πόσον οι ετούντες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσει τους ε, στην επικράτεια ενός κράτους μέλους της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο διαμένουν. Και επίσης το θέμα των ε, επαρκών συνθήκων, των κατάλληλων συνθήκων διαβίωσης. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πώς όμως ορίζει κανείς την επαρκή διαβίωση, ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης ή πώς ορίζει κανείς ένα μη υπερβολικό επίδομα, non-excessive allowance. Σε κάποια κράτη-μέλη εκφράζονται ανησυχίες ότι στο κείμενο ο εργοδότης είναι αυτός ο οποίος είναι αρμόδιος να εξασφαλίσει αυτό το ε, παρκές επίπεδο διαβίωσης και στα κράτη-μέλη εκείνα που δεν ε, ε, υπάρχουν μάλλον άλλα κράτη-μέλη στα οποία όχι ο εργοδότης αλλά ο ίδιος ο εργαζόμενος πρέπει να φροντίσει για το κατάλημά του. Και υπάρχει το εξή θέμα. Πώ μπορεί να αποδείξει ένα εργοδότη ότι διαβεί υπό επαρκεί συνθήκε ένα εργαζόμενο ε, δικό του. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια άλλα ζητήματα εν συντομία, κυρίε και κύριοι, θέματα τα οποία θα εξακολουθήσουμε να συζητούμε στο πλαίσιο τη Προεδρία μα. Και βέβαια πρέπει να σα πω ότι συνεργαζόμαστε στενά με την Κομισιόν, αλλά και με την επερχόμενη Πολωνική Προεδρία που έπεται. Και παρακολουθούμε τις διαπραγματεύσεις και τις συζητήσεις εδώ στο Κοινοβούλιο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είμαστε ανοιχτοί επίσης να ακούσουμε τα σχόλια όλων των ε, υπόλοιπων ενδιαφερομένων φόρων που παρίστανται εδώ σήμερα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Προτείνω λοιπόν ε, να ακούσουμε για πέντε λεπτά τους εισηγητές από την Επιτροπή Απασχόληση και μετά από ε, την Επιτροπή Γυναικών. Τον λόγο έχει ο κύριος Σέρτζο Κονφεράτη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο θέμα που κατά την άποψή μου πρέπει να έχουμε κατά νου γιατί δεν είναι δεδομένο αντίθεση με ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί είναι η σημασία που έχει η οδηγία αυτή. Πολλοί πιστεύουν ότι η οδηγία είναι άχρηστη και μόνο αυτό, αλλά πολλοί πιστεύουν ότι είναι και αντιπαραγωγική. Εγώ όμως πιστεύω ότι είναι καθοριστική σημασία για να ορίσουμε τα δικαιώματα τόσων πολλών εργαζομένων. Η εποχική εργασία μεταξύ άλλων έχει ως στόχο να αυξήσει την ε, εργασία γενικότερα γιατί κατά τα παρελθόντα έτη η εργασία αυτή υπήρχε κυρίως στον γεωργικό τομέα και τα τελευταία χρόνια η εποχική εργασία εμφανίζεται κυρίως στον τριτογενή τομέα δηλαδή ε, σε όλα, όλες, όλους τους κλάδους και όλες τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με τον τουρισμό και τις διακοπές. Καταλαβαίνετε πολύ καλά γιατί υπήρξε αυτή η αύξηση. Γιατί στη Γεωργία ένα μεγάλο κομμάτι της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων ήδη τώρα λαμβάνει χώρα από εποχικούς εργαζόμενους. Όσον αφορά τον τουρισμό έχει αλλάξει ο τρόπος διαβίωσης και γι' αυτό το λόγο η ζήτηση, η τουριστική ζήτηση στην Ευρώπη αυξάνεται και θα αυξηθεί περαιτέρω. Κατόπιν τούτου ε, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια οδηγία όσο το δυνατόν σαφέστερη. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να εντοπίσουμε τους τομείς εφαρμογής. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ πρέπει να υπάρχει κάποιο στοιχείο ευελιξίας. Η Ευρώπη είναι κάτι το πολύ ευρύ και μακρύ αν θέλετε οι εποχές ε, ορίζονται με την έννοια των δύο-τριών μηνών, όμως η εποχική εργασία ε, δεν είναι δύο-τριών μηνών, γιατί ας πούμε η εποχή στη Φιλανδία είναι διαφορετική από ό,τι σε άλλο κράτος. Θεωρώ λοιπόν ότι θα ήταν χρήσιμο να ορίσουμε το κατώτατο όριο και μετά όσον αφορά τη διάρκεια ή όσον αφορά μεμονωμένους κλάδους, να αφήσουμε εκεί τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να έχουν εποχές μεγαλύτερης διάρκεια, αυτό βέβαια θα προβλέπεται στην οδηγία και να προσθέσουν και άλλους επιπλέον κλάδους. Το δεύτερο θέμα, τρίτο αν θέλετε, γενική φύση που θέλω να, να θέσω είναι το εξή. Μιλάμε για ίση μεταχείριση. Όμω, ε, ίση μεταχείριση δεν σημαίνει μόνο ίδια αμοιβή για ίδια εργασία. Μιλάμε για τι γενικότερε συνθήκε εργασία. Ασφάλεια, παραδείγματο χάρη, εσωτερικά δικαιώματα όταν κανεί εργάζεται και φτάνουμε μέχρι εκείνο που ε, συνθέτει τα υλικά αγαθά του εργαζομένου, εκείνου που παρέχει εργασία. Άρα δηλαδή η συμμεταχείριση αυτό είναι πολύ ευρύτερο από αυτό που εννοούμε σήμερα γιατί εδώ συμπεριλαμβάνονται και άλλα δικαιώματα που δεν έχουν σχέση άμεσα με την αποζημίωση. Το εργαλείο εκείνο το οποίο ε, ρυθμίζει τις ε, ενιαίες προδιαγραφές και ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η ενιαία ρύθμιση επιθυμεί και τη διαφάνεια γιατί υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες και αυτό αναπόφευκτα οδηγεί στο κοινωνικό ντάμπινγκ. Το εργαλείο λοιπόν το οποίο πρέπει να ρυθμίζει την ίση μεταχείριση δεν μπορεί να είναι άλλο παρά οι συλλογικές συμβάσεις οι συλλογικές συμβάσεις ε, ποικίλουν στα κράτη-μέλη και πρέπει να αναγνωριστούν όλες οι διομορφίες των συλλογικών συμβάσεων. Υπάρχουν ε, συλλογικές συμβάσεις που ρυθμίζουν συγκεκριμένους κλάδους και υπάρχουν άλλες που ρυθμίζουν γενικότερα όλες τις εργασίες ε, που λαμβάνουν χώρο. Και αυτά πρέπει να τα ρυθμίσει η οδηγία. Κατόπιν, ένα άλλο θέμα είναι η έλεγχη και οι κυρώσεις. Αυτά είναι πολύ σημαντικά για να αποφύγουμε εκφυλιστικά φαινόμενα, γιατί δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όταν μιλάμε για εποχική εργασία, πολύ συχνά μιλάμε για και παράνομη εργασία, γιατί ε, είναι πολύ πιο δύσκολο να ελεγχθεί η εποχική εργασία. Έλεγχοι λοιπόν και κυρώσεις, έλεγχοι και κυρώσεις είναι καθοριστική σημασία για την ποιότητα της μελλοντική εποχικής εργασίας. Αν δεν υπάρχουν έλεγχοι και κυρώσεις, θα, γίνει κάποια πρόοδος, αλλά όχι η ευκταία πρόοδος στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν πολύ επικίνδυνα φαινόμενα ε, που έχουν σχέση με την παράνομη εργασία. Εγώ λοιπόν ότι θα ήταν χρήσιμο και αυτή την πρόταση καταθέτω να υπάρχει μια μεταβατική φάση. Δηλαδή όταν η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ θα υπάρχει στην Ευρώπη ένα σημαντικός αριθμό παράνομων εργαζομένων. Και αυτό πρέπει να ρυθμιστεί. Να ρυθμιστούν οι σχέσεις ε, των μελλοντικών εποχικών εργαζομένων, ε, γιατί αν δεν ρυθμιστεί αυτό πιστεύω ότι είναι λάθο. Να υπάρχει λοιπόν μια μεταβατική περίοδος που θα επιτρέπει σε αυτούς που ήδη βρίσκονται στην Ευρώπη να, να έχουν μια κάποια αναγνώριση, γιατί αλλιώς θα ε, μπλακούμε σε ένα φαύλο κύκλο που που θα έχει επιπτώσεις τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κοφεράτη. Δίνω το λόγο τώρα στην συνάδελφό μας, ε, την κυρία Αντιγόνη Παπαδοπούλου, που είναι η συγγήτρια για την Επιτροπή Γυναικών για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Τώρα, μια κοινή μεταναστευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στι μέρε μα μια αναγκαιότητα. Η εποχική εργασία ε, έχει αυξηθεί σημαντικά σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι σημαντικό να έχουμε ενώπιον μα μια πρόταση οδηγία, γιατί είναι ένα, ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Η πρόταση στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών για την ειδική κατηγορία Τη της προσωρινής μετανάστευσης και ο στόχος είναι να υπάρχουν δίκαιοι και διαφανείς κανόνες για την εισδοχή και διαμονή εποχιακών εργατών αλλά και κίνητρα και διασφαλίσεις ώστε η προσωρινή διαμονή να μην γίνεται μόνιμη και αφού θα επιβάλλονται ελάχιστα πρότυπα, κυρώσεις και μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες. Από την οπτική γωνιά της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων τονίζουμε ότι πρέπει οι γυναίκε που αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό ανάμεσα στου εποχικού εργάτε, πραγματικά να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη ευαισθησία γιατί οι γυναίκε είναι ευάλωτε, αρκετέ προέρχονται από φτωχέ χώρε, αναλφάβητε, με χαμηλό βιωτικό επίπεδο έχουν παιδιά είναι λεχόνες είναι εγκυμονούσε. Πολλέ φορέ όταν εργάζονται σε μια ξένη χώρα έχουν να αντιμετωπίσουν εμπόδια προκαταλήψει και στερεότυπα πέραν από τι δυσκολίε που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα και γι' αυτό πρέπει να διασφαλίζεται ότι τους παρέχονται όλα εκείνα τα εχέγγυα για να μπορούν να αποδώσουν στους χώρους στους οποίους διαμένουν αλλά και παράλληλα να είναι ενημερωμένες πλήρως με απλή και κατανοητή γλώσσα για τα δικαιώματα, της υποχρέωσής τους από την αρμόδια αρχή του κράτους υποδοχής και να ξέρουν πως τυχόν παραβίαση είτε της σύμβασης είτε των δικαιωμάτων τους πρέπει να καταγγέλλονται. Η εργασία είναι καθαρά εποχικού χαρακτήρα στη βάση προκαθορισμένη συμφωνίας και όπω ζητείται από αυτές να εργαστούν είτε περισσότερες ώρες είτε με χαμηλές απολαβές είτε να κάνουν κάτι έξτρα από ό,τι προβλέπει η σύμβαση θα πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, να καταγγέλουν και το κράτος που τις φιλοξενεί θα πρέπει να έχει εκείνους τους μηχανισμούς και τους λειτουργούς που να γίνονται ακριβώς συστηματική έλεγχη συστάσεις στον εργοδότη, κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται. Θεωρούμε ότι ε, έχουν μπει οι βάσεις σε αυτή την οδηγία ε, για να προχωρήσουμε σε ένα διάλογο. Είναι σημαντικό κάποια θέματα που έχει θίξει και ο κύριος Κλωτ Μωράης στην εισαγωγική του ομιλία να συζητηθούν εκτενώς και με τα κράτη-μέλη αλλά και με τους εμπλεκόμενους όπως είναι το θέμα της επικουρικής η οι τομείς απασχόλησης. Εμείς ως Επιτροπή θεωρούμε ότι οι τομείς απασχόλησης είναι κυρίω η γεωργία και ο τουρισμό. Ε, δεν έχουμε βάλει τον κατασκευαστικό τομέα γιατί ποικίλει από χώρα σε χώρα. Οπωσδήποτε το θέμα στέγασης είναι καυτό γιατί πρέπει οι συνθήκε όπου διαμένουν οι εποχιακοί εργάτε και ειδικά οι γυναίκε να είναι τέτοιε που να είναι υγιεί οι συνθήκε. Και ε, όσον αφορά τους μηχανισμούς κυρώσεων, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί και με τα κράτη-μέλη. Ως Επιτροπή χαιρετίζουμε την πρόταση οδηγίας και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις ερωτήσεις, σα σας για να δώσουμε τις σχετικές απαντήσεις. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Παπαδοπούλου. Σημειώνουμε όσους θέλουν να λάβουν, λάβουν ε, μέρος στην ε, συζήτηση. Βλέπω ότι πολλοί από εσά θέλουν ήδη να κάνουν σχόλια ή ερωτήσεις. Δύο λεπτά ο καθένας για να απαντήσουν και τα μέλη του πάνελ. Η κυρία Ρομέρο Λόπεθ. Gracias, presidente. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να θέσω το εξή θέμα. Πώς μπορούμε να ευνοήσουμε την νόμιμη μετανάστευση αποφεύγοντας την αύξηση της παράνομης μετανάστευσης. Ακριβώς ε, για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο ε, λέει ο είναι αποτελεσματική δηλαδή όταν έχουμε τόσο μεγάλα ποσοστά παράνομης μετανάστευσης ο μόνος τρόπος νομίζω είναι να συνεργαστούμε με τις χώρες προέλευσης αν παραδείγματο χάρη μιλάμε για τις χώρες ε, από τον Νότο ή Λατινική Αμερική ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη, θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να οργανωθούμε όπως έγινε στις ευρωπαϊκές χώρες όταν εμείς ε, μεταναστεύουμε πολίτε των χωρών μα μεταναστεύουν προ άλλε χώρε. Θα πρέπει και εμεί τώρα από την πλευρά μα, που είμαστε χώρε υποδοχή, να δημιουργήσουμε του φορεί που θα διεκπεραιώνουν αυτέ τι ε, ε, ζήτηση, αν θέλετε, αυτέ τι αιτήσει και να ενημερώνουμε του μετανάστε και για τι υποχρεώσει και για τα δικαιώματά του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα ήταν καλό να ξέρουν οι εργαζόμενοι που έρχονται από τι χώρε καταγωγή, από τι χώρε προέλευση και ποια είναι τα δικαιώματά του και ποιε είναι οι υποχρεώσει εργασία του. Ιδίω σε χώρε που βρίσκονται τώρα σε δημοκρατική μετάβαση. Ε, Παραδείγματο χάρη, μια χώρα που έχει δικτατορικό καθεστώ θα είναι δύσκολο να μπορέσουμε να προωθήσουμε κάτι τέτοιο. Αλλά σε γειτονικέ μα χώρε που έχουμε και το μέσο γειτονία θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε για την μετανάστευση και για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων αυτών. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό πρώτο στοιχείο. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά την ευελιξία. Είναι γεγονό ότι θα πρέπει να καταλάβουμε τι εστί ευελιξία. Η ευελιξία δεν σημαίνει υποτίμηση δικαιωμάτων. Η ευελιξία δεν θα πρέπει να πλήξει την ισότιμη μεταχείριση, αλλά να αντιμετωπίζει κάποιες ιδιαιτερότητες ε, κρατών μελών. Τα είπε και ο κύριος ε, Κοφεράτη, ο στη Μάλτα και την Ανταλουσία τα πράγματα δεν μοιάζουν παραδείγματο χάρη με τη Φιλανδία. Η τουριστική περίοδο ε, ε, σε κάποιες χώρες είναι 9 μήνες. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα φορητότητας των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Γιατί κάποιες φορές ε, έχουμε εργαζόμενους που έρχονται κάθε χρόνο στην ίδια χώρα για να εργαστούν. Υπάρχει ένα σε επαναληπτικός χαρακτήρας και θα πρέπει ο εργαζόμενο αυτό, ο εργάτη αυτό να γνωρίζει, επαναλαμβάνω, τα δικαιώματά του αλλά και τι υποχρεώσει του. Τα συνδικάτα λοιπόν, είναι σημαντικό αυτό, όχι τα ευρωπαϊκά μόνο, αλλά και τα συνδικάτα των χωρών καταγωγή των χωρών προέλευση, να έχουν κάποιε επαφέ, κάποια σχέση με τα ευρωπαϊκά συνδικάτα. Να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν πληροφορίε ε, μεταξύ του. και νομίζω ότι και με τη Διεθνή Οργάνωση εργασία. Αυτό θα μπορούσε να καθοριστεί, να υπάρχει δηλαδή μια ανοιχτή γραμμή συνεργασία με τι χώρε καταγωγή αυτών των εργαζομένων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι κυρώσει, γιατί δεν μιλάμε για προστασία ε, των εργαζομένων, μιλάμε για προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, μιλάμε ε, για το ευάλωτο ε, αυτών των εργαζομένων, των εποχιακών. Και σε ό,τι αφορά και τα συνδικαλιστικά, δεν είναι η μόνη αυτή η ενδιαφέρουσα πτυχή, είναι και μια άλλη. Πώ οι επιθεωρήσεις εργασία των κρατών μελών, πώς μπορούν να έχουν ένα είδο συνεργασία. Γιατί φυσικά οι αγορέ εργασία αυτή τη στιγμή είναι κατά κάποιο τρόπο στεγανοποιημένε. Έχουν η κάθε χώρα τη δική τη αγορά εργασία. Ίσως έχουμε όμω το μέλλον μια συγχώνευση κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί να υπάρχει μεσογειακή αγορά εργασία, είπε παραδείγματι. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις ε, κυρώσεις. Πώς θα οργανωθούν, υπάρχουν κυρώσεις ενός ευρωπαϊκού οργανισμού. Όχι αυτή τη στιγμή, αλλά θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κάποια παρατηρητήρια, κάποιες υπηρεσίες, κάποιοι οργανισμοί οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιολογήσουν την κατάσταση. Τι γίνεται λοιπόν με τις επιθεωρήσεις εργασίας των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Και Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά υπάρχει πραγματικότητα αυτή των πολλών εποχιακών εργαζομένων στα, σε πολλά κράτη-μέλη. που δυστυχώς ε, δεν έχουν νόμιμο καθεστώς ε, στις περισσότερες χώρες και έχουν ε, το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης. Σε πολλές περιπτώσεις όμως είναι πάρα πολύ ευάλωτοι και συμφωνώ με τις απόψεις όλων των ε, ομιλητών ότι είναι διαφορετικές οι απόψεις ε, των κρατών μελών για το θέμα αυτό και βέβαια πρέπει να βρούμε έναν τρόπο διαχείρισης ε, της κυκλικής μετανάστευσης. Το ερώτημα όμως είναι το εξής και θα ήθελα μία απάντηση από τους ομιλητές για το ζήτημα αυτό. Προφανώς ε, η έγκριση της οδηγίας ε, για την εποχική εργασία φαίνεται να είναι ένα πολύ ε, σημαντικό εργαλείο. Δεν υπάρχει διαφωνία από αυτού. Ειδικότερα για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης που αυτή τη χρονική περίοδο επηρεάζονται περισσότερο από αυξανόμενο αριθμό μεταναστών λόγω της κρίσης στις αραβικές χώρες, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα παραμείνουν περισσότερο οι μεταχειακοί ή οι εποχικοί εργαζόμενοι και δεν θα γίνουν παράνομοι μετανάστες μετά ε, που θα εκπνεύσει η περίοδος διαμονής τους. Πώς θα αποφύγουμε την κατάχρηση μιας τέτοιας οδηγίας. Και το δεύτερο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω είναι το εξής. Εγώ με τον... είμαι, είμαι ισχυώδης συζητή στην έκθεση του Κλοντ και συμφωνούμε σε πολλά ε, από τα επιχειρήματά μας. Ε. Isn't it important to Στην έκθεση για τους εποχιακά εργαζομένους. Υπάρχουν όμως και διμερεί συμφωνίες, θα ληφθούν αυτές οι υπόψεις. Υπάρχουν και μερικές συμφωνίε μεταξύ των κρατών μελών για το θέμα αυτό. Για παράδειγμα, είδα το παράδειγμα της Ισπανίας που έχει διμερεί συμφωνίες με έξι τρίτες χώρες. Και για να ολοκληρώσω, είναι προφανές ότι υπάρχουν απαντήσεις στα ερωτήματά μας, αλλά πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές, τα μέλη του πάνελ που παρουσίασαν τη δουλειά τους, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική για τη διαχείριση του φαινομένου αυτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην νόμιμη μετανάστευση έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το πρόβλημα αυτό είναι το εξής. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της στρατηγικής ευρωπαϊκό επίπεδο και της στρατηγικής του κάθε κράτους μέλους. Η, η διαφορά αυτή της στρατηγικής δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ως προς την νόμιμη μετανάστευση, ειδικότερα στο τομέα της εποχική εργασίας. Έχουμε πολλά στοιχεία που μας δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι αυτοί που έρχονται από τρίτες χώρες ε, και εκείνοι που προέρχονται από τις ίδιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, την κάνουν εκμετάλλευση. Υπάρχουν δίκτυα εκμετάλλευση των εργαζομένων αυτών και πρέπει να πω ότι υπάρχουν για παράδειγμα τα γραφεία ευρέσεως εργασίας ε, που εξασφαλίζουν τη μεταφορά των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας τους. Και αναφέρομαι και στις δημόσιες αρχές. Υπάρχει ένα νομικό κενό στον τομέα της εργασία και συνεπώ χρειαζόμαστε ισχυρή νομοθεσία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα. Οι συνθήκες εργασίας των εποχιακών εργαζομένων πρέπει να βελτιωθούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε και ένα πρόβλημα μετανάστευσης των Ευρωπαίων εργαζομένων και μιλάω για παράδειγμα ε, πολίτες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ε, που ε, την χάνουν διακρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν εργαζόμενοι που έρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εργάζονται και διαβιούν σε καλύτερες συνθήκες από ότι οι πολίτες των, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί για τους Ευρωπαίους εργαζομένους ε, στις ευρωπαϊκές χώρες και πρέπει να ενισχυθεί η σχετική νομοθεσία. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πρέπει καταρχήν να έχουμε κατά νου τι ακριβώς επιθυμούμε και επιδιώκουμε με αυτή την πρωτοβουλία. Ε, πού στοχεύουμε. Δηλαδή, το θέμα είναι να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των εποχιακά εργαζομένων, να μην υπάρχουν διακρίσεις ή σε τελική ανάλυση αυτό που ενδιαφέρει είναι να προσελκύσουμε εργαζόμενους για δραστηριότητες που κανείς δεν θέλει ε, να τις ε, αναλάβει επειδή οι άλλοι είναι πιο φτηνοί. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα και επίσης να δούμε τι μας ενδιαφέρει εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως το πρώτο ερώτημα που σας ανέφερα γιατί πρέπει να δεχτούμε ότι έρχονται αυτή τη στιγμή εποχιακά εργαζόμενοι στην Ευρώπη και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Πρώτον λοιπόν εποχιακά εργαζόμενοι. Τι είναι ακριβώς αυτό. Μπορεί να είναι τα πάντα ε, ε λόγω κάποιου γεγονότος που μπορεί να είναι μια πλημμύρα, ένα σεισμός, οτιδήποτε άλλο. Ε, μπορεί να είναι η εποχή που παίζει ρόλο, είτε είναι άνοιξη, φθινόπωρο, οτιδήποτε άλλο. Είναι ανοιχτό το ότι είναι η εποχιακή εργασία. Πρέπει κανείς να το διευκρινίσει. Ή αλλιώς να πούμε εποχιακή εργασία είναι εκείνο που δεν θέλει να κάνει κανείς. Το άλλο που ενδιαφέρει είναι η κυκλική μετανάστευση. Ε, για μένα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στον κόσμο. Ε, όσοι επιθυμούν να εργαστούν στην Ευρώπη ε, θα συνεχίσουν να εργάζονται γιατί θέλουν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Εγώ το βρίσκω φυσιολογικό και δεν το εποκρίνω. Δεν το επικρίνω και ας μην προσποιούμε οτιδήποτε άλλο. Μετά μιλήσατε για έρευνα στην αγορά εργασίας. Εμείς αυτό το κάνουμε στην Γερμανία και έχουμε καταλήξει, όπως σας είπα, στο ότι υπάρχουν εργασίες που κανείς δεν θέλει να τις αναλάβει, τις αναλαμβάνουν ορισμένοι με πολλές γραφειοκρατικές δυσκολίες. Γι' αυτό λοιπόν, όταν γίνεται λόγος εδώ για μία ρύθμιση, εγώ θέλω να ληφθούν υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία. Και όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, θέλω να πω το εξή. Ε, αξιοπρεπής διαβίωση. Τι σημαίνει αξιοπρεπής ή ικανοποιητική. Το κριτήριο είναι για μένα η αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Οι άνθρωποι πρέπει να ζουν σωστά, καλά. Να μην συμβαίνει αυτό που συνέβη παραδείγματο χάρη στο Ροζάνο στην Ιταλία. Πρέπει λοιπόν και αυτό να, να διευκρινιστεί. Το αξιοπρεπή δεν είναι σαφέ. Μετά, ε, αποζημίωση. Εμεί θέλουμε ίση αμοιβή για ίση εργασία. Ε, να μην υπάρχει κοινωνικό ντάμπινγκ και να μην δεχτούμε εδώ νέου σκλάβου οι οποίοι αναλαμβάνουν τη βρώμικη δουλειά. Και κάτι τελευταίο. Συνδικαλιστικά δικαιώματα. Κοιτάξτε, στην Ευρώπη, εφόσον εργάζεται κανείς ε, πρέπει να έχει και δικαίωμα συνδικαλισμού. Δεν μπορεί κανεί να είναι λιγάκι έγκυος ή είτε είναι έγκυο ή όχι. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά που σας λέω τα βρίσκω σημαντικά. Η κυρία Μορβάη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω και εγώ τη γλώσσα μου, ουγγρικά. Στη συζήτηση αυτή για τη μετανάστευση, την εποχιακή εργασία, εργαζόμενους που έρχονται να εργαστούν στην Ευρώπη εκτός και προέρχονται από χώρες εκτός Ένωσης. Αυτό το οποίο με ενοχλεί σε όλη αυτή τη συζήτηση είναι ότι τελικά είναι κάτι το οποίο ε, λέμε ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και πρέπει έτσι να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί μιλάμε όμως ακριβώς. Μιλάμε για πολίτες, για πολίτες που ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης, οι οποίοι τελικά ε, πιέζονται και είναι υποχρεωμένοι λόγω της της αδικίας που υπάρχει στον κόσμο να ε, πάνε σε μια άλλη χώρα για να κάνουν δουλειές που οι πιο τυχεροί πολίτες άλλων χωρών δεν θέλουν να κάνουν ε, τη δουλειά, τις δουλειές αυτές ή δεν μπορούν γιατί μπορεί να μην υπάρχουν ε, αρκετοί εργαζόμενοι να κάνουν αυτές τις δουλειές κτλ. Επομένως πρέπει να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Δεν μιλάμε για υπηκόους ε, τρίτων χώρων. Πρέπει να λέμε τα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Εγώ προέρχομαι από την Ουγγαρία, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και κάποια χρόνια. Και αυτή τη στιγμή ασκεί η χώρα μου την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξακολουθούμε να είμαστε χώρα ε, που ε, στέλνει μετανάστες ε, προς ε, άλλες χώρες. Ε, πρέπει να δούμε τα πράγματα. Παραδείγματο χάρη, έχουμε ένα νοσοκομείο με νοσηλεύτερες πάρα πολύ μεγάλης ειδίκευσης. Όταν αυτές οι νοσηλεύτερες ή νοσηλευτές παίρνουν τις θερινές τους διακοπές και παίρνουν 250-300 ευρώ. Τι κάνουν το καλοκαίρι, πηγαίνουν σε μια άλλη χώρα, την Αυστρία και εκεί εργάζονται. Εργάζονται εποχιακά, κάνουν κάποια γεωργική εργασία οι καθηγήτριες ε, που έχουν δίπλωμα, έχουν ένα πτυχίο και πόσα παίρνουν 250-300 ε, ευρώ στη χώρα τους, ε, στη χώρα μας. Πηγαίνουν και καθαρίζουν, καθαρίζουν σπίτια στην Αυστρία, στη Γερμανία. Μιλάμε για ισότητα λοιπόν. Μα λέτε ότι αυτό το έγγραφο μεταξύ άλλων απαραίτητο για να έχουμε ισότητα, ισότητα μεταχείριση. Εγώ θα σας πω το εξή. ισότητα θα έχουμε όταν μόνο το, οι, ίδιες, ο ίδιος αριθμός καθηγητών και καθηγητριών από την Αυστρία και την Γερμανία έρχονται στην ε, Ουγγαρία ή όταν έρθουν να κάνουν γεωργική εργασία Γερμανοί και Αυστριακοί εργάτες. Ζητώ συγγνώμη ε, αλλά δώσατε το λόγο για τέσσερα ή πέντε λεπτά ε, σε άλλους συναδέλφους και εδώ τώρα μου λέτε να προσέχω το ρολόι. Λοιπόν, υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, έχουμε το φαινόμενο της μετανάστευσης και ίσως θα πρέπει στις χώρες ε, που υποδέχονται μετανάστες να προσκληθούν κάποιοι από τις χώρες που στέλνουν μετανάστες για να δουν τις συνθήκες εργασίας να δουν επίσης οι εποχικοί εργαζόμενοι τι ε, μπορούν να κάνουν και τι μπορούν να προσφέρουν. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για κάτι φυσιολογικό, είναι, α, πρόκειται για αδικία όλα αυτά που γίνονται. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο πράγματα. Πρώτον, Για ποιο λόγο θέλουμε ρύθμιση για τους εποχιακά εργαζομένους. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν ε, παράτυπα, είτε σε μόνιμη εργασία είτε σε εποχιακή εργασία και που έρχονται από τρίτες χώρες. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρειαζόμαστε μια ρύθμιση αυτών των εργασιών ε, που δεν απαιτούν πολλά επαγγελματικά προσόντα, που δεν πληρώνονται πολύ καλά, γιατί διαφορετικά οι άνθρωποι αυτοί κάνουν τις δουλειές αυτές παράνομα. Χρειάζεται λοιπόν μια ρύθμιση, η οποία θα ήταν μια πρώτη λύση για την καταπολέμηση της παράνομης εργασίας ε, ή για την ε, νομιμοποίηση των ανθρώπων αυτών που τους χρειαζόμαστε τόσο πολύ για την οικονομία μας. Δεύτερο σημείο. Είναι προφανές ότι όσοι έρχονται να εργαστούν εποχιακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πληρώνονται με τους ίδιους μισθούς. Όμως το πρόβλημα είναι τα άλλα τους δικαιώματα και στις παρατηρήσεις του Συμβουλίου διαπίστωσα ότι αυτό που προτείνει το Συμβούλιο είναι τελείως διαφορετικό όταν μιλάμε για παράδειγμα για συμβάσεις 12 εβδομάδων. Η εποχή δεν έχει τελειώσει σε 12 εβδομάδες και είναι δύσκολο συνεπώ να εργαστούμε για ένα τέτοιο χρονικό διάστημα και να διατηρούμε και μία αλφα οικονομική κατάσταση στη χώρα προέλευσης. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι εμεί καλύπτουμε μια ανάγκη ε, εργασίας που υπάρχει στη δική μας τη χώρα. Αυτό δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Thank you. Um, <clears throat> to allow immigration, even to για να επιτρέψουμε και να ενθαρρύνουμε τη μετανάστευση, μερικές ε, φορές έχουμε μια πολύ φιλελεύθερη και γενναιόδορη πολιτική. Όμω αυτό προποθέτει ότι υπάρχει και κάποια ε, ανάγκη και επιθυμία των ανθρώπων να φύγουν από την, ε, τα οικεία του μέρη και να πάνε σε μέρη που τους είναι εντελώ ανίκια. Υπάρχουν βέβαια και συνέπειες ε, από τον πόλεμο, από ε, διάφορα προβλήματα που προκαλούν συχνά οι δυτικέ χώρες ε, και πολλές φορές λόγω της, της βιομηχανίας ψυχαγωγίας Συνεπώ, ε, τα αποτελέσματα και όλα αυτά που δίνουμε στους ανθρώπους αυτούς δεν είναι καθόλου γενναιόδωρα. Ε, θέλουμε να τους πετάξουμε του ανθρώπους αυτούς όταν πια δεν τους χρειαζόμαστε γιατί του θεωρούμε αναλώσιμα. Η εποχιακή και η τα μετατιθέμενοι ε, έχουν τα ίδια κίνητρα και πολλές φορές οι πολιτικοί τους χρησιμοποιούν. Δεν τους βλέπουν ως ανθρώπους ε, που έχουν επιθυμίες, αλλά ως μηχανές παραγωγής που απλώς τους πηγαίνουν από εδώ και από εκεί για να κάνουν τη δουλειά τους και μάλιστα μερικές φορές χωρίς συγκεκριμένο κόστος. Είδαμε τις καταστάσεις στο Ροζάρνο, ήταν τραγικές η τραγική κατάσταση. Άνθρωποι που δούλευαν ε, για 3 ευρώ την ημέρα, 12 μέρες. Ε, μιλάμε για φοβερές καταστάσεις. Κάτι άλλο που μάθαμε εκεί είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι ε, που πληρώνονται κάτω από το βασικό μισθό και δεν έχουν καν συμβάσεις εργασίας. Ε, τουλάχιστον θα μπορούσαν ε, να τη θέση σε αυτές εργασίες με σωστό μισθό εργασίας από ντόπιου εργαζομένους. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν θεωρούνται μερικές φορές, θεωρούνται προνομιούχοι, όμως είναι παράλληλα και πολύ πιο ακριβή για την παραγωγή αν χρειαζόμαστε λοιπόν ανθρώπους χαμηλότερης εξειδίκευσης από τις τρίτες χώρες, ε, ε, τους συμπεριφερόμαστε έτσι γιατί χρειαζόμαστε, ε, τον, ε, χρειαζόμαστε τους ανθρώπους αυτούς, ε, νομίζουμε ότι μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε. Όμως ε, υπάρχουν και άλλες χώρες που μπορούν να τους προσφέρουν εργασία. Επίσης, μερικές φορές Υπάρχει και το θέμα των εργοδοτών, γιατί χρησιμοποιούν ε, τους εποχιακά εργαζομένους ε, για να αυξήσουν τα κέρδη τους και δεν πρέπει να επιτρέψουμε στους ανθρώπους αυτούς να εκμεταλλεύονται τους εποχιακά εργαζομένους. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπλινκεβιτσιούτε και μετά θα απαντήσουν οι προσκεκλημένοι μας. Παρακαλώ, είστε σύντομοι. Ε, Πρόεδρε, Είμαι απόλυτα σίγουρη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται και τα δύο. Και τους ε, εξειδικευμένου και του ανειδίκευτου ε, που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να τη δούμε κατάματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενεθάρρυνε για μεγάλο χρονικό διάστημα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταθέσει ε, μια οδηγία που θα ρυθμίζει την εποχιακή εργασία. Σήμερα λοιπόν έχουμε την πρόταση αυτή και νομίζω πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε η οδηγία αυτή να ωφελήσει τόσο τους πολίτες της Ένωσης όσο και εκείνους που έρχονται εδώ για να εργαστούν. Επιθυμώ να εστιάσω την προσοχή μου σε ένα στοιχείο της πρότασης. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που ισχυρίστηκαν ότι οι εποχιακά εργαζόμενοι πολύ συχνά εργάζονται ως σκλάβοι και οι συνθήκες διαβίωσης τους ε, είναι τρομακτικές. Κατόπιν τούτου η οδηγία οφείλει να προβλέψει τη δημιουργία εκείνων των συνθήκων που θα καθιστά αδύνατο αυτό που συμβαίνει σήμερα. Οι εποχιακά εργαζόμενοι να μην είναι σκλάβοι. Άρα δηλαδή χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό ελέγχου, χρειαζόμαστε επίσης ένα μηχανισμό καταγγελιών, ε, οι επιθορήσεις ε, εργασίας ε, που ελέγχουν την εφαρμογή των οδηγιών πρέπει να εργαστούν σκληρότερα. Υπάρχει κάτι που κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όπως και τα συνδικάτα. Πιστεύω επίσης ότι οι κοινωνικοί εταίροι νομίζω ότι εκλήθησαν να συμμετάσχουν σε αυτή την ακρόαση. Ένας εργαζόμενος που έρχεται από μία ε, τρίτη χώρα ενδέχεται να δεχτεί να δουλέψει ως σκλάβος γιατί δεν μπορεί να φανταστεί κάτι καλύτερο. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός να ενημερωθεί για τα δικαιώματά του ε, να γνωρίζει ότι μπορεί, μπορεί, μπορεί να πει όχι δεν θέλω να εργαστώ ως σκλάβος. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ε, έγιναν πολλά σχόλια, λίγες βέβαια ερωτήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, προτείνω ε, κάθε ένας από τους ομιλητές στο πάνελ να προσπαθήσει να εστιάσει την προσοχή του σε αυτά που τον αφορούν σε αυτά που ελέγχθησαν είτε με τη μορφή σχολείου είτε με τη μορφή ερώτησης. Η Επιτροπή πολιτικών ελευθεριών, ο κύριος Μωράη καταρχήν. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ε, καταρχήν είμαι ευγνώμων ε, στους ευρωβουλευτές ε, που ήρθαν εδώ ίσως την τελευταία μέρα πριν από τις διακοπές. Εκείνο το οποίο ακούστηκε στις ερωτήσεις είναι ότι για πρώτη φορά ένας μια οδηγία που ασχολείται με αγορά εργασία, ασχολείται με ανειδίκευτους. Μέχρι τώρα ασχοληθήκαμε με όλους τους άλλους. Ε, τώρα λοιπόν μιλάμε για αυτά τα οποία μίλησε η κυρία Μπλανκεβίτς, ε, κοιτάμε την αλήθεια κατάμετα Και όποια και είναι η φιλοσοφική συζήτηση για την ε, μετανάστευση, σε τελική ανάλυση υπάρχει μία πραγματικότητα. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένων εποχιακών που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλοι νόμιμα, άλλοι παράνομα. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα. Αν θέλετε μπορούμε να έχουμε μία φιλοσοφική συζήτηση για τη μετανάστευση ε, αλλά πάση εγώ είμαι ευγνώμων για την πρώτη γενιά των μεταναστών οι γονεί μου ε, ήρθαν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήρθα και εγώ εμείς είχαμε βέβαια τη γλώσσα που μας συνέδεε δεν ήρθαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον καλό του καιρό για να δουλέψουμε ήρθαμε αυτή λοιπόν είναι μια πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι είτε εξετάζει κανείς την κατάσταση τώρα ως έχει με όλα τα περίπλοκα παρακλάδια της είτε την αγνοεί. Πρόκειται για επιλογή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει και μια φιλοσοφική συζήτηση για τη χρήση της εργασίας, για την εκμετάλλευση, ε, για ε, τα κίνητρα που προκύπτουν από τη φτώχεια. Πολλά ελέγξαν από τους συναντέλφου. Η κυρία Ρομέρα Λόπες έφυξε αυτά τα θέματα όμως ε, Νομίζω ότι μαζί με την κυρία Αργεντίνη και με τον κύριο Κοφεράτη κυρίως ε, έθιξαν το θέμα της ε, πολυπλοκότητας στην πρακτική. Τι συνέπειες θα υπάρχουν ε, για τους εποχιακούς εργαζόμενους. Η διάρκεια παραμονής είναι ένα κρίσιμο θέμα. Αυτή τη στιγμή ορισμένες χώρες έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες, κάτι που ανέφερε και ο κύριος αλλά πρέπει να έχουμε μια πιο προχωρημένη προσέγγιση η κυρία Ρομέρο Λόπες μίλησε για την ενημέρωση των εργαζομένων, για την ευελιξία, για την συμμεταχείριση, τη φορητότητα. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν αποδεικνύουν πώς μπορεί να βελτιωθεί η έκθεση. Γιατί ε, δεν πρόκειται για ε, μία μαγική συνταγή. ή συλλογικέ συμβάσει είναι ένα σημαντικό θέμα που το έθιξε ο κ. Κοφεράτη και θα εξαστεί κυρίω στην Επιστροπή Απασχόληση. Είναι όμω καθοριστική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωρίζω ότι θα το εξετάσουν τα συνδικάτα και η Ένωση. Ο κ. Παπα-Νικολάου έθιξε το θέμα των παράνομων μεταναστών ε, και πώς μπορούν αυτοί να παραμείνουν σε μια χώρα και να μην επιστρέψουν. Πρώτα απ' όλα, όπως είπε και η κυρία Ρομέρο Λόπες, ε, στην πρόταση υπάρχει ένα κίνητρο. Καταρχήν, να μην είναι πλέον ελκυστική η εποχιακή εργασία. Αυτό είναι εγγενές στην πρόταση, ε, δημιουργώντας ε, τις νόμιμες οδούς προς τη μετανάστευση που είναι κομμένες και ραμμένοι ε, ραμμένες ε, στον τομέα όπου υπάρχει ζήτηση, με τον τρόπο αυτό παρεμποδίζει κανείς την παράνομη μετανάστευση. Βασική αρχή αυτή που διέπει την πρόταση. Υπάρχουν όμως και άλλα κίνητρα ε, για να παρεμποδιστούν οι άνθρωποι να παραμείνουν. Υπάρχουν ταχύρυθμες διαδικασίες που μπορούν να τις εκμεταλλευτούν οι εποχιακοί εργαζόμενοι, όμως δεν θα ισχύουν αυτές εφόσον ε, παραμένουν και μετά το χρονικό διάστημα που προβλέπεται για αυτούς. Ε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν αντικίνητρα για κάποιον ας πούμε, που θέλει να έρχεται κάθε χρόνο για εποχιακή εργασία. Αυτά όλα υπάρχουν στην έκθεση. Βεβαίως το θέμα του ελέγχου ε, και εφαρμογής του νόμου, αυτό είναι θέμα κρατών μελών. Πάντως ε, η ε, πρόταση περιλαμβάνει κίνητρα. Κατά τα άλλα, βεβαίως υπάρχει και το θέμα των οικονομικών εμβασμάτων. Για όσους πιστεύουν αντιμετωπίζουν την απασχόληση πάλι κάτω από φιλοσοφικό επίπεδο πρέπει να δούμε ότι ε, τα εμβάσματα ε, προέρχονται και από εποχιακά εργαζόμενους ε, και από νόμους μετανάστες. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν δουλειά που κανείς δεν θέλει να κάνει και αυτό είναι αλήθεια, όμως η ισορροπία ανάμεσα σε πολλές από τις χώρες που προσφέρουν τέτοιου είδου μετανάστες και η οικονομική του ανάπτυξη, αυτά τα δύο στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Σε κάθε πρόταση μετανάστευσης που κατατίθεται υπάρχουν δύο πολιτικές κατευθύνσεις. Είτε μπορεί κανείς να ζητήσει περισσότερο έλεγχο ή ε, περισσότερη φιλελεύθερη προσέγγιση. Αυτή η περισσοτερη φιλελευθερη προσεγγιση αυτη η δικη μας η πρόταση έχει ως στόχο να περιορίσει την εκμετάλλευση και να συστήσει έναν οικονομικά λογικό μηχανισμό εφόσον επιθυμούμε να λύσουμε το θέμα της Ετέθηκε το θέμα των ε, γραφείων διαμεσολάβησης. Ε, ε, αυτό δεν το αντιμετωπίζει η έκθεση και είναι ένα θέμα που ίσως θα έπρεπε να εξεταστεί. Ε, έγιναν πολλές συζητήσεις στην οδηγία τη σχετική που προβλέπει το θέμα των γραφείων προσφοράς εργασίας. Η κυρία Μπλίνκεβιτσιούτα και ο κύριος Κοφεράτη μίλησαν για το θέμα των κοινωνικών εταίρων. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό οι κοινωνικοί εταίροι να συμμετέχουν, αλλά και οι ΜΚΟ, οι, οποίοι, οποίες ε, έχουν να κάνουν με εκατομμύρια εργαζομένων. Ε, δεν μιλάμε για αυτούς ε, γιατί ζουν κάπου σε μία γκρίζα ζώνη. Πάντως γίνεται λόγος ε, για τον τρόπο που ζουν και για τον τρόπο ε, που γίνονται θύμα εκμετάλλευση. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουν και άλλοι και ζητώ συγγνώμη από τους αντέλφους εκείνους ε, των οποίων δεν απάντησα στις ερωτήσεις τους. Η κυρία Σίγκαν, παρακαλώ θέλετε να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Πολλά επιχειρήματα, πολλά σχόλια είναι ήδη γνωστά αλλά από τη στιγμή που επαναλαμβάνονται σημαίνει ότι έχουν μεγάλη σημασία για αυτή τη συζήτηση. Δεν θέλω να κάνω φιλοσοφική συζήτηση, αλλά όταν άκουσα τα σχόλια περί στρατηγικής ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο κρατών μελών, το ζήτημα της αντιμετώπισης αυτής της οδηγίας ως ενός εργαλείου για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης. Θα ήθελα να επαναλάβω κάτι που προσπάθησα να το πω και ευθύ εξ αρχής. Αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη είναι μια συνεκτική διαχείριση ε, της μετανάστευσης, μια καλή διαχείριση που όχι να μην είναι μόνο φιλοσοφική και ιδεολογική, αλλά πρώτα απ' όλα ρεαλιστική, πραγματιστική. Και σχεδιάζουμε ακριβώς ε, το ίδιο που είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε και στο παρελθόν όπως ε, και η Κομισιόν έτσι και εμείς έχουμε εντολή να προχωρήσουμε τομεακά με αυτό το πρόγραμμα. Ναι, θα το κάνουμε αυτό, αλλά αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα περιέχει σαφείς κανόνες που θα ρυθμίζουν ε, την ομετανάστευση είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να συνεχίσουμε να συγκροτούμε την όλη αυτή πρόταση με διάφορα στοιχεία και να έχουμε υπόψη μας και το απότερο μέλλον. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο τώρα τομέα εργαζομένου. Θα εργαστούμε βάσει διαβουλεύσεων και βάσει των πρακτικών που παρατηρούμε στα κράτη-μέλη. Και θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε μια οδηγία η οποία θα ρυθμίζει την κατάσταση για το συγκεκριμένο αυτό τομέα που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μιλάμε για άτομα ευάλωτα, όλοι αναφερθήκατε στην ε, πιθανή εκμετάλλευση και κατάχρηση που υφίστανται. Και αυτό το οποίο προσπαθούμε να προτείνουμε είναι ομοιόμορφη, καλά καθορισμένη, ταχεία διαδικασία που θα μπορεί να ελέγχεται, να παρακολουθείτε και θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα άτομα αυτά πράγματι ε, την χάνουν μιας αξιοπρεπούς μεταχείρισης. Ε, φυσικά και δεν είναι σκλάβοι που έρχονται να κάνουν δουλειές που κανείς άλλος δεν θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσει κάποιες και να καλύψει κάποια κενά που έχει ε, ε, σε διάφορους τομείς, σε ό,τι αφορά δηλαδή το εργατικό δυναμικό. Αλλά πρέπει να αυτό να γίνει με αξιοπρεπή τρόπο. Τώρα σε ό,τι αφορά κυρώσει σε περίπτωση που υπερβαίνουν το διάστημα νόμιμης διαμονής τα άτομα αυτά. Θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα των ε, εποχιακών εργαζομένων. Εν μέρη βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί από τα κράτη-μέλη, αλλά η Κομισιόν που είναι θεματοφύλακα των συνθήκων θα παρακολουθεί την υλοποίηση της οδηγίας. Πιέζει ο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Τέλο πάντων, θέλω να επαναλάβω ότι παραμένουμε στη διάθεσή σα και αν θέλετε να έχουμε διάλογο ή να απαντήσουμε οποιοδήποτε συγκεκριμένο ερώτημα για να εξηγήσουμε ε, τι σημαίνουν κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο του μηχανισμού ή τη πρόταση, μπορείτε να έλθετε άμεσα σε επαφή μαζί. Κυρία Βαντάση, σύντομα σα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για όλη αυτή τη συζήτηση και βλέπω και εγώ ότι υπήρξαν κάποια συγκεκριμένα επιχειρήματα, κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα πολύ παρόμοια με τη συζήτηση που έχουμε και εμείς στην ομάδα εργασίας για τους ορισμούς, για τους τομείς, για την διάρκεια της παραμονής και επίσης τα πολύπλοκα ζητήματα του των δικαιωμάτων που έχουν ή πρέπει να έχουν οι εποχιακοί εργαζόμενοι. Είναι όπω σα είπα, έντονε και εντατικέ συζητήσει και στην ομάδα εργασία, αλλά και η σημερινή συζήτηση ήταν πάρα πολύ χρήσιμη, αλλά θα επακολουθήσουν επίση ε, επικοδομητικέ, ελπίζω, συζητήσει. Θα ήθελα να τονίσω το εξή. Όταν εγώ έκανα λόγο για ευελιξία Αυτό το εννοούσα ως ανάγκη τα κράτη-μέλη τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα να έχουν αυτή τη δυνατότητα της ευελιξίας. Δηλαδή ήδη υπάρχουν εμπειρίες και μάλιστα καλές εμπειρίες αν λοιπόν τα κράτη-μέλη θέλουν να χρησιμοποιήσουν κάποια θετικά στοιχεία, να μπορούν να το πράξουν, να, υπάρχει δηλαδή αυτή η ευελιξία. Αυτό εννοούσα. Οι συζητήσει στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου θα συνεχιστούν με πολύ εντατικού ρυθμού και φυσικά βασιζόμαστε και προσβλέπουμε στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριο Σκοφεράτη, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επειδή συμφωνούμε όλοι ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, νομίζω ότι είναι σκόπιμο να μην το υπεραπλουστεύσουμε ε, και να μην καταλήξουμε σε καταπροσέγγιση ορισμούς. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα το οποίο θα ήθελα ταχύτατα να αναφέρω. Η εποχιακή εργασία δεν αφορά μόνο τους μετανάστες. Η εποχιακή εργασία αφορά μετανάστες και εργαζόμενους ντόπιου της χώρας εδώ λοιπόν τίθεται το πρώτο πρόβλημα. Είναι ε, το θέμα της ε, ίσης μεταχείρισης. Ε, για να μην έχουμε για την ίδια δραστηριότητα ένα ντάμπινγκ το οποίο τελικά θα τιμωρήσει όλους. Όταν λοιπόν εγώ μίλησα για ευελιξία, το έπραξα αυτό διότι υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία θέλω τώρα πολύ γρήγορα να εξηγήσω. Ποια είναι η ευελιξία που έχω εγώ κατά νου. Ε, ευελιξία αφορά καταρχήν ε, τους κλάδους και η ευελιξία αφορά κατά δεύτερον τους χρόνους. Όσον αφορά τους ε, κλάδους, κλάδοι καθαρά εποχιακοί υπάρχουν μόνο δύο. Δηλαδή ο τουρισμός και η γεωργία. Εγώ δεν νομίζω ότι ο κατασκευαστικός τομέας είναι εποχιακής εργασίας ε, γιατί ίσως ε, μπορεί ε, να είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον εποχιακά εργαζόμενο να κατασκευάσει μόνο τη σκεπή ενός σπιτιού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εποχιακή εργασία. Κατόπιν υπάρχουν κάποιες άλλες μικρές δραστηριότητε μεταποίησης που όμως ποικίλουν από κράτος σε κράτος. Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα του τι συμβαίνει στην Ιταλία και έτσι να μην προσβάλλω κανένα, να μην προσβάλλω την ευαισθησία του. Στην Ιταλία υπάρχουν πολλές αγελάδε που το πρωί αρμέγονται για το γάλα. Και αυτό είναι μια δουλειά που εδώ και δεκαετίες δεν την κάνουν οι Ιταλοί. Δεν υπάρχει ούτε ένας ε, Ιταλός κτηνοτρόφος που να αρμέγει τους, ε, τις αγελάδες. Τώρα η ΣΥΧ είναι εκείνη που στην ε, ε κοιλάδα του Πάντου αρμέγουν τις ε, αγελάδες ή το κρασί που πίνετε και σας αρέσει παραδείγματο χάρη το βίνο από το πιεμόντε ε, το κρασί με το κρασί αυτό δεν κατασκευάζεται από Ιταλούς αλλά από Μακεδόνες οι οποίοι ε, τα κάνουν πάρα πολύ καλά, τα καταφέρνουν πολύ καλά στα, στα Τα σταφύλια τα μαζεύουν οι Ιταλοί, μετά όμως ε, μπαίνουν οι Μακεδόνες που τώρα πια είναι βιομηχανικοί εργάτες. Δηλαδή βλέπετε σε μία χώρα μιλάμε για μία μεταποιητική εργασία η οποία είναι εποχιακής μορφής. Ε, ε, γιατί βεβαίως αν έχετε ένα κρασί το οποίο το βάλ μίξ δικαιωμένοι εργαζόμενοι σε, μία, σε ένα μπουκάλι αυτό δεν θα αρέσει κανέναν, θα το πετάξουν. Ως εκ τούτου που θέλω να καταλήξω, η οδηγία κατά τη δική δική μου άποψη οφείλει να αναφέρεται σε αυτό που είναι διαρθρωτικό. Σε δύο τομεί, όπως σα είπα. Και μετά βέβαια τα κράτη-μέλη έχουν δυνατότητα να προσθέσουν άλλες μικρές δραστηριότητε. Το ίδιο ισχύει και για τη διάρκεια. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι τα, οι τρει μήνες είναι λάθος. Είναι λάθος καταρχήν ως παραδοχή το όριο πρέπει να είναι πολύ πιο ψηλά και πρέπει να καθορίσουμε ένα κατώτατο όριο διάρκειας και μετά να μπορούμε να επιτρέψουμε λύσεις ε, που να είναι πιο προχωρημένες γιατί όσο πιο πολύ προς τα κάτω κατεβαίνει το όριο τόσο πιο πολύ δίνουμε κίνητρα για την παρανομία γιατί πιστεύετε ότι θα έρθει κάποιος από το άλλο μέρος του κόσμου στην Ευρώπη για τρεις μήνες μα είναι δυνατόν ε, για δέστε αυτά τα οποία ε, συζητάμε και μόνο ο χρόνος που χρειάζεται για την εφαρμογή του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι έξι μήνε είναι το κατώτατο όριο. Όμω για πάρα πολλέ χώρε τη Μεσογείου οι εννέα μήνε τώρα πλέον είναι μία πραγματικότητα, είναι μία κατοχυρωμένη εποχιακή εργασία. Και αν μιλάμε για σωστή διάρκεια, αυτό διευκολύνει και την ομοποίηση. Μπορούν να μεταφερθούν κάποια δικαιώματα, κυρίως όσον αφορά την κοινωνική περίθαλψη. Εγώ δεν, ε, ε, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ευελιξία στα δικαιώματα. Δικαιώματα είναι άκαμπτα. Όμως εκείνο που με εκπλήσει είναι η ε, η εχθρική διάθεση ορισμένων απέναντι στη φορητότητα, αν θέλετε, των συντάξεων ή των καταβληθέντων εισφορών. Κάποιος που έχει γεννηθεί σε άλλο μέρος του κόσμου τον εμποδίζεται να έρθει στην πατρίδα του και τον εμποδίζεται να πάρει τη σύνταξή του στην πατρίδα του όταν κάποιος βγαίνει στη σύνταξη δεν έχει υψηλότερο εισόδημα. Έχει απλά το εισόδημα το οποίο προέκυψε μέσα από την καταβολή των εισφορών του. Ως εκ τούτου η φορητότητα ε, των ασφαλιστικών εισφορών είναι καθοριστική σημασίας για να υπάρχει διαφάνεια και κυρίως για να κινητροδοτηθεί η επιστροφή. Υπάρχει ένα φαινόμενο που είναι πιο περίπλοκο από τη μετανάστευση. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στην Ευρώπη και εδώ παραμένουν ε, για όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι που θέλουν να επιστρέψουν. Κατόπιν τούτου υπάρχει ε, διαφοροποιημένη προσέγγιση. Βλέπουμε ότι δεν τους θέλουμε, μετά έρχονται εδώ, ε, τους χρειαζόμαστε όμως και αφού έρχονται εδώ θέλουμε κάπως να τους φυλακίσουμε προσφέροντας τους πολύ εχθρικές συνθήκες εργασίας. Αυτές λοιπόν λοιπόν είναι αντιφάσεις οι οποίες πρέπει κατά κάποιον τρόπο να αντιμετωπιστούν. τις ερωτήσεις ε, και τις επισημάσεις. Έχω ομαδοποιήσει τρεις κατηγορίες στις οποίες θα κάνω παρέμβαση. Η πρώτη είναι ότι οι εποχικοί εργάτες ε, συνήθως είναι άτομα με χαμηλή ειδίκευση που κάνουν εργασίες που δεν κάνουν οι ντόπιοι. Μπορεί να είναι άτομα που προέρχονται από τρίτε χώρε, μπορεί όμω να είναι και Ευρωπαίοι που διακινούνται από χώρε φτωχότερε σε άλλε όπου υπάρχουν θέσει εργασία. Επομένω, οι κοινή συνισταμένοι που εμεί επιδιώκουμε και με την οδηγία, και εκεί είναι που πρέπει να προσπαθήσουμε, είναι να μην υπάρχει εκμετάλλευση των ανθρώπων αυτών που αναγκάζονται να κάνουν εργασίε συγκεκριμένε, ε, να μην αποτελούν φτηνά εργατικά χέρια και πρωτίστω ε, να υπάρχουν μηχανισμοί μηχανισμοί στις χώρες υποδοχής που να διασφαλίζουν ότι οι νέοι συνθήκε διαβίωση του είναι σωστέ, είναι αξιοπρεπεί, γίνονται συστηματικοί έλεγχοι από αρμοδίου του κράτου για να μην υπάρχει ακριβώ αυτή η εκμετάλλευση που συνήθω ε, είναι σε βάρο ευάλωτων ομάδων, όπω έχω πει, των γυναικών. Ε, το δεύτερο, η δεύτερη επισήμαση είναι ότι αυτό που έχει πει ο κ. Παπα-Νικολάου, ότι οι νότιε χώρε τη Ευρώπη χρήζουν κοινοτική αλληλεγγύη, γιατί δέχονται μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα ιδιαίτερα σήμερα που γίνονται τόσε πολλέ ανακατατάξει στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή. Και εδώ θα πρέπει να το προσέξουμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι τελείω διαφορετικέ οι συνθήκε που αντιμετωπίζει η Νότια Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Κύπρο, η Μάλτα, αυτέ οι χώρε που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, παρά οι υπόλοιπε χώρε τη Κεντρική ή τη Βόρεια Ευρώπη. Εδώ ακριβώ θα πρέπει να υπάρξει σωστή μεθόδευση ε, της οδηγίας ώστε αυτές οι χώρες να βοηθηθούν στην καταπολέμηση της παράνομης εισρωής εποχικών εργατών και άλλων παρανόμων και ε, να υπάρχει ε, μια εκτενής, ένας εκτενής διάλογος για να μπορεί να ακούσουμε και τις φωνές των κρατών μελών τέτοιων χωρών που βρίσκονται στην νότια ευρώπη που αντιμετωπίζουν άμεσα πρόβλημα. και το τελευταίο είναι ότι χρειάζονται στατιστικά στοιχεία για την εποχική απασχόληση στα διάφορα κράτη μέλη και οπωσδήποτε δεν υπάρχει μακικό ραβδί που να διασφαλίσει όλους αυτούς τους εποχικούς εργάτες. χρειάζεται πολιτική βούληση διάλογος και είναι τελείως ξεχωριστό θέμα πώς αντιμετωπίζονται οι νόμιμοι εργαζόμενοι και πώ αντιμετωπίζονται οι εποχικοί εργάτε αλλά και οι παράνομοι, εργαζόμενοι. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις, πάταξη της παραοικονομίας, της αδούλωτης εργασίας και να υπάρχουν συμβάσεις όσον αφορά τους εποχικούς εργάτες οι οποίες να διασφαλίζονται ότι τηρούνται και δεν υπάρχει εκμετάλλευση σε βάρος των ευάλωτων ομάδων των εποχικών εργατών. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοδομητική συζήτηση του πρώτου τμήματο της ε, ε, πρωινή μα συνεδρία και επειδή έχουμε αργήσει να πάμε αμέσω. Υποδεχόμαστε λοιπόν τα, δεύτερα, τα μέλη του δεύτερου πάνελ, τους καλωσορίζουμε και τους ζητούμε να έρθουν εδώ, να πάρουν τη θέση τους και ευχαριστώ τους προσκεκλημένους του πρώτου πάνελ για την συμβολή τους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 Now, if you please, be kind enough to help us out. Παρακαλώ βοηθήστε με να προχωρήσουμε στο δεύτερο τμήμα της συνεδρίασης.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 Έχουμε τρία διαφορετικά πάνελ και αυτό το δεύτερο. Αυτό που θα αρχίσουμε τώρα. Με τους κοινωνικούς εταίρους. Για τους εποχιακά εργαζομένους. Θα ακούσουμε τώρα από τους κοινωνικούς εταίρους. Αρχίζουμε λοιπόν. Επαναλαμβάνω κοινωνικοί εταίροι να μας πούν τις απόψεις τους για την πρόταση της Επιτροπής και για το έγγραφο εργασίας του εισηγητή. Έχουμε προσκαλέσει την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων, την ΕΤΟΥΚ, τον κύριο Ντεκαγιό, ο οποίος δεν μπορεί να έρθει και τον αντικαθιστά ο κύριος Σοριάνο. Καλώς ορίσατε. Μετά, θα ακούσουμε τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων. Εκπροσωπείται από τον κύριο Ρούντεμπεργκ. Καλώς ήρθατε. Επίσης έχουμε καλέσει εκπρόσωπο της Ιταλικής Ομοσπονδίας Εργαζομένων ε, που εργάζεται με εποχιακούς εργαζομένους επιτόπου από την CG. ο κύριος Μεσίνα. Κυρία, κυρία Μεσίνα, συγγνώμη. Καλώς ήρθατε. Και επίσης έχουμε και την άποψη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που εκπροσωπείται από την κυρία Χόφμαν. Αρχίζουμε λοιπόν και ελπίζουμε να έχουμε χρόνο μετά για τη συζήτηση. Πρώτο, ο κύριος Σουριάνο. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντικαθιστώ τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικάτων που λόγω ασθενείας ε, δεν μπόρεσε να παραστεί εγώ προσωπικά είμαι αρμόδιος για τον τομέα της μετανάστευσης της ΕΤΟΚ. Έχω ένα περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μου. Δεν θέλω πρώτα απ' όλα να εκφράσω κάποια ε, μικρή ανησυχία που έχω. Αυτό το οποίο με ανησύχησε ακούγοντα την προηγούμενη συζήτηση είναι το γεγονό ότι κάποιε φορέ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντί να καθησυχάζει και να ηρεμεί του πολίτε το αντίθετο κάνει, προκαλεί ανησυχία και φόβο. Γιατί πρέπει να σας πω ότι επειδή σημείωνα κάποια πράγματα, μία από τις λέξεις που ακούστηκε τις περισσότερες φορές στην προηγούμενη συζήτηση ήταν η λέξη παράνομη, παράνομη μετανάστευση, μαύρη εργασία. Νομίζετε ότι με αυτή την οδηγία θα επιλύσουμε τα προβλήματα της μαύρης εργασίας και της λαθρομετανάστευσης. Γι' αυτό έχουμε αυτή την οδηγία. Γιατί μιλάμε για αυτά τα ζητήματα εδώ, αν δεν είναι αυτό ο στόχο οδηγία, αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ. Εμεί από την ΕΤΟΚ συνεχίζουμε να τονίζουμε την αοριστία, την ε, αμφισημία των πολιτικών. Υπάρχουν διάφορες ταχύτητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα έχουμε την οδηγία για τους εποχιακούς εργαζομένου, ε, την ε, οδηγία που έχει ως στόχο να έχουμε μία μεν εποχιακή αλλά κάπως βιώσιμη ε, μετανάστευση. Επίσης έχουμε πιέσεις από μεταναστευτικά ρεύματα, κάτι που οδήγησε τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών να θεωρούν από τράγους τράγους ε, για την ε, πολιτική ε, στρατηγική τους μετανάστες. Πρόκειται για μια σχιζοφρένεια. Πάρα πολύ όμως επικίνδυνη για το μέλλον της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Επίσης, κάτι άλλο που διαπιστώνουμε στη συζήτηση για την ενιαία άδεια που έχει συζητήσει το Κοινοβούλιο και ψήφισε μάλιστα το Μάρτιο ή πουλά θα κατακαιρματιστεί ακόμη περισσότερο η αγορά εργασίας. Ιδίως τη στιγμή που βιώνουμε μία άνευ προηγουμένου κρίση, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην έναυση συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων μεταξύ των ίδιων των εργαζομένων. Γι' αυτό νομίζουμε ότι για μια ακόμη φορά η ευθύνη των ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι και προφανής πολιτική κίνδυνη. Για την ΕΤΟΥΚ είναι προφανές επίσης, όπως το έχουμε πει και επαναλάβει και θα το ξαναπούμε τώρα που ξεκίνησαν και αυτές οι εργασίες, έχουμε την έννοια της ισότιμης μεταχείρισης, της εφαρμογής του δικαίου της χώρας ε, διαμονής. Μιλάμε για συνοδευτικές κοινωνικές πολιτικές για πολίτες επικώς τρίτων χωρών. Όλα αυτά πρέπει να είναι τα βασικά στοιχεία που θα αποτελούν γνώμονα για όλη αυτή τη διαδικασία. Η οδηγία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να βοηθήσει τελικά στο να προσλαμβάνεται φθηνό εργατικό δυναμικό σε βάρος του ε, εργατικού δυναμικού της ίδιας της χώρας. Οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές πραγματικά ανησυχούν για την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα. Η σύνδικη της Ρώμης την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και ε, υπηρεσιών τη θεωρούσε μία από τις σημαντικότερες ελευθερίες, αλλά μετά σήμερα τις αποφάσεις ε, του ΔΕΚ για τις Λαβάλ, αποφάσεις Ρουφ κτλ και μετά τις προτάσεις Κομισιόν, η οποία συνεχίζει να επιμένει να νομοθετεί με στόχο ε, την πρόθεση της, ε, του αθέμητου ανταγωνισμού τελικά μέσα στην εσωτερική αγορά, τελικά υπονομεύεται η ισότιμη μεταχείριση των εργαζομένων και διαβρώνεται η αρχή της υποδοχής στην χώρα που κάποιος διαμένει, που κάποιος διαβεί. Ακριβώς ε, αντιθέτως εμείς πιστεύουμε ότι με τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας η οποία εγγυάται μια κοινωνική οικονομία της αγοράς κοινωνική οικονομία της αγοράς και μεγαλύτερο πρωταγωνιστικό ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομίζω ότι πρέπει να εργαστούμε ώστε η κοινωνική πρόοδο και ο σεβασμό στη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων που εγγυάται με το άρθρο 20 την ισότητα και με το άρθρο 21 τη μη διακριτική μεταχείριση θα πρέπει να είναι μια πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την οδηγία λοιπόν για τους εποχιακούς εργαζομένους, αυτή η οδηγία πρέπει να αφορά όλους τους εργαζόμενους, όχι μόνο τους εποχιακούς. Υπενθυμίζουμε ότι τα μεγάλα σκάνδαλα τα οποία ανακάλυψε ο τύπος στην τελευταία χρονική περίοδο αφορούσαν την Ιταλία όπου Πολωνοί και Βούλγαροι εργάτες πραγματικά δουλεύουν υπό καθεστώ δουλεία, σαν σκλάβοι. Επομένω, πρέπει να δούμε ευρέω ε, το θέμα αυτό των εποχιακών εργαζομένων και όχι μόνο των εποχιακών ε, αλλοδαπών εργαζομένων. Η αποτελεσματικότητα των νόμων λοιπόν πρέπει να αποτελέσει ένα ακόμη θεμελιακό στοιχείο τη όλη αυτή ε, προβληματική. Βλέπω ότι δεν έχω καθόλου σχεδόν χρόνο, οπότε συνοψίζω κύριε Πρόεδρε. Αυτό που θέλουμε εμείς να προτείνουμε με βάση αυτή την πρόταση είναι κάτι επαναστατικό, κάτι ρηξικέλευτο. Η Επιτροπή πρέπει να κάνει καλύτερα τη δουλειά της. Γιατί εδώ μιλάμε ουσιαστικά για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας για πολίτες. Είτε προέρχονται από τρίτες χώρες είτε όχι. Και ποιος ενδιαφέρεται περισσότερο για τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας, τα συνδικάτα και οι επιχειρηματίες, οι εργοδότες. Η Κομισιόν τώρα και την οδηγία αυτή αλλά και την οδηγία για την ενιαία άδεια την έχει βάλει από την πίσω πόρτα και από το παραθυράκι. Δεν είχε διαβουλεύσεις μαζί μας. Δεν ζητήθηκε η άποψή μας. Και νομίζω ότι και εσείς ουσιαστικά ως κοινοβούλιο αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πείτε στην Επιτροπή κύριοι και κυρίες της Κομισιόν εσείς πρέπει να ρυθμίσετε το θέμα της εποχιακής εργασίας συνολικά, όχι μόνο σε αφορά τους αλλοδαπούς εποχιακούς εργαζομένους και πρέπει να συνομιλήσετε και με τα συνδικάτα και με τους εργοδότες για να έχουμε μια δομή που θα μας δώσει εργαλεία στα χέρια μας για να λύσουμε τα προβλήματα, όχι να γεννήσουμε και άλλα προβλήματα. Η κυρία Ρομέρο το είπε πάρα πολύ καλά ήταν ε, από του λίγου που μίλησε για τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, συνδικάτων κτλ. Γιατί ίσω γνωρίζει πολύ καλύτερα την Ανταλουσία, την περιοχή της, οι εργοδότε, τα συνδικάτα, οι κοινωνικοί εταίροι δηλαδή. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με τι διοικητικέ αρχές για να ρυθμίσουμε ένα σωρό ζητήματα και εμπειρίες ε, που εμείς έχουμε βιώσει και που θα πρέπει να τις ε, έχει υπόψη και η Κομισιόν. Λοιπόν, πέρασε ο χρόνος μου. Θέλω να σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας και γιατί επιχειρήσατε να μείνετε στο χρόνο που είχαμε ορίσει για να ολοκληρώσουμε αυτή τη δεύτερη συζήτηση, αλλά να μείνει χρόνος και για τη συζήτηση με όσους βουλευτές θα ήθελα να κάνουν κάποιο σχόλιο. Θα ακούσουμε τώρα το δεύτερο ομιλητή μας, τον κύριο Σβέρκερ Ρούντεμπεργκ, πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας σχετικά με τη μετανάστευση και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Ο κύριος Ρούντεμπεργκ προέρχεται από τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων, το Business Europe. Χαίρομαι κύριε Ρούντεμπεργκ που είστε εδώ και σας παρακαλώ και εσείς να έχετε υπόψη σας ε, το χρόνο. Thank you very much. As said, my name is... Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο Σβέρκε Ρούντεμπερκ, και εκπροσωπώ τη Business Europe, ε, τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων για τη μετανάστευση και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Θα σας αφήσω και το PowerPoint την παρουσίαση που έχω προετοιμάσει, αλλά επίση και το έγγραφο θέσεώ μα για το θέμα των εποχιακών εργαζομένων. Όταν βλέπει κανείς την προτινόμενη οδηγία, νομίζω ότι πρέπει κανείς να απαντήσει δύο ερωτήματα για να καταλήξει στα ακατάλληλα συμπεράσματα. Το πρώτο ερώτημα είναι η ανάγκη για εποχιακούς εργαζομένους είναι ε, θεμητή. Επίσης, θέλουμε η εποχιακή εργαζόμενη να είναι νόμιμη ή παράνομη. Τα ερωτήματα αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία ότι οι εταιρείε ε, έχουν ανάγκε σε ολόκληρη την Ευρώπη ε, εποχιακών εργαζομένων για να καλύψουν τις τοπικές ε, ανάγκες τη αγοράς εργασίας και όπως είπε και η κυρία Βαντάση, Υπάρχει το θέμα του τι είναι εποχή και επίσης οι ανάγκες ποικίλουν ανάλογα με του τομεί. Είναι κάτι το οποίο το είπε και ο κύριο Κοφεράτη. Όμως ε, είναι γεγονός ότι χρειάζονται εργαζομένους. Ε, υπάρχει ένα πρόβλημα λοιπόν εξέβρεσης νομίμων εργαζομένων. Δεν είναι, ένα πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα να βρει κανείς παράνομους ε, εργαζομένους, αλλά η παράνομη εποχιακή ε, χρησιμοποιούνται σε τέτοιο βαθμό τελικά αυτοί που έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα είναι αυτοί που θέλουν να ε, που έχουν τη διάθεση να προσλάβουν παράνομους ε, εργαζομένους. Όμως εμείς θέλουμε αυτό να μπορεί να γίνεται υπό νόμιμες ε, συνθήκες, να γίνεται νόμιμα. Και αυτό έχει να κάνει και με τα δικαιώματά τους, γιατί αυτό που ξεχνάμε συχνά είναι ότι αυτοί που είναι σε μια δύσκολη κατάσταση είναι οι παράνομοι εργαζόμενοι. Αυτοί την κάνουν εκμετάλλευση. Και αν δείτε για παράδειγμα την, την οδηγία η νομοθεσία του κράτους μέλους ισχύει, αλλά ανεξαρτήτως από την, εφαρμό, από την ισχύω νομοθεσία υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα ο μισθός των ανθρώπων αυτών και αυτό συνδέεται, συγκρίνεται με το μισθό των παρανόμων εργαζομένων που είναι εντελώς διαφορετικό. Αν δει για παράδειγμα την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει εναρμονισμένε και ταχείες διαδικασίες ε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε μια άλλη χώρα, θέλουν να βρουν μια δουλειά και είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η εναρμόνιση. Λόγω της φύσης της ε, η εποχιακή εργασία πρέπει να, καλύπτεται η εργασία, πρέπει να καλύπτει την εργασία πριν τελειώσει η εποχή και γι' αυτό οι διαδικασίες πρέπει να είναι πάρα πολύ ταχείες. Και όπως είπα, πρέπει να είναι ευκολότερο, πρέπει να είναι πιο δυνατό να είναι κανείς ένας ε, νόμιμος εργοδότης εποχιακού εργαζομένου και όχι με τίμημα να μην γίνεται η δουλειά, γιατί ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται. Θέλουμε να γίνει η δουλειά που χρειάζεται να γίνει. Και επιπλέον όταν μιλάμε για τη μεταναστευτική πολιτική γενικότερα, όλοι είναι υπέρ ε, της μετανάστευσης ε, των υψηλά ε, ειδικευμένων, αλλά πολύ λίγοι έχουν τη διάθεση να καλύψουν τις ανάγκες και να εκπροσωπήσουν τους εργαζομένους χαμηλότερης ειδίκευσης. Αν δει τη μεταναστευτική πολιτική για τους εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης, είναι σαν να τους αφήνουμε στην άκρη για να μπορούν ε, να προσληφθούν παράνομα. Δεν έχει νόημα λοιπόν, δεν υπάρχει νομιμότητα μια ευρωπαϊκής πολιτική που περιορίζεται σε τέτοια μέτρα. Χρειαζόμαστε μια οδηγία η οποία καθιστά σαφές το ότι οι χαμηλή ειδικεύσεις εργαζόμενης ε, με να, υπάρχουν, να έχουν την νόμιμη δυνατότητα να ε, ε, εργαστούν σε αξιοπρεπείς συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν υπάρχει ζήτηση θα υπάρχει και προσφορά και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να καλυφθεί νομικά. Όταν βλέπει κανείς την ίδια την οδηγία να σας πω ποια είναι η άποψή μας σε σχέση με τις λεπτομέρειες. Καταρχάς, δικαίως ε, ότι ο γενικός κανόνας είναι ο νόμος του κράτους μέλους και του εργοδότη αλλά βέβαια πρέπει να καλύπτονται και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Κάτι το οποίο επίσης είναι σωστό και νομίζω το είπε ο κύριος Κοφεράτη, ότι σωστό είναι να γίνεται μια προαιρετική εξέταση της ανάγκης της τοπικής αγοράς, ε, γιατί μερικές φορές υπάρχει φοβερή γραφειοκρατία ε, με δεδομένα πολύ παροχημένα και τα οποία δεν είναι τα κατάλληλα. Δεν είναι αυτά που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να, για να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματική ανάγκη για εργασία. Όμω στην οδηγία υπάρχει μια διάταξη που λέει ότι μπορεί το κράτο μέλο να απορρίψει μια αίτηση βάσει βάση του αριθμού ε, ε, των εισδοχών. Σωστό είναι αυτό, αλλά όταν μιλάμε για την αγορά εργασίας αναφέρεται μετά δραστηριότητα ανάλογα με την εποχή. Κάτι το οποίο αφορά όμως ε, περιπτώσεις που είναι πολύ παραπάνω και εμείς θέλουμε αυτό το πολύ παραπάνω να διαγραφεί. Τώρα, Οι περισσότερες χώρες, αν όχι όλες, έχουν κάποιους ε, κανόνες που αφορούν τους εποχιακούς εργαζομένους. Είναι και διαφορετική η διάρκεια της εποχής ε, σε κάθε κράτος μέλος και γι' αυτό υπάρχει η νομοθεσία που δίνει τη δυνατότητα μετανάστευσης ε, εργαζομένων για εννέα μήνες και όχι για έξι. Στην οδηγία πρέπει να παραμείνουμε στις έξι μήνες, αλλά τα κράτη-μέλη που έχουν μεγαλύτερης διάρκειας ε, εποχής ε, και έχουν καλύτερες διατάξεις θα έπρεπε να έπρεπε πιο ευνοϊκές, θα έπρεπε να μπορούν να τις διατηρήσουν και αυτό δεν αναφέρεται στην οδηγία. Είναι σαν να λέτε λοιπόν στην Ισπανία ότι λάθος κάνετε, η εποχή σας δεν είναι νέα μήνες, είναι έξι μήνες. Οπότε πιστεύω ότι υπάρχει και ένα θέμα επικουρικότητας. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι πίσω από την έννοια της εποχικής εργασίας δεν πρέπει να μπερδεύουμε την νόμιμη και την παράνομη εργασία όταν μιλάμε για τη συγκεκριμένη κατάσταση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γιατί μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την νομοθεσία των κρατών μελών και έχουν και τα βασικά δικαιώματα του άρθρου 16. Δεν ε, μπαίνουν δηλαδή σε μια επικράτεια στην Αγριά Δύση. Μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχει, ένα που υπάρχει μια συγκεκριμένη νομοθεσία, αν και για το συγκεκριμένο θέμα δεν υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Τζουλιάνα Μεσίνα, που είναι επικεφαλή του τμήματο Πολιτικών Μετανάστευσης της Ιταλικής CGIL, Ομοσπονδία Εργαζομένων. Αν μπορείτε κι εσείς να τηρήσετε τα πεντε λεπτά, 5-6 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επιτροπή που μου έδωσε τη δυνατότητα να εκφράσω και εγώ την άποψη της ε, δικής μου της ε, Ομοσπονδίας που εντάσσεται στην, που είναι η CGL και εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία γενικότερα. Εμείς ασχολούμεθα με τον τουρισμό μεταξύ άλλων. Η πρόταση οδηγίας για τους εποχικούς εργαζόμενους ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η πρόταση αυτή δείχνει ότι το φαινόμενο της ε, εποχιακής εργασίας ε, έχει λάβει ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις. Η Ιταλία είναι μια χώρα με εξωτερικά σύνορα και αυτές ακριβώς Εβδομάδε εβδομάδες ζει την αντίφαση στο πετσί της, μια αντίφαση που προκύπτει από το εποχιακό φαινόμενο. Μιλάμε για 5 εκατομμύρια μετανάστες ε, που έχουν φτάσει στην Ιταλία, ένας αριθμός ο οποίος περιλαμβάνει και τους νόμιμους και τους ε, περίπου 550.000 ε, παράνομους εισαγωγικά. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να εξτάσει κανείς ε, το φαινόμενο κάτω από το πρίσμα ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί θα είχαμε αρνητική δημογραφική εξέλιξη στην Ιταλία. Επίσης θεωρώ ότι στην η Ιταλία πρέπει να υποθεί ότι στην Ιταλία οι μετανάστες εργαζόμενοι συμβάλλουν σημαντικά στο ΑΕΠ περίπου κατά 12% ή αν θέλετε με 33 δισεκατομμύρια φόρο εισοδήματος που καταβάλουν. Και εδώ εξαιρείται η μαύρη εργασία και η αδήλωτη εργασία. Πάνω από τα 2 τρίτα των μεταναστών εργαζομένων απασχολούνται στον τριτογενή τομέα. Και ε, εδώ επικρατούν τα εποχιακά επαγγέλματα όπως είναι στον τομέα των κατασκευών και στον τομέα των ξενοδοχείων. Μάλιστα ε, στην Γεωργία και στον τουριστικό τομέα έχουμε περισσότερους εποχιακούς από ε, άλλους εργαζόμενους. Κάθε χρόνο στην Ιταλία διαπιστώνεται καταρχήν η ζήτηση και η ανάγκη που υπάρχει για εργαζόμενους αλλά με ένα αποστασιοποιημένο τρόπο. Για το 2011 ε, αναφέρθηκε ότι επιτρέπεται είσοδος 60.000 μεταναστών εργαζομένων για να απασχοληθούν αυτοί στην γεωργία και στον τομέα των ξενοδοχείων. Όμως ε, με τον τρόπο αυτό υποτιμούν την πραγματικότητα και αν θέλετε και ορίζοντας αυτό χαμηλό αριθμό δεν εκφοβίζουν τους υπόλοιπους να έρθουν με αποτέλεσμα αποτέλεσμα να καταλήγουμε στην εκμετάλλευση που είναι μια τραγική πραγματικότητα στο γεωργικό τομέα. Εξάλλου, Μιλάμε κυρίως ε, για εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται σε Ιταλικό έδαφος και οι οποίοι εμπλέκονται σε μια τεράστια γεωγραφική ταλαιπωρία. Στην Ιταλία υπάρχει μια πολιτική ε, απόθεση και από την άλλη υπάρχει μια πολιτική που λέει ότι πρέπει να έρθουν περισσότεροι εργαζόμενοι για να καλυφθεί η ζήτηση. Εδώ λοιπόν εντάσσεται η πρόταση οδηγίας που αφορά στην εποχιακή απασχόληση. Εμείς βλέποντας την οδηγία αυτή καταλήγουμε στο ότι τελικά τα πράγματα μπορεί να γίνουν ακόμα χειρότερα. Πιο συγκεκριμένα η οδηγία ορίζει τις προϋποθέσεις εισόδου εργαζομένων από τρίτο χώρες και η οδηγία προβλέπει Βλέπει διαφοροποίηση ανάμεσα σε εποχιακούς και μη εποχιακούς εργαζόμενους, οι οποίοι όμως κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Άρα με τον τρόπο αυτό παραβιάζεται η αρχή για την ίδια εργασία, ίδια αμοιβή. Και με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για το κοινωνικό ντάμπινγκ και για την περαιτέρω υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας. Ο ορισμός της εποχιακής εργασίας είναι πάρα πολύ γενικός και δεν ε, ε, προβαίνει σε ορισμούς για σημαντικούς τομείς. Παραδείγματο χάρη, ε, ο ορισμός ε, του εποχιακά εργαζόμενου των 6 μηνών είναι σε αντίφαση με αυτό που ισχύει στην Ιταλία που είναι 9 μήνε και είναι ε, κάτι που ισχύει κυρίω στη Γεωργία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ορίσουμε τα επίμαχα σημεία της οδηγία, να προσπαθήσουμε βέβαια να δώσουμε απαντήσεις στην ζήτηση που υπάρχει, αλλά παράλληλα να αποφύγουμε να υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία διακρίσεων. Παραδείγματο χάρη, ε, όταν μιλάμε για την έκδοση άδεια, ε, πολλές φορές ε, υπάρχει η περίπτωση όπου μερικοί λαμβάνουν ειδοποίηση απέλαση, άλλοι πάλι όχι. Ο ορισμός λοιπόν των περιπτώσεων όπου ισχύουν κυρώσει, είναι ένας ορισμός πάρα πολύ γενικός και δεν πείθει κανένα γιατί δεν είναι και σαφή οι διατάξεις για την απόρριψη ή την ανάκληση άδεια του εργαζομένου όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας όπως αυτές ορίζονται στην νομοθεσία ή σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εδώ θέλουμε να πούμε ότι δεν υπάρχει ένα σύστημα το οποίο να είναι δεσμευτικό, να αποδίδει ε, στις συλλογικέ συμβάσεις δεσμευτική μορφή έναντι όλων, το περίφημο εργαόμνες κατόπιν τούτου είναι καθοριστική σημασία να υπάρχει μια δέσμευση όσον αφορά την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων για να μην υπάρξουν και άλλα φαινόμενα εκμετάλλευσης, ε, ε, στιγνής εκμετάλλευσης σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι εργοδότες ε, πρέπει να αποδείξουν ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν ικανοποιητικό κατάλημα και συνθήκες εργασίας. Μάλιστα πρέπει εφόσον καταβάλλεται νίκιο, το νίκιο αυτό να μην είναι υπερβολικό. Όμως δεν υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος και τελικά αυτό μοιάζει είναι απλά λόγια. Ε, μεταξύ άλλων θέλω να σας πω είναι ντροπή το ότι ο εργαζόμενος ε, ε, πρέπει να πληρώνει πολλές φορές υψηλό ενίκιο για ένα κατάλημα που το προσφέρει ο ίδιος εργοδότης. Μεταξύ άλλων πρέπει να σας πω δεν υπάρχει καμία δυνατότητα κατοχύρωση των εποχικά εργαζομένων. Και αυτό εμάς ως συνδικαλιστικό φορέα μα ενδιαφέρει πάρα πολύ για όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από την ε, ηθαγένειά του. Υπάρχει συλλογική ε, σύμβαση για τον τουρισμό και εκεί προβλέπεται ότι ε, εάν υπάρξει πρόσληψη περαιτέρων εποχικών, δεν ρυθμίζεται το θέμα της ηθαγένειας. Και τι θα γίνει αν όμως χρειαστεί να προσληφθούν περαιτέρω εποχιακοί εργαζόμενοι, Μαζί λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων, εμεί ω CGL, Ιταλικό Συνδικάτο, ζητήσαμε να υπάρξει τροποποίηση οδηγία για την ενιαία άδεια, μια οδηγία που περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενου, κυρίω και τους εποχικούς που προέρχονται από τρίτε χώρε και ε, προσωπικό ε, που ε, έχει μεταφερθεί μέσα στην ίδια την επιχείρηση. Βέβαια αυτά δεν συνέβησαν, όμως εμείς εξακολουθούμε να θέλουμε να υπάρχει η ίδια αμοιβή για την ίδια εργασία και αυτό να ισχύει και για τους κοινοτικούς και τους εξοκοινοτικούς εργαζόμενους. Σήμερα οι επιχειρήσεις δεν έχουν καμία δέσμευση όσον όταν απασχολούν εξοκοινοτικούς εργαζόμενους. Γι' αυτό λοιπόν τους λόγους και λόγω του ότι υπάρχουν πάρα πολλά επίμαχα σημεία που αυτή την οδηγία, εμεί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να ότι δεν είναι δυνατόν εμείς να δεχτούμε μία νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να περιλαμβάνει διακρίσεις ει βάρο των επιχειρηματικά εργαζομένων από τρίτες χώρες και σε νομικό και σε πρακτικό επίπεδο. Εξάλλου, όσον αφορά την ε, προσχώρηση στην αγορά εργασία δημιουργείται ένα διπλό καθεστώς γιατί δεν υπάρχουν αποτελεσματικοί έλεγχοι και αποτελεσματικές κυρώσεις. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να ξαναξεκινήσει η συζήτηση για το να ανοίξουν νόμιμες δίωδοι ως προς την απασχόληση, να μην περιοριζόμαστε μόνο σε εξειδικευμένους εργαζόμενους και να ξεπεραστεί αυτή τη στιγμή αυτή η διάταξη που αφορά στην ε, ασφάλεια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά την άποψή μα, οι νομοθεσίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίω όσον αφορά τα θέματα των δικαιωμάτων, δεν πρέπει να βασίζεται μόνο σε διακρίσει, αλλά στη βασική αρχή για την ίδια εργασία, η ίδια αμοιβή και ανεξάρτητα από το ποια εργασία κάνουν οι εργαζόμενοι. Ω εκ τούτου, οι πρώτε οδηγίε θα πρέπει να περιλαμβάνει και τι διορθώσει που έχουμε προτείνει. Γιατί αλλιώ, αν δεν γίνουν δεκτέ αυτέ οι διορθώσει, εμεί θα παραμείνουμε αντίθετοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Χέλεν Χόφμαν, Σύμβουλα Επικοινωνικών Θεμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Παρακαλώ να λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο και θέλουμε να έχουμε και συζήτηση. Και δυστυχώς έχουμε μείνει πολύ πίσω. Έχετε το λόγο. Πρώτα απ' θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από την ΟΕΑΠΜΕ και σας κύριε Πρόεδρε αλλά και τον κύριο Μωράς που μας καλέσατε σε αυτή την ακρόαση. Επειδή είμαι η τελευταία ομιλήτρια θα έρθω κατευθείαν στο θέμα, στην ουσία του θέματος. Εμείς ε, καλωσορίζουμε και το πεδίο εφαρμογή αλλά και το στόχο της πρόταση αυτή για του εποχιακού εργαζομένου που έχει ω στόχο τη θέσπιση μια κοινή διαδικασία για την είσοδο και για την διαμονή υπηκών τρίτων κρατών που απασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως εποχιακοί εργάτες. Ε, εν γέννη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται και να προσελκύσουν αλλά και να προσλάβουν εργαζόμενους, μεταξύ αυτών και εποχιακούς εργάτες, σε πολλούς τομείς. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι αυτή η νέα πρόταση θα βοηθήσει να υπάρξει καλύτερη αντιστοιχία της προσφοράς και της ζήτησης ε, και αυτό θα συμβάλλει σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και θα δημιουργήσει πιο διαφανείς ε, κανόνες. Συμφωνούμε κυρίως ότι αφορά δύο τομείς. Πρώτα απ' όλα τον ορισμό εποχιακός εργαζόμενος και δεύτερον ότι αφήνεται στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν ποιοι είναι οι τομείς που πληρούν τα κριτήρια για εποχιακή εργασία. Εγκρίνουμε επίσης ε, την ε, διαδικασία της ενίας ε, αίτησης και την διευκόλυνση της επανιστοχής. Έτσι, οι επιχειρήσεις, ε, οι εργοδότες θα έχουν ε, περισσότερη ασφάλεια δικαίου και θα μπορούν και οι χώρες να επωφεληθούν εργατικού δυναμικού το οποίο έχει αποδείξει ότι έχει ικανότητες και επομένω θα επιτρέπεται να υπάρχει αυτή η συνέχεια και για τον εργοδότη αλλά και για τον απασχολούμενο. Τούτου λεχθέντος παρόλα αυτά νομίζουμε ότι χρειάζεται βελτίωση ή διασαφήνιση σε κάποιους τομείς. Η πρόταση θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να περιπλέκει περισσότερο τα πράγματα για τους εργοδότες ε, σε σχέση με αυτά που προβλέπονται για την υποχρέωση παροχής καταλήματος. Υποχρέωση που βαρύνει τους εργοδότες. Φυσικά και συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα κατάλληλο επίπεδο διαβίωσης και κατάλληλη στέγαση, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να είναι καθήκον των εργοδοτών διότι αυτό θα, θα αυξήσει πολύ το εργασιακό κόστος και έχει να κάνει και με την ιδιωτική σφαίρα και των εταιρείων και των εργαζομένων. Και νομίζουμε ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα να δυσκολευτούν ακόμη περισσότερο οι ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προσλάβουν τους τόσο αναγκαίους για, αυτούς, ε, για αυτές εποχιακούς εργαζομένους. Θα πρέπει επίσης οι διατάξεις να είναι πιο ευέλικτες ε, σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της διαμονής ε, και να λαμβάνεται υπόψη το τι ισχύει ήδη σε κάποια κράτη-μέλη. Επίσης ο περιορισμός σε ένα ημερολογιακό έτος νομίζω ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Γιατί δεν είναι τόσο ξεκάθαρε ε, οι εποχέ, οι διακρίσει μεταξύ των εποχών. Υπάρχουν μεγάλε παραλλαγέ και διαφορέ. Ανάλογα με το πώ η τουριστική περίοδος, η εποχή ε, αντιλαμβάνεται, να αντιλαμβάνεται το ένα κράτος μέλος ή το άλλο. Από ό,τι προβλέπετε μέχρι είσαι σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, μπορεί να αρνηθεί ένα κράτος μέλος μια αίτηση αν έχει τιμωρηθεί ο εργοδότης για δήλωτη εργασία ή παράνομη απασχόληση. Θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα στην ε, πρώτη ε, στο πρώτο παράπτωμα, στην πρώτη παραβίαση, παράβαση εκ μέρους του εργοδότη αυτή, αυτό το μέτρο, αλλά μόνο όταν αυτό επαναλαμβάνεται και με βάση του εθνικούς νόμους πάντοτε. Επίσης, θα πρέπει να είναι ένα λογικό ανάλογα με το είδος της παράβασης, το είδος του αδικήματος. Τέλος, εμείς δεν είμαστε υπέρ της δυνατότητας αλλαγής εργοδοτών, εργοδότη. Και αυτό για τον πολύ απλό λόγο ότι θα μπορούσε να επιτρέπει το να παρακάμπτονται κάποια πράγματα και επίση η διαχείριση αλλά και ο σχεδιασμός ε, για το εργατικό δυναμικό το εποχιακό θα γίνει ακόμη πιο δύσκολο για τους εργοδότες. Ένα τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι η πρόταση για τις ενδοεπιχειρησιακές, μεταθέσει, μεταθέσεις συστηθεί δηλαδή το απόγευμα. Είναι μια οδηγία που πιο πολύ αφορά μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά θεωρούμε ότι μπορεί να επηρεάσει αρνητικά και τις μικρές ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις βιοτεχνίες σε κάποιους τομείς, όπως οικοδομή για παράδειγμα. Και ναι μεν συμφωνούμε με το πεδίο εφαρμογή τη ε, πρόταση αυτή για τις ενδοϊπηρεσιακές μεταθέσει, αλλά θα θέλαμε να υπάρξουν κάποιε προσαρμογέ. Τρει κυρίως τομεί πρέπει να καλύπτονται. Πιο περιορισμένο ο ορισμό του ειδικού μεγαλύτερη τήρηση της συμφωνίας GATS και πιο, σημαντικ, πιο πολλά ακαδημαϊκά προσόντα ή μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία. Πέντε χρόνια. Επίσης, τα κριτήρια ε, αποδοχής θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικά για να μην έχουμε κάποιες παρατυπίες ή ατασταλίες, όπως οι λεγόμενες letterbox companies. Και τέλος, θα πρέπει να ενισχυθούν ε, οι όροι για τη γεωγραφική κινητικότητα μεταξύ κρατών μελών για να μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη συμμόρφωση προς την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ανοίξει η συζήτηση. Μπορείτε να πάρετε το λόγο, να κάνετε σχόλια. Όπως είπα και προηγουμένως, ε, η ενδοεπηρεσιακός μετατιθέμενη θα είναι το θέμα μας το απόγευμα, οπότε παρακαλώ ε, επικεντρώστε τις ερωτήσεις σας στους εποχιακούς εργαζομένους, που είναι το θέμα μας για σήμερα το πρωί. Οπότε, άρχεται η συζήτηση, ο κύριος Μπουσούτιλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση Υπάρχουν κάποιες ε, κατηγορίες ε, και πρόκειται για το πεδίο εφαρμογής της ε, οδηγίας. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες εργαζομένων και θα ήθελα να μου πείτε για αυτές τις κατηγορίες κατά πόσο θα πιστεύετε ότι θα έπρεπε να καλύπτονται. Για παράδειγμα, άνθρωποι που ήδη νομίμως διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να καλύπτονται από την οδηγία αυτή. Και υπάρχει επίσης μια κατηγορία ανθρώπων που παρανόμως διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η οδηγία θα μπορούσε να τους δίνει μια δυνατότητα νομιμοποίησης αντί να, παραμείνει, να παραμένει κρεμίσι η κατάστασή τους όπως ισχύει τώρα. Πιστεύουν λοιπόν οι ομιλητές ότι αυτές οι κατηγορίες ε, των εργαζομένων θα έπρεπε να καλύπτονται στο πεδίο εφαρμογή της ε, οδηγίας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρομέρο Λόπεθ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε σχέση με τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους που θα έπρεπε να είχε κάνει η Κομισιόν στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας. Δεν ξέρω εάν ε, είναι ένα προπατορικό αμάρτημα αυτό, ε, μπορεί να λυθεί τώρα ή όχι, γιατί έχουμε ήδη την οδηγία. Πράγματι όμως όταν υπάρχει τέτοιου είδους ε, πρόταση πρέπει να έχει προηγηθεί διαβούλευση ώστε το κείμενο να την χάνει μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή. Τώρα έχουμε το κείμενο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς τώρα στο Κοινοβούλιο είναι να τροποποιήσουμε αυτό το κείμενο και με το, μέσω των τροπολογιών μας να προσθέσουμε στο κείμενο αυτά που δεν έκανε η Κομισιόν, χάρη στο διάλογο που μπορούμε να έχουμε εμεί εδώ με του κοινωνικού αφού δεν τον έκανε το διάλογο αυτό η Κομισιόν. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλύτερο να έχουμε δύο οδηγίες ή θα αρκούσε μία οδηγία όπως αυτή που έχουμε επιτάπητος. Δηλαδή μία να είναι για τους αλλοδαπούς εργαζομένους και μία να είναι για τους Ευρωπαίους εργαζομένους, πάντα στο πλαίσιο της εποχιακής εργασίας. Μία πρώτη πολύ σημαντική επιλογή που έχει θέσει η Κομισιόν ως πρόταση, ε, στην πρότασή της. Ε, εγώ αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης ε, των ευρωπαϊκών συνδικάτων προς ξένα χέρια, εργατικά χέρια από ξένες χώρες. Και αυτό είναι λογικό γιατί έχουμε το ζήτημα του dumping και έτσι είναι τα πράγματα. Δεν έχουμε φθηνό εργατικό δυναμικό φθηνά εργατικά χέρια, αλλά και στην ίδια την ισπανική ορολογία έχουμε δύο λέξεις που λένε το ίδιο πράγμα ακριβώς Έχουμε το τεμπορέρο που αφορά τους εργαζομένους, τους εποχιακούς στην εργασία και το temporal που είναι για τον εργαζόμενο τον εποχιακό στον τουρισμό. Και ενώ είναι το ίδιο πράγμα, μιλάμε, έχουμε δύο διαφορετικές λέξεις. Ε, επί της ουσίας ε, υπάρχει ένα ζήτημα κοινωνικό, κοινωνικής βάσης, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να το πάμε και στο συνδικαλιστικό επίπεδο δεν μπορούμε να έχουμε συνδικάτα μόνο για τους Ευρωπαίους, γιατί αν υπάρχουν συνδικάτα μόνο για τους Ευρωπαίους, τότε οι εργαζόμενοι που έρχονται από τρίτες χώρες, ποιος θα τους προστατεύσει αυτούς τους εργαζομένους, όχι τα συνδικάτα της χώρας καταγωγής ή προέλευσής τους, άρα Υπάρχει αυτή η καχυποψία και αυτή η δυσπιστία που πρέπει όμως να καταπολεμηθεί στο επίπεδο των συνδικάτων. Και για να έχουμε μεγαλύτερη και να διευκολύνουμε την νόμιμη πρόσληψη θα πρέπει να έχουμε καλύτερη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και να δημιουργήσουμε σε αυτές τις χώρες προέλευσης οργανισμούς, φορείς. Και νομίζω ότι πραγματική, η πραγματιστική προσέγγιση για την οποία έκανε λόγο εκπρόσωπος της Κομισιόν ε, αυτό που έχει ε, καταφέρει να δημιουργήσει ένα κενό, ένα πλήρες κενό το γερμανικό θαύμα της δεκαετίας ε, του 60 και του 70 ήταν γιατί υπήρξε μια ρεαλιστική διαχείριση. Οι Ισπανοί εργαζόμενοι και σε καθεστώς δικτατορίας μάλιστα από το Σοσιαλδημοκρατική τότε γερμανική κυβέρνηση ε, υπήρξε αυτή η διαχείριση αυτών των εργαζομένων. Και δεν είχαμε το καθεστώς και αυτή την κατάσταση δουλείας που βλέπουμε σε πολλές χώρες. Δεν υπάρχουν ε, διμερείς συλλογικές συμβάσεις. Φυσικά διαφέρει, ε, θα διαφέρει η κατάσταση στην Ιταλία αν υπήρχαν πιο πολλές διμερείς συλλογικές συμβάσεις ή ε, σε συνταλεί σε άλλες χώρες. Η Κομισιόν μέχρι τώρα έχει εστιάσει ε, ε, στην ουσία, αλλά δεν έχει κάνει μια ρεαλιστική προσέγγιση. Ευχαριστώ. Κυρία Σαρτζεντίνη. Dank Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων ε, επιθυμεί ρύθμιση Και μάλιστα αυτή η ρύθμιση να καλύπτει εξίσου τους ε, ενδοκινοτικούς και τους εξοκινοτικούς εποχιακούς εργαζομένου. Νομίζω όμω ότι υπάρχει μία παρεξήγηση σε σχέση με αυτούς τους εποχιακούς στην Ευρώπη. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν το εξή. Οι διατάξεις για τους εποχιακούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο κακοί, ώστε να μην υπάρχει καν έλεγχος του τόπου εργασίας ε, και της εφαρμογής των κανόνων εργασίας, γιατί το βασικό στοιχείο, αν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε σε κάποιον ελάχιστο κανόνα, πώς θα εφαρμοστεί πράγματι ο κανόνας αυτός, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα προσλαμβάνονται οι άνθρωποι αυτοί νόμιμα και όχι παρανόμως μπορούμε μόνο αν υπάρχει μία κύρωση για όσους δεν σέβονται τους ε, ε, κανόνες. Θα ήθελα να μου πούν λοιπόν τα συνδικάτα την άποψή τους, γιατί τα εμπόδια που βλέπετε εσείς ε, υπάρχουν και σε άλλα επίπεδα εφαρμογής των ισχυών των κανόνων. Οπότε θα ήθελα μία ακόμη φορά να επαναλάβω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και πρέπει να συμφωνήσω τώρα με τον κύριο Ρούντεμπεργκ. Δεν μπορούμε να μην κάνουμε τίποτα, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με παράνομους εργαζομένους και να μην δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους ε, που νομίμως θέλουν να εργαστούν να εργάζονται. Κυρία Χέντς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως στα σημαντικά σχόλια που έκαναν τα συνδικάτα, ο εκπρόσωπος των συνδικάτων. Είναι ένα ζήτημα δύσκολο. Είναι δύσκολο να υπάρχει εναρμόνιση και, κατα... και κατηγοριοποίηση των εργαζομένων. Μία ερώτηση προς την κυρία Χόφμαν. Εσείς πώς ορίζετε τους ε, εποχιακούς. Κατά τη γνώμη σας, τι θα πει εποχιακός εργαζόμενος, ποιος θα ήταν ο δικός σας ορισμός, πόσο διευρύνεται τη χρονική διάρκεια ας πούμε. Επίσης είπατε ότι οι εργοδότες δεν θα έπρεπε να είναι υπεύθυνοι για τη στέγαση, για την παροχή στέγασης. Ποιος θα έπρεπε λοιπόν να είναι υπεύθυνο. Και αν δεν είναι ο εργοδότης, ποιος θα είναι. Και τρίτον, ποια είναι η θέση σας και ποια είναι η θέση της οργάνωσης που προσωπείτε για το θέμα των μισθών και της ίσης αμοιβή. Νομίζετε ότι έχει νόημα αυτό ή δεν έχει. Και κυρίως σε σχέση με τους εργαζόμενους που μένουν ε, στη χώρα εργασίας τους. Ο κύριος Μωράης. Ναι, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για, το, προς την κυρία Μεσίνα για να τονίσω αυτό που το θέμα που έθεσε η κυρία Ρομέρο Λόπεθ, το θέμα δηλαδή του κατά πόσο φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση, πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση, πώς φτάσαμε. Και το είπα κάπως στην αρχή της συνεδρίασης, δεν ήταν η έλλειψη της διαβούλευσης ε, των κοινωνικών εταίρων, αλλά είναι, από τις, είναι λόγω της φύσεως ε, τη νόμιμη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κοινή μεταναστευτική πολιτική, την οποία ξεκινήσαμε το, την οποία θέλαμε για το 1999 δεν έγινε εγκαίρος, ε, υπήρχαν πολλές καθυστερήσεις ε, και δεν υπάρχει ιδιαίτερη πρόοδο σε σχέση με την κοινή ε, μεταναστευτική πολιτική και πολιτική ασύλου. Άρα λοιπόν κάθε φορά κατηγορούνται οι πολιτικοί, οι, οι υπουργοί ε, και Και θα ήθελα να επικεντρωθώ κυρίως ε, σε, μία συγκεκριμένη, ε, σε, ένα σε συγκεκριμένο θέμα της ίσης μεταχείρισης. Για όλες τις κατηγορίες θέλουμε να ασχοληθούμε με το θέμα της εκμετάλλευσης των εποχιακών εργαζομένων και αυτό δεν είναι θέμα μιας πολιτικής ομάδας, είναι όλοι σύμφωνοι. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, δεν θέλουμε να έχουμε κοινωνικό dumping, δεν είναι μόνο ζήτημα έλλειψης ε, διαβούλευσης, αλλά είναι ένα πρόβλημα γιατί το Συμβούλιο δημιούργησε ένα ολόκληρο χάος στις διάφορες συνεδριάσεις του ε, για την ενιαία άδεια, για την μπλε κάρτα, για όλη τη διαδικασία ε, και πρέπει να δούμε κατά πόσο η μπλε κάρτα εφαρμόζεται όντω ε, σωστά από τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από του συναδέλφου από τα συνδικάτα να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα τη ε, κυρία Ροπέρο Λόπεθ, γιατί είπατε κι εσεί ότι χρησιμοποιείτε πολλού εποχιακού εργαζόμενου. Αν έχουν βελτιωμένα δικαιώματα, ποια θα είναι η σχέση μεταξύ των συνδικάτων και των εποχιακών. Θα είναι ένα ζήτημα πρόσληψη εργαζομένων, είναι η σχέση, εν πάση περιπτώσει, και ποια είναι η σχέση τώρα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ε, θέλουν και εκείνοι να έχουν δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μωράες ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις ερωτήσεις και για τη συνεισφορά σας. Τώρα θα δώσω το λόγο και πάλι στους ομιλητές. Ένας-ένας θα πάρουν το λόγο. Αλλά παρακαλώ να σας ζητήσω μία ακόμη φορά να είστε συγκεκριμένοι, να επικεντρωθείτε σε ερωτήσεις που σας ετέθησαν Πρώτα ο κύριος Σοριάνο. Ε, Ακούστε, όπως είναι λογικό, σε μια παρέμβαση των 2, 5 ή 7 τέλο πάντων λεπτών, μια οργάνωση όπως η ΕΤΟΚ, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων, πρέπει να εκθέσει πρώτα απ' όλα τις αρχές της. Και από εκεί και πέρα να πει κάποια πράγματα τα οποία είναι συνεπή με τις αρχές και τις πρακτικές. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στα πρακτικά θέματα από, την πρώτη, από το πρώτο λεπτό αν δεν έχουμε πρώτα εκθέσει τις αρχές μας και βασική η αρχή μας για αυτό το θέμα είναι ότι θα επιθυμούσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο το θέμα της εποχιακής εργασίας να αντιμετωπιστεί για όλους. Όχι μόνο για τους ξένους, όχι μόνο για τους αλλοδαπούς, εγώ ζήσα στην ε, χώρα σας 7 χρόνια κυρία Σαρτζεντίν και ε, είδα ότι υπήρξαν πάρα πολλές αντιπαραθέσει με Ισπανούς εργάτες που έρχονταν στη χώρα σας να εργαστούν εποχιακά διότι δεν υπήρχε ρύθμιση της εποχική εργασίας και τελικά λείπουν μηχανισμοί που να εγγυώνται την εφαρμογή των δικαιωμάτων και του δικαίου σε κάθε χώρα. Και νομίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν περισσότερα στοιχεία ελέγχου για τους εποχιακούς εργαζόμενους. αλλοδαπούς και μη. Γίνεται λόγος αυτή τη στιγμή στην Ισπανία συγκεκριμένα που έχουμε μια διαπραγμάτευση αυτόν τον καιρό για το θέμα της ε, αδήλωτης εργασίας, της μαύρης εργασίας ε, συγκεκριμένα. Αλλά εγώ θα ήθελα αυτή η συζήτηση να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βέβαια γι' αυτό χρειάζονται πόροι. Και αυτό που δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι ούτε η Ευρώπη ούτε τα κράτη θέλουν να βάλουν ούτε και ένα ευρώ παραπάνω για αυτή τη δραστηριότητα. Ας μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν θα ανοίξουμε την πόρτα για να μπουν στην Ευρώπη εργαζόμενοι τρίτων χωρών χωρίς να υπάρχει εγγύηση ότι όταν έρθουν αυτοί οι εργαζόμενοι θα μπορούμε να του εγγυηθούμε μια αξιοπρεπή μεταχείριση για να μην πω ίση, ισότιμη με όλους τους υπόλοιπους. Αυτή είναι η βασική μας ανησυχία. Δεν μα ανησυχούν οι αλλοδαποί εργαζόμενοι. Τα συνδικάτα μα έχουν πάρα, ε, ε, πάρα πολλά μέλη από του. Ε, από ξένε χώρε. Και έχουμε στι 28 του μήνα στην Ευρωπαϊκή Συνοσπονδία Συνδικάτων μια ε, συνάντηση και σα προσκαλούμε ε, σε αυτήν που ε, θα συζητήσουμε διάφορα θέματα και όχι μόνο με αλλοδαπού εργαζομένου. Θέλουμε να δούμε αυτοί που δεν έχουν χαρτιά, που δεν διαμένουν νόμιμα. Πρέπει να προσπίσουμε κάποια δικαιώματά του και αυτή τη διαχείριση την κάνουμε εμεί από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων. Δεν θα θέλαμε, το είπα και πριν, η οδηγία αυτή να αντιμετωπιστεί ως κάτι που θα αντιμετωπίσει την λάθρο μετανάστευση. Δεν συμφωνούμε. Έχουμε προτείνει κάποιες συναλλακτικέ, δηλαδή άτομα τα οποία έχουν ένα, ε, μια θέση εργασίας, άτομα τα οποία μπορούν να πιστοποιήσουν ότι είναι στη χώρα που ε, διαμένουν και έχουν ρίζες εκεί, ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να νομιμοποιηθούν. Αλλά όχι για την ε, οδηγία αυτή. Να μην είναι αυτή η οδηγία το, η αφορμή. Δεν υπάρχει χρόνος. Ο κύριε Ρούντεμπεργκ, ευχαριστώ. Θα αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Μπουσούτιλ για το πεδίο εφαρμογή. Κάτι είπατε για τους νομίμους και μη νομίμους διαμένοντες εργαζομένους. Ε, το πρώτο που, πρέπει, που θέλω να πω είναι ότι η οδηγία δεν μιλά για δικαιώματα χορήγησης ε, εισόδου ή χορήγησης άδεια διαμονής, αλλά θεσπίζει κάποιους βασικούς κανόνες και μια διαδικασία. Νομίζουμε ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Η οδηγία τώρα απαιτεί να υπάρχει έγκυρη σύμβαση εργασίας. Αν τηρούνται οι κανόνες αυτοί, και να δούμε αυτοί που διαμένουν είναι νόμιμοι ή δεν είναι. Δεν αλλάζει τίποτα μέχρι να εφαρμόσει τη νέα οδηγία για στο κράτος μέλος. Και για να είμαι ειλικρινή, και οι νομίμως διαμένοντες θα κάνουν αίτηση για μια νέα άδεια εποχιακής εργασίας. Οι παράνομα όμως διαμένοντες θα... Και δεν καταλαβαίνω ακριβώς γιατί θα πρέπει να περάσει από αυτή τη διαδικασία ένας ε, εργαζόμενος ε, που είναι παράνομος ή ε, δουλεύει εποχιακά. Δεν υπάρχει βέβαια ε, ουσιαστικά διάταξη λόγος που αποκλίνει να κάνει την αίτηση ένας παράνομος εργαζόμενος, αλλά ουσιαστικά το κράτος μέλος αποφασίζει. Ε, η κυρία Μεζίνα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να τονίσω δύο-τρία σημεία και ενδεχομένω έτσι να απαντήσω και στις διάφορες ερωτήσεις. Για να μην υπάρχει σύγχυση. Όσον αφορά τι συνδικαλιστικέ οργανώσει, ναι, πρέπει να προστατεύσουμε του εργαζόμενου. Αυτό δεν υπάρχει καμία ε, αμφιβολία από αυτού και δεν έχει να κάνει και με την προέλευση του εργαζομένου. Όταν ένα εργαζόμενο απευθύνεται σε ένα συνδικάτο, ε, του συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφέρονται και στου υπόλοιπου. Επομένω, Διαφωνώ με τις υποψίες που υπάρχουν ε, κατά των μεταναστών, των εργαζομένων που μεταναστεύουν. Έτσι λοιπόν εμείς είμαστε μια ομοσπονδία που είναι πολύ μακριά από τις συντεχνίες. Συντεχνίες είναι κάτι τελείως ε, διαφορετικό εμείς πάντα ήμασταν σε αντιπαράθεση με τις συντεχνείς και το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Κατόπιν όσον αφορά στην κατάσταση που προσπάθησα και προηγουμένως να σας παρουσιάσω δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι εργαζόμενοι που ήδη βρίσκονται στο έδαφος των κρατών μελών και είναι παράνομοι. Εδώ λοιπόν υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί μια ουσιαστική σύγκρουση με την οδηγία και με τις δεσμεύσεις που προσβλέπει η οδηγία. Γιατί γνωρίζουμε ότι στη δική μας την αγορά εργασίας οι συμβασιακές ε, σχέσεις είναι πάρα πολύ ανασφαλείς, ε, ο χρόνος δεν ορίζεται. Είναι πολύ δύσκολο ε, να μπει κανείς σε μια κανονική σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Έτσι λοιπόν

οι εργαζόμενοι αυτοί είναι σαφές ότι προσπαθούν να αποκτήσουν μια σταθερότητα αλλά αυτοί με την οδηγία αυτή θα αντιμετωπίσουν περισσότερα προβλήματα. Όσον αφορά τώρα εκείνους που είναι νόμιμοι, ε, ο κύριος Κονφεράτη είπε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος η οποία θα επιτρέψει τη νομιμοποίηση των εργαζομένων εκείνων που εργάζονται παράνομα δυστυχώς ως εποχή εκεί εργαζόμενοι. Τέλος, όσον αφορά αυτή τη ρεαλιστική ερώτηση που μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι από και ως εκ τούτου η ερώτηση είναι σαφώς ρεαλιστική. Υπάρχει μία αντίφαση, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά εγώ βλέπω να υπάρχει μία αντίφαση που ε, διέπει την ε, ευρωπαϊκή πολιτική. Γίνεται λόγος για την κυκλική μετανάστευση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, και σε επίπεδο κρατών μελών όσον αφορά τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μας τις διμερείς ε, συνθήκες ε, και ε, συμβάσεις που συνάπτονται. Είναι σαφές λοιπόν ότι κάποιος που βρίσκεται σε ευρωπαϊκό έδαφος πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσει στο μέλλον να επανέλθει στη χώρα του προέλευσης. Κατόπιν τούτου σας λέω υπάρχει μία αντίφαση εδώ με την ανακοίνωση που έχει γίνει με την έννοια ότι αναφέρθηκε μία από τις αρχές που ενέπνευσαν ε, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι η κυκλικότητα. Ε, εξάλλου, εμείς εδώ στο οχυρό της Ευρώπης είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσουμε για την ποιότητα που πρέπει να έχει ένας μετανάστης που θέλουμε να μπει εδώ. Γιατί αν το κάνουμε αυτό θα είμαστε απλά υποκριτές. Κατ' ουσίαν ξέρετε ποια μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρουν εκείνοι που κάνουν τις ε, βρώμικες δουλειές, ε, τις ε, δουλειές που οι εργαζόμενοι των πλούσιων ευρωπαϊκών χωρών δεν επιθυμούν πια να κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι ε, θα δημιουργηθούν πολιτικά προβλήματα στα κράτη-μέλη. Κατόπιν τούτου εμείς ε, προτιμούμε να ε, μιλάμε για, για τις προϋποθέσεις που θα διέπουν την εργασία των μεταναστών και να μην δημιουργήσουμε και μια δεύτερη οδό που θα επιτρέψει, όπως σας είπα, να υπάρχουν παρεξηγήσεις. Η κυρία Χόφμαν. Um, Ευχαριστώ. Θα επανέλθω στα ερωτήματα που έθεσε η κυρία αλλά Υπάρχουν δύο θέματα που θα ήθελα να σχολιάσω. Πρώτα απ' όλα, και συμφωνώ με όλα όσα υπόθηκαν σήμερα το πρωί για το στόχο της οδηγίας που είναι να υπάρχει μια περιεκτική προσέγγιση για την μετανάστευση και πρέπει να είμαστε και ρεαλιστικοί παράλληλα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, τις απόψεις διαφόρων ε, εταίρων ε, και για τους εργοδότες ε, και για τους ε, εργαζόμενους. Για το ζήτημα λοιπόν της στέγαση συμφωνούμε με την αρχή δηλαδή να υπάρχει κατάλληλη στέγαση αλλά δεν θα πρέπει να είναι υποχρέωση του εργοδότη. να προβλέψει κάτι τέτοιο. Και φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί μπορούμε να συζητήσουμε δηλαδή ποιο είναι ο καλύτερος τρόπος για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Τώρα όσον αφορά τη μη διάκριση. Βεβαίω εμεί είμαστε υπέρ τη μη διάκρισης. Υποστηρίζουμε την αρχή της ίση μεταχείριση, όπως αναφέρεται στην πρόταση και είναι αυτονόητο ότι οι εργαζόμενοι που έρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν τα ίδια κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα με τους ε, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα έπρεπε να ε, την χάνουν ε, διακριτικής μεταχείρισης βάσει της εθνικότητάς τους ή οποιοδήποτε άλλο κριτηρίου. Έχουμε ακόμη και ένα τρίτο πάνελ και νομίζω ότι θα έπρεπε να περάσουμε αμέσω στο τρίτο αυτό πάνελ γιατί Μέχρι τις 12.30 έχουμε προβλέψει χρόνο. Καλωσορίζω λοιπόν τους επόμενους ομιλητές, το επόμενο πάνελ και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους προσκεκλημένους του δεύτερου πάνελ. As I Όπως είπα, έχουμε ένα τρίτο πάνελ. Part of this morning session of the... Έχουμε και ένα τρίτο τμήμα της σημερινής μας συνεδρίασης που είναι αφιερωμένη στον, στους εποχιακούς εργαζόμενους, διεθνείς οργανισμοί και κοινωνία των πολιτών με συμμετοχή διεθνών οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων που εργάζονται με ε, μετανάστες εργαζομένους. Θα ακούσουμε λοιπόν τις απόψεις τους για το της εργασίας του γιατί Έχουμε καλέσει τον κύριο Χέμινουέι, περιφερειακός αντιπρόσωπος του Διεθνού Οργανισμού Μετανάστευσης. Καλώς ήρθατε. Μετά. Εκπρόσωποι δύο μη κυβερνητικών οργανώσεων, της Solidar, την οποία εκπροσωπεί κύριος Ρόιτερ. καλώς ήρθατε, και της Picum από την, με την εκπροσώπηση από την κυρία ε, Λεβουά. Καλώς ήρθατε. Πέντε λεπτά παρακαλώ ο καθένας για να έχουμε μετά συζήτηση και λίγο χρόνο για να συνοψίσει ο συγητής μας ο κύριος Μωράες. Πρώτα ο κύριος Πέρντ Hemingway, που είναι ο περιφερειακός αντιπρόσωπος του Διεθνού Οργανισμού Μετανάστευσης. Έχετε το λόγο. Um, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι και μετέχοντες. Είναι τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ σήμερα και είμαι ευγνώμων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσκληση που μου απίφτεινε να συμμετάσχω σε αυτή την ακρόαση και χαίρομαι πάρα πολύ που μου προσφέρεται η ευκαιρία να ε, συμμεριστώ μαζί σας τις απόψεις μας ε, και την τοποθέτησή μας πάνω στην οδηγία. Εμείς χαιρετίζουμε ε, το γεγονός ότι όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρξει βελτίωση της νομοθεσίας. Θεωρούμε ότι έχει φτάσει πλέον η στιγμή ε, να υπάρξει ένα θετικό μήνυμα προς εκείνους τους μετανάστες εργαζόμενους, ε, τους οποίου προσελκύσαμε εμεί, Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2010, του Δεκεμβρίου 2010, ζήτησε να υπάρχει μια καλύτερη μεταναστευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη και το δημογραφικό πρόβλημα, ε, γιατί αυτό δεν αφορά το απότερο μέλλον, είναι κάτι το οποίο ε, αφορά τις ε, γενιές με έντονη ε, εμφάνιση στην αγορά εργασία, οι οποίοι σύντομα θα βγουν στη σύνταξη. Έγινε μία μελέτη για, τις, για την ομοθεσία στα 27 κράτη-μέλη και ε, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία μεγάλη διάσταση απόψεων. Βέβαια, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι πολλές φορές επειδή υπάρχει μια, μια ε, ε, ε, άκαπτη νομοθεσία ε, δημιουργούνται προβλήματα και για τους εργοδότες και για τους εργαζόμενους. Κατόπιν τούτου οφείλουμε να δούμε πώς μπορούμε να καλύψουμε ε, και τη ζήτηση που προκύπτει, αυξανόμενη ζήτηση που προκύπτει κατά καιρούς. Το να επιτευχθεί λοιπόν συμφωνία ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη ε, για κοινέ προδιαγραφές ως προς την μετανάστευση και κυρίως για την είσοδο και την παραμονή των μεταναστών εργαζομένων, αυτό παραμένει ένας σημαντικός και φιλόδοξος φιλόδοξους στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οδηγία για τους εποχιακά εργαζόμενους ε, προβλέπει μια κοινή διαδικασία και δικαιώματα για τους εργαζόμενους αυτούς. Μία ε, συνεκτική προσέγγιση για όλες τις κατηγορίες των μεταναστών όπως έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό βέβαια θα ήταν προτιμότερο, όμως διαπιστώνεται επικάλυψη ε, της ε, τρομοθετικών διατάξεων σε διάφορες κατηγορίες. Εμείς θεωρούμε ότι εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το πρώτο βήμα για να συμφωνήσουμε σε περισσότερο ευέλικτες διαδικασίες νόμιμης μετανάστευσης. Η δική μας η έρευνα για τους εργαζόμενους με ελάχιστα προσόντα που έρχονται αυτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέδειξε ότι εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε αλλοδαπούς εργαζόμενους συμπεριλαμβανομένων και αυτών με πολύ λίγα προσόντα έτσι ώστε αυτοί να κάνουν τη δουλειά που δεν επιθυμεί να κάνει ο γηγενής πληθυσμός. Βέβαια, Δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται σωστά το θέμα της ε, προσέλκυσης εποχιακών εργαζομένων από τις ε, τρίτες χώρες. Και για το λόγο αυτό διαπιστώνεται αύξηση της ε, παράνομης μετανάστευσης και της παράνομης απασχόλησης με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα για την κοινωνική και την φορολογική πολιτική. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ρύθμιση του θέματο τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η προτινόμενη λοιπόν οδηγία αναγνωρίζει τη διαρθρωτική ανάγκη εποχιακή εργασία στι οικονομίε ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και ε, προσπαθεί και να καθορίσει το νομικό καθεστώ του εποχιακού εργαζόμενου. Αυτό είναι πολύ μεγάλη σημασία γιατί οι εποχιακοί εργαζόμενοι είναι οι περισσότερο ευάλωτοι στην ευρωπαϊκή αγορά εργασία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αδιαφανεί διαδικασίε που πολλέ φορέ συμβάλλουν στο να καθίστε οι μετανάστες εργαζόμενοι περισσότερο ευάλωτοι. Οι εποχιακά εργαζόμενοι και οι προσωρινώς εργαζόμενοι πολλές φορές εξαρτώνται πλήρως από τον εργοδότη ως προς το νομικό τους καθεστώς. Σε μάλιστα περιπτώσεις μάλιστα οι άδειε εργασίες ε, δίδονται στον εργοδότη και όχι στον ε, υπήκο της ε, τρίτης χώρας. Ε, βέβαια αυτό εμποδίζει τον εργαζόμενο να αλλάξει εργοδότη όπως προτείνεται από την οδηγία και αυξάνεται ο κίνδυνος ε, ε, εκμετάλλευσης. Εξάλλου παρεμποδίζεται και η κυκλική μετανάστευση. Πέρα από αυτό, η οδηγία περιλαμβάνει διάφορες ασφαλιστικές δικλίδες, όπως την υποχρέωση του εργοδότη να διασφαλίζει την σωστή αξιοπρεπή διαβίωση, και την ε, παραλαβή καταγγελιών. Η κυκλική μετανάστευση δεν είναι η τελική λύση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Έχει προβλεφτεί η λύση αυτή έτσι ώστε να προκύψουν περισσότερα ωφέλη τόσο για τις χώρες προέλευσης όσο και για τις ε, χώρες προορισμό. Η μετακίνηση των εργαζομένων μπορεί να συμβάλλει στις χώρες προέλευσης να υπάρχει καλύτερη εκπαίδευση των εργαζομένων. Το γεγονός ότι οι μετανάστες ενδεχομένως να έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως εποχιακοί εργαζόμενοι, τούτο αντιμετωπίζει το ε, εξή πρόβλημα, ότι πολλές φορές ε, οι εργαζόμενοι δεν ε, μετακινούνται στην αγορά εργασίας για την οποία καταρχήν είχε προβλεφτεί. Έχουμε πολλές προκλήσεις ε, που αφορούν στο πρόγραμμα κυκλικής ε, μετανάστευσης. Ε, μία εξ αυτών είναι ότι πρέπει να διασφαλίζεται το μεταβατικό στοιχείο που προβλέπεται στην οδηγία. Ε, διαφάνεια επίσης. Οι ίδιοι μετανάστες πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένοι από την αρχή και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έτσι ώστε και οι προσδοκίες τους να είναι ρεαλιστικές. Εδώ ε, πρέπει να υπάρχει σωστή συνεργασία ανάμεσα στα Υπουργεία και ανάμεσα στα κράτη. Επίσης θα ήθελα ε, στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω και το σημαντικό ρόλο των υπηρεσιών δημόσιας απασχόλησης όπως επίσης και τον ρόλο των ιδιωτικών φορέων. Να υπογραμμίσει τον ρόλο των δημόσιων και των ιδιωτικών φορέων τόσο στη χώρα προέλευσης όσο και στη χώρα προορισμού. Επιθυμώ επίσης να υπογραμμίσω ότι η τακτική έλεγχη από τις αρμόδιες αρχές είναι καθοριστική σημασία για να παρεμποδίσουν ε, κατάχρηση κανονισμών ε, από τους εργοδότες. Θα ήθελα να ολοκληρώσω υπογραμμίζοντας ότι η προτινόμενη οδηγία είναι ε, θετική συνεισφορά διότι προβλέπει την επιτάχυνση των διαδικασιών και προβλέπει και ένα νομικό, νομικό καθεστώς για τους εποχιακά εργαζόμενους. Με τον τρόπο αυτό ε, θα διοριστεί το ευάλωτο στοιχείο που χαρακτηρίζει τους μετανάστες εργαζόμενους. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Ρόιτερ ε, από τη Σολιντά και θα σας είμαστε ευγνώμονες ε, αν μπορείτε να τηρήσετε χρόνο. Άρα, περάσω στα συμπεράσματα αστείευομαι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω που μας ε, προσκαλέσατε. Εγώ δεν προεδρεύω, ε, απλά συμμετέχω και θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν ήδη. Δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα συνεργαζόμαστε μαζί με μια συμμαχία μη κυβερνητικών οργανισμών. Έχετε ένα έγγραφο έξω, δεν θέλω να επαναλάβω τα πράγματα. Η προστασία των πολιτών έχει ένα πολύ σημαντικό στόχο Θέλουμε να εργαζόμαστε συμπληρωματικά με τα συνδικάτα σε ό,τι αφορά την αγορά εργασία, τι ανησυχίε αφενό. Αλλά σε ό,τι αφορά αφετέρου την ιδιαιτερότητα των μη κυβερνητικών οργανώσεων, εμεί εργαζόμαστε με ευάλωτε ομάδε. Δεν μου αρέσει και πολύ ο όρο, αλλά ευάλωτε ομάδε είναι οι ομάδε που είναι ακάλυπτε, αν θέλετε. Δεν είναι ενταγμένε σε προγράμματα κοινωνική προστασία, κοινωνική ασφάλιση Κάποιοι μιλούν για λατρομετανάστες, αλλά δεν μου αρέσει ο όρος γιατί είναι και ε, κάποιοι που δεν, δεν εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Απλά δεν είναι τακτοποιημένη η κατάστασή τους, θα έλεγα. αν οι εποχιακοί εργαζόμενοι τώρα δεν εντάσσονται σε βάλλοντε ομάδε, τότε ποιοι εντάσσονται. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σα και την Επιτροπή Απασχόληση για το έργο που έχει επιτελέσει. Ο Κλοντ Μωράη, ο Σέρτσο Κοφεράτη, οι συνεισηγητέ έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε. Δεν είναι η ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών. Αυτή είναι μια ε, πραγματικότητα πολυπρόσωπη. Στη Στοκχόλμη ε, ε, μιλάμε και για τις διάρκειες σχολής κτλ. Αλλά το πρόβλημα το βασικό είναι πώς θα μεταφέρουμε στην πράξη κάποιες καλές έννοιες και θεωρίες και την συγκεκριμένη πρωτοβουλία την καλωσορίζουμε γιατί νομίζουμε ότι είναι ένας τρόπος να προστατεύσει άτομα τα οποία και θα είναι και θα συνεχίσουν να είναι. Η Frontex δεν πρόκειται να χτίσει ε, στη Μεσόγειο τύχη. Θα έρχονται λοιπόν οι μετανάστες. Ε, αυτή είναι μια πραγματικότητα και έχουν πολλούς λόγους. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες ε, που και πουλ όπως λέμε που πιέζουν αυτούς τους ανθρώπους. Θα έρχονται λοιπόν. Άρα τι θα τους πούμε, δεν σας θέλουμε ή θα τους πούμε, θα σας φροντίσουμε. Και είναι μια πολιτική πρόκληση αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς βλέπουμε τι γίνεται. Ε, το είδαμε. Είδαμε πόσο αδύναμη είναι η κατάσταση των βάλει ομάδων. Αλλά βλέπουμε και κάποιε πολιτικέ επιπτώσει. Δείτε τι εκλογέ στη Φινλανδία, δείτε τι έγινε στι κάτω χώρε. Ε, οι δεξιοί εξτρεμιστέ και τέτοιου είδου πολιτικέ ομάδε ε, εποφελούνται από το ότι δεν βοηθάμε κάποια άτομα να είναι σε μια πιο ξεκάθαρη κατάσταση. Άρα, τι θέλουμε. Αφενός πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη για την οδηγία αυτή και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θα πει προστασία, αλλά και άλλες πτυχές πρέπει να καλυφθούν για την αγορά εργασίας. Ας αναφέρω δύο-τρία πράγματα. Νομίζω ότι πολλές φορές αναφέρθηκε ποιες είναι οι προϋποθέσεις εισόδου. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτές, εισόδου και αποδοχής. Ναι, μιλάω γρήγορα, αλλά έτσι έχω πολύ μεγάλη, ακόμη και αυτή την ώρα ε, είμαι πολύ Λοιπόν, να κάνω λίγο τάιτσι. Λοιπόν, ποιος θα είναι αρμόδιος. Αυτοί που καλούν αυτούς τους εργαζόμενους είναι αρμόδιοι κατ' Και ποιοι, κάνουν, ποιοι δίνουν τα στοιχεία. Μπορεί κάποια συνδικάτα, κάποιες ενώσεις να δίνουν ε, πληροφορίες πριν εισέλθουν εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστό είναι αυτό, αλλά τι είδου πληροφορίε πρέπει να δίνουμε, τι είδου μεταχείριση, τι είδου βοήθεια πρέπει να εξασφαλίσουμε για του ε, ανθρώπου αυτού. Άρα, το πρώτο βασικό, ποιο είναι υπεύθυνο, ποιο είναι αρμόδιο. Μία προπόθεση λοιπόν είναι να υπάρχει μία τακτική, μία νόμιμη, ε, ένα συμβόλαιο εργασία νόμιμο, γιατί ετέθηκε το θέμα του κοινωνικού dumping και έγκαιρα είναι τα συμβόλαια τα οποία διέπονται από τι αρχέ ε, του εργατικού δικαίου και τα δέχονται και οι δύο πλευρέ. Και ο εργοδότη και ο Απασχολούμενο. Επίσης είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο ρόλος των μεσαζόντων, γιατί υπάρχει μια γκρίζα αγορά πολύ μεγάλη και εκεί υπάρχει ε, εκμετάλλευση. Είναι η λεγόμενη παραοικονομία και αν αυτή η οδηγία βοηθήσει να βγούμε έξω από αυτή την παραοικονομία αυτή την κρίζα ζώνη, τότε κάτι μπορεί να γίνει. Και υπάρχει βέβαια και ένα άλλο θέμα τη ισότιμη μεταχείριση. Ακούσαμε από τα συνδικάτα τι έχουν να πούν, ακούσαμε και οι εργοδότε τι έχουν να πούν. Η ισότιμη μεταχείριση δεν αφορά μόνο ε, το ίδιο το εργασιακό κομμάτι, ξεκινά από εκεί, αλλά η εργαζόμενοι αυτοί. Είναι ανθρώπινα όντα που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα δικαιώματα. Και πρέπει να έχουν πρόσβαση και σε κάποιου συστήματα κοινωνική προστασία. Δεν μπορούμε να του πούμε ναι, είστε εδώ, αλλά δεν θέλουμε να σα φροντίσουμε, να σα αναλάβουμε, γιατί είναι άνθρωποι και αυτοί. Έχουμε κοινωνική ευθύνη να του συνδράμουμε. Το θέμα λοιπόν είναι ότι ναι, πράγματι χρειαζόμαστε αξιοπρεπή εργασία, προγράμματα κοινωνική προστασίας και πρέπει να καταστήσω σαφέ ότι αυτό το οποίο εμεί περασπιζόμαστε και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε τη μετανάστευση με ένα, ένα πραγματικό φαινόμενο, μια πραγματικότητα που είναι η εποχιακή εργασία και η εποχιακή μετανάστευση. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε συγκεκριμένε απαντήσει. Θα σταματήσω εδώ και θα δώσω το λόγο στην συνάδελφό μου, τη Μισελ Λεβουά από την Πίκουμ. Συγγνώμη έτσι που ήμουν έτσι. Είχα ιδιαίτερο ίστρο, αλλά ε, έτσι είμαι. Ευχαριστούμε, αλλά είπατε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και πολλά και γρήγορα. Όπως ε, θα παρατήρησαν και οι διερμηνείς. Λοιπόν, τρίτος ομιλητής, τρίτη ομιλήτρια, η κυρία Μισελ Λεβουά, Διευθύντρια της ΠΙΚΟΥΜ, πλατφόρμα για τη διεθνή συνεργασία με τους, μετανάστες, με τους μετανάστες χωρίς επίσημα έγγραφα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για την πλευρά για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ε, εμείς έχουμε μια κοινή δήλωση που υπέγραψαν πάνω από 10 δίκτυα που συνεργάζονται με τους μετανάστες. Ε, θα σας τη διανύμουμε, απλώς για την ώρα δεν έχουμε, αρκετές, ε, δεν έχουμε αρκετά αντίγραφα. Θα ήθελα να πω ότι πολλές φορές ακούσαμε σήμερα το πρωί ότι είναι μία από τις πρώτες ευκαιρίες που έχουμε σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συζητήσουμε νομοθεσία για τους ε, χαμηλής ειδίκευσης ε, μετανάστες και εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια σημαντική συζήτηση και πιστεύουμε ότι η ίση μεταχείριση είναι μια αρχή που πρέπει να διατηρηθεί. Έχουμε διάφορες απόψεις, έχουμε συμπεριλάβει στην κοινή αυτή δήλωση των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε σχέση με την οδηγία. Πρώτον, τα δικαιώματα των χαμηλόμισθων εργαζομένων, να μην υπάρχει δηλαδή διάκριση μεταξύ ε, υψηλόμισθων και χαμηλόμισθων. Οι εργαζόμενοι είναι εργαζόμενοι άνθρωποι που έχουν δικαιώματα. Ο ορισμός της εποχικής εργασίας, όπως υπόθηκε πολλές φορές, ε, είναι αόριστος και μπορεί να οδηγήσει σε ε, μεγάλη εκμετάλλευση των ανθρώπων αυτών και αύξηση του κοινωνικού ντάμπινγκ. Μία από τις πρώτες συστάσεις μας είναι λοιπόν ότι θα έπρεπε να υπάρχουν ε, οι απαραίτητες προϋποθέσεις ε, για την ε, ύπαρξη εποχιακών με την με, την, με το σεβασμό των δικαιωμάτων τους και τη ίση τους και να υπάρχει και η δυνατότητα καταγγελιών και αποζημίωσης. Το θέμα είναι ποιος καλύπτεται. Για την ώρα η οδηγία καλύπτει μόνο τους ε, ε, εργαζόμενου τρίτων χωρών, του μετανάστε τρίτων χωρών. Το ερώτημα όμως ετέθη. Μήπως θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε στην οδηγία και τους ε, επικόου τρίτων χωρών που διαμένουν ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνω να δούμε και αυτή τη δυνατότητα. Προτείνουμε όμω και στη συζήτηση να συμπεριλάβουμε και την κατάσταση του κάθε τομέα. Υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι που αυτή τη στιγμή δεν έχουν επίσημα έγγραφα και δουλεύουν σε πολύ επισφαλείς συνθήκες. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η οδηγία ως έχει, που δίνει τη δυνατότητα δηλαδή νόμιμης μετανάστευσης για τους εργαζόμενους που το επιθυμούν, ότι ε, θα επιστρέψουν ε, στις χώρες τους μετά την εξάμηνη περίοδο οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη να εργαστούν στην Ευρώπη. Οπότε, όταν δεν υπάρχει καμία επιλογή αλλαγή του καθεστώτο των ανθρώπων αυτών, μήπω υπάρχει ένα κίνδυνο να, δημιουργηθούν, ε, να δημιουργηθεί επιπλέον παράνομη μετανάστευση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν εδώ μετά θα μείνουν εδώ. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη και τα πορίσματα του προγράμματο Κλαντεστίνο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα από τα πορίσματα έλεγε ότι παρά την διάθεση που έχουμε να μειώσουμε την παράνομη μετανάστευση, υπάρχει νομοθεσία που οδηγεί κατά κάποιο τρόπο στην αύξηση της. Άρα υπάρχει μια ανισότητα μεταξύ των στόχων και του αποτελέσματος. Οι περισσότεροι μετανάστευση που έρχονται στην Ευρώπη υπό την οδηγία αυτή θέλουν να το κάνουν νομίμως. Άρα είναι σημαντικό η νομοθεσία αυτή ε, να δώσει αυτή τη δυνατότητα της νόμιμης μετανάστευσης. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη τη δυνατότητα ενός μεταβατικού καθεστώτος για όλους όσους αυτή τη στιγμή δεν έχουν έγγραφα και δουλεύουν σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Μήπως θα μπορούσαν και αυτοί να ληφθούν υπόψη είτε από αυτή την οδηγία είτε από άλλου μηχανισμού. Είναι επίση σημαντικό να δούμε και το θέμα των κυρώσεων. Αναφέρθηκε πολλέ φορέ σήμερα. Η οδηγία προβλέπει κυρώσεις, αλλά θα έπρεπε να έχει έναν πλήρη μηχανισμό, ώστε όσοι την χάνουν εκμετάλλευση να θεωρούνται θύματα. Είναι σημαντικό επίσης ε, και για τη συζήτηση αυτή να ληφθεί υπόψη το θέμα των κυρώσεων για τους εργοδότες. Η μεταγραφή είναι μέχρι τις 20 Ιουλίου του 2011 για την οδηγία αυτή Νομίζω ότι η κυρία Ρομέρο Λόπεθ το έπεθε σε αυτό το θέμα. Να δούμε ένα σύστημα διαχείριση σε σχέση με τι κυρώσει σε γενικέ γραμμέ και για αυτήν την οδηγία αλλά και για τι άλλε οδηγίε. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τι κυρώσει. Ε, γιατί πολλές φορές ε, είναι ο εργαζόμενος ο οποίος επηρεάζεται από την κύρωση και όχι ο εργοδότης. Είναι λοιπόν μια περίπλοκη συζήτηση που πρέπει να γίνει. Πολύ σύντομα τώρα στο πλαίσιο του οικογενειακού βίου τι θα γίνει, γιατί πολλοί άνθρωποι έρχονται εδώ για μία περίοδο τριών ετών ε, περνούν μεγάλο χρονικό διάστημα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν προβλέπεται ένα δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης και είναι κάτι που θα έπρεπε επίσης να συζητηθεί. Και θα θέλαμε να επισημάνουμε και κάτι το οποίο είπε και ο Κόνη αλλά και άλλοι ε, ομιλητές προηγουμένως. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι οικονομικές μονάδες, είναι άνθρωποι. Και γι' αυτό πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση για την οικογενειακή επανένωση και να υπάρχει μια δυνατότητα ε, Αλλαγή του καθεστώτος του από εποχιακή σε κάτι πιο μόνιμο. Το θέμα τώρα της στέγασης. Όλοι γνωρίζουμε νομίζω ότι υπάρχουν πολλέ καταχρήσει που λαμβάνουν χώρα και το θέμα αυτή της ε, στέγαση των ε, εποχιακών εργαζομένων είναι μεγάλο θέμα στην Ευρώπη. Πρέπει να υπάρχει υποχρέωση των εργοδοτών για παροχή στέγαση, αλλά θα πρέπει να αφήσουμε την επιλογή στον εργαζόμενο να δεκτεί ή όχι. Ε, αυτό βέβαια εξαρτάται από το τι ποσό θα πρέπει να πληρώσουν για τη στέγαση αυτή και ακριβώς τι θα πει ορισμό, ποιος είναι ο ορισμός της στέγασης. Ίσως πρέπει να ε, αναβαθμιστεί για να ε, συμπεριλάβει κάποια κοινωνικά και οικονομικά ε, κριτήρια, γιατί υπάρχει ένα διεθνές πρότυπο ορισμού της στέγασης. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λεβουά. τώρα λοιπόν υπάρχει χρόνος για συζήτηση. Ε, η κυρία Ρομέρο Λόπεθ είναι η πρώτη που ζήτησε το λόγο. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος ε, θέλει να πει κάτι ή να κάνει μια ερώτηση. Κυρία Ρομέρο. Ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση με αυτά που είπε ο φίλος από τη Solidar, αυτό νομίζω ότι σκεφτόμαστε και όλοι οι Ευρωπαίοι σε σχέση με αυτή τη εποχιακή μετανάστευση. Λέμε αυτοί οι εργαζόμενοι θα μείνουν στις χώρες μας, θα μείνουν εδώ. Αυτό σκεφτόμαστε. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά εισοδήματος μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και των χωρών προέλευσης, ιδίως αν αυτές είναι κάποια χώρα της Βόρειας Αφρικής ή πιο από πιο μακριά. Και άρα υπάρχει αυτό το θέμα. Στα στενά του Γιβραλτάρ είναι η πιο τεράστια διαφορά εισοδήματος. Αν υπάρχουν λοιπόν τόσο μεγάλες διαφορές εισοδήματος, ε, φυσικά και οι εποχιακοί εργάτες θέλουν να μείνουν γιατί είναι τελείως διαφορετικές προσδοκίες τους, ε, προσδοκίες διαβίωσης. Αλλά θα πρέπει να ξεχάσουμε και την ιδέα ότι εξαρτάται και από την ηλικία κατά την οποία έρχονται στη χώρα μας αυτοί οι εποχιακοί εργαζόμενοι και επίσης την ανάπτυξη των χωρών της Βόρειας Αφρικής που αρχίζει να βελτιώνεται. Και η συνεργασία με τις χώρες αυτές πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί κάποιες χώρες βελτιώνονται και πρέπει βέβαια να τις βοηθήσουμε Πράγματι αυτή η κυκλική εργασία, όταν υπάρχει φορητότητα, αυτή η εποχιακή εργασία, πήγαινε έλα δηλαδή των εποχιακών εργαζομένων, πρέπει να μπορεί να είναι πραγματικότητα. Αν δεν είναι για πάρα πολύ χρόνο. Παραδείγματο χάρη στη Γερμανία, με κάποιε γειτονικέ χώρε μπορεί να γίνει αυτό, γιατί όταν πράγματι έχουμε μια ολιγόχρονη εργασία και όμορε χώρε, αυτό είναι διαφορετικό από το να έχουμε ε, μεγαλύτερης διάρκειας ε, εποχή ή περίοδο ή απομακρυσμένες μεταξύ τους χώρες. Εξαρτώνται λοιπόν πολλά από τις συνθήκες και από τους όρους. Επειδή είναι πολύπλοκο λοιπόν το ζήτημα αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει να το μελετήσουμε σε βάθος για να δούμε τι ακριβώς ε, προσδίδει αυτόν τον εποχιακό χαρακτήρα, πώ ορίζει το εποχιακό χαρακτήρα, και επαναλαμβάνω, συνεργασία με τι χώρε καταγωγή, γιατί κανεί δεν θέλει να φύγει από την πατρίδα του εάν εκεί έχει ευνοϊκέ συνθήκε διαβίωση. Κανένα. Και νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε και αυτό το ενδεχόμενο. Θα ήθελα να ξέρω πόσοι Ισπανοί μετανάστε γύρισαν στην Ισπανία πόσοι παλινόστησαν ίσω τι τελευταίε ε, δεκαετίε ή χρονιέ τη ζωή του. Αν είχαν όμω καλύτερε συνθήκε διαβίωση, να είχαν γυρίσει νωρίτερα. Θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε κάποια στοιχεία. Και για την άλλη τώρα συνάδελφο, μάλλον την τη Πικούμ, σε ό,τι αφορά το μεταβατικό καθεστώ. Από το να είναι παράνομοι να γίνουν νόμοι, από το να ε, είναι μη τακτοποιημένοι να του ε, ε, τακτοποιήσουμε εντό αγωγικών. Νομίζω ότι θα έπρεπε να μελετήσουμε έναν τρόπο ώστε αυτή ότι η σύμβαση εργασία, αυτό το συμβόλαιο εργασία να μπορεί να ανανεωθεί και στη χώρα καταγωγή, στη χώρα προέλευση. Μιλάμε για συντονισμό δηλαδή. Ε, δεν είναι κάτι το αδύνατο και το ανέφικτο. Ε, μελετήθηκε, δεν μελετήθηκε. Ίσως δεν έχει εκδηλωθεί απαραίτητο, ε, το απαραίτητο ενδιαφέρον για τη ρύθμιση όλων αυτών των ορών. Ο κύριος Προτασίεβιτς νομίζω ότι θέλει το λόγο και όλοι οι υπόλοιποι που σηκώνουν τις κάρτες τους. I will be speaking in Polish if you allow me, so please keep your phones on. I mean, okay, maybe in English, because thank you. Λοιπόν, θα μιλήσω αγγλικά. Ε, ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που είπατε, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ε, συνέβαλαν τα μάλα στη συζήτησή μας για τη μελλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη μετανάστευση. Πριν από δύο εβδομάδες ε, ψηφίσαμε στο Στρασβούργο για την έκθεση του κυρίου Προβέρα σχετικά με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό ως ένα παράγοντα για να επηρεάσουμε θέματα μετανάστευσης. Για μένα λοιπόν είναι προφανές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ε, πρέπει να έχει πολιτική μετανάστευση. Ε. Από την άλλη φορά πρέπει να εμποδίσουμε ανθρώπους να έρχονται παράνομα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε σχέση με αυτά που ο κύριος Ρότερ, δεν το κατάλαβα αυτό που είπατε τη διαφοροποίηση ανάμεσα σε ε, παράνομους μετανάστες και αυτούς που δεν έχουν τακτοποιηθεί. Ο... Τι εννοείται, δηλαδή το περιβάλλον παίζει ρόλο ή ο πόλεμος, μα αν υπάρχει πόλεμος αυτοί είναι αιτούντες άσυλο. Όμως αν έρχονται εδώ αναζητώντας εργασία ή καλύτερη ζωή, δηλαδή αν δεν έχουν προσκληθεί και δεν καλύπτονται από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εποχιακή ή όχι εργασία αυτό δεν παίζει όλο αφού όμως ε, έρχονται χωρίς να έχονται προσκληθεί γιατί πιστεύετε ότι είναι μη τακτοποιημένοι σε αντίθεση με παράνομους είναι παράνομοι αυτοί Mrs. Η κυρία Γιώτοβα. Εγώ θα μιλήσω βουλγαρικά και έχω ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Πρώτα απ' όλα όμως ε, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους μιλητές. Ακριβώς όπως και οι συνάδελφοι και εσείς επισημάνατε ότι η πρόταση της Κομισιόν δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε μια νέα νομοθεσία η οποία θα ρυθμίζει γενικότερα την εποχιακή εργασία τόσο τους εποχιακά εργαζόμενους που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και αυτούς από τρίτες χώρες. Ε, πολλοί επισήμαναν την ε, θέση των Πολωνών εργαζομένων. Πιστεύετε λοιπόν ότι αυτή η νέα νομοθεσία θα πρέπει να είναι συμπληρωματική της υπάρχουσας. Ε, πιστεύετε ότι η Κομισιόν πρέπει να καταθέσει μια νέα πρόταση η οποία να προτείνει ένα ευρύτερο πλαίσιο τόσο για υπηκόους Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για υπηκόους ε, τρίτων χωρών ή μήπως θα πρέπει οι δύο αυτές ομάδες ε, να ρυθμιστούν με διαφορετική νομοθεσία. Λοιπόν, ε, τώρα παρακαλώ τους εκπροσώπους του πάνελ να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τέθησαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, και για τις ερωτήσεις. Νομίζω ότι κάπως χάσαμε το θέμα. Η οδηγία αυτή για την οποία συζητάμε δεν έχει ως στόχο να καταστήσει ε, την κατάσταση πιο περίπλοκη. Θα υπάρχει πάντα κάποιος ανταγωνισμός ανάμεσα στην νόμη και την παράνομη μετανάστευση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βρούμε νομοθεσία που να είναι πιο ελκυστική ε, που να καθιστά πιο ελκυστικό το μονοπάτι της νόμιμης μετανάστευσης των εποχιακά εργαζομένων. Θα ήθελα να προβάλλω το πόσο σημαντική είναι η παλινόστηση. Εμείς όταν μιλάμε για πολιτικές επαναπροώθησης, ε, αυτό συνήθως ε, το σχετίζουμε με παράνομους ε, μετανάστες, αυτούς που έχουν εργάζονται παράνομα ή έχουν ζητήσει παράνομα άσυλο. Η αστυνομία παίζει ρόλο στην οικονομική μετανάστευση, πώς μπορεί κανείς να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να επιστρέψουν, ε, πώς μπορεί κανείς να ε, εξασφαλίσει ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα πιστούν να ξανάρθουν στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά. Ε, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, ε, ας πούμε Συμφωνία Γουατεμάλας-Καναδά. Η κάτοικοι της Γουατεμάλας έμεναν στον Καναδά και ξέρετε γιατί τα γύριζαν, γιατί κόστιζε πάρα πολύ. Και δεν ήταν και σίγουροι αν θα μπορούσαν να γυρίσουν. Να υπάρχει λοιπόν κάτι το οποίο να δίνει τη δυνατότητα τους μετανάστες να ε, πηγαίνουν σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε ότι θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει συνεργασία και πρέπει να υπάρχει συνεργασία και ως προς τα ε, κοινωνικά δικαιώματα των ε, μεταναστών. Να μπορούν να τα πάρουν μαζί τους, ε, στην πατρίδα τους αυτό. Θα είναι κίνητρο για να επανέλθουν. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ρόιτερ. Ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβω ότι προ... Ε, ε, ε, ελέγχθη, αλλά θα επανέλθω πάλι σε αυτούς τους παράγοντες pull and push. Στόχος δεν είναι να μείνουν όλοι φυσικά, γιατί υπάρχει το ζήτημα της ταυτότητας που ζει κανείς, οικογενειακοί δεσμοί, τέλος πάντων πολύ καλοί λόγοι που έχει κανείς, που έχει μια πολιτιστική ταυτότητα και κάποιες ρίζες, αλλά η επιλογή πρέπει να είναι επιλογή του ατόμου δεν είναι θέμα διαχείριση μεταναστευτική ροής. Ε, δεν είμαι τόσο σίγουρος. Κάτι άλλο είναι νομίζω. Και ίσως το πρόβλημα της ακρόαση είναι ότι εδώ μιλάμε για ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι μόνο και όχι για το γενικό φαινόμενο. Ή τα γενικά φαινόμενα που τα ανέφερε η κυρία Ρομέρο Λόπεθ. Ας δούμε το παράδειγμα της Βορειοαφρικής. Το θέμα δεν είναι πώς θα ελέγξουμε, αλλά πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση να επενδύσει στη Βόρεια Αφρική και να διατυπώσει προτάσεις για έναν πραγματικό δημοκρατικό μετασχηματισμό προς, ένα δημοκρατικό και οικονομικά βιώσιμο κίνημα, γιατί αυτό δεν είναι ε, ήδη δεδομένο και έτσι για να κάνω και λίγη διαφήμιση στον εαυτό μου θα πάω ε, με άλλες χώρες ε, ε, και από την Ισπανία ε, στο Βόρειο Αφρική για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εκεί. Και αν μπορούμε κάτι να κάνουμε, που δεν είναι βέβαια η σημερινή συζήτηση, ε, δεν έχει αυτό το αντικείμενο, αλλά είναι στο μυαλό μας, το καλύτερο παράδειγμα που μπορεί κανείς να δώσει είναι κάτι το οποίο έρχεται από το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, το μοντέλο κοινωνικής πρόνοιας της Ευρώπης. Ξέρουμε ότι το 3 με 5% του ΑΕΠ των χωρών αυτών θα τους έδινε τη δυνατότητα να έχουν συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Και στις 12.30 ξέρετε η Solidar διοργανώνει ένα θέμα, ένα σεμινάριο με το θέμα αυτό. Ε, δεν είναι θέμα διαχείριση και ελέγχου των ροών, είναι πώς μπορούμε να αντιστρέψουμε τα ρεύμα και να δώσουμε καλά παραδείγματα. Και ένα τελευταίο, ατυπικές συμβάσεις εργασίας. Νομίζω ότι αυτό είναι κλειδί. Αυτό που βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αύξηση της ατυπικής εργασίας αν με ρωτήσατε, ε, ρωτήστε και τη Eurostat αν υπάρχουν στατιστικά. Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε. Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Το μόνο επίσημο στοιχείο είναι από τη χώρα που προέρχομαι, όπου η Γερμανική Ομοσπονδία ε, Συντροφικές μας έδωσε κάποια στοιχεία. Το 45% των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν πρόσφατα στη Γερμανία είναι προσωρινές, από προσωρινά γραφεία. Το 41% είναι ορισμένου χρόνου και μόνο το 15% είναι επίσημες τυπικές, οργάσεις, ε, τυπικές ε, συμβάσεις εργασίας. Αυτά βέβαια τα στοιχεία μόνο από τη Γερμανία. Λοιπόν, πρέπει να δούμε όλα αυτά τα θέματα και βέβαια και το τι είναι ε, illegal και τι irregular. Γιατί δεν είναι το ίδιο. Πίσω από τον όρο illegal, παράνομος, υπάρχει και πολύ διάκριση. Εδώ λέμε ότι δεν είναι κάποιο, δεν έχει τακτοποιηθεί σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο. Όχι ότι είναι παράνομο. Η λέξη παράνομο στιγματίζει, ε, αποκλείει και αποτελεί διακριτική μεταχείριση. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι για καλό και για καλό, ε, καλκό λόγο είναι εδώ, είναι εδώ όμως και πρέπει να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις. Γι' αυτό δεν είναι ουδέτερος ο όρος ε, illegal migration και γι' αυτό προτιμώ το ρόλο irregular migration. Λιβόη. Ευχαριστώ πολύ σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Ρομέρο Λόπετ για μια συζήτηση που έγινε για τις κόρες προέλευσης. Νομίζω ότι τη συζήτηση αυτή πρέπει να τη συνδέσουμε με τις συζητήσεις που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ε, παράτυπη μετανάστευση, αλλά και για την νόμιμη μετανάστευση. Η Επιτροπή Αρμόδια των Ηνωμένων Εθνών ε, θα, γίνει, θα κάνει μια συζήτηση, μια ολόκληρη μέρα, ε, στην σύνοδό της το Σεπτέμβρη και είναι ανοιχτή η πρόσκληση και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπάρχουν και οι χώρες προέλευσης και οι χώρες προορισμού και βασικά ζητήματα που θα συζητηθούν ε, είναι ε, οι μετανάστες και κυρίως οι πιο ευάλωτοι λόγω του καθεστώτος τους. Επίσης, να μην ξεχνούμε τη συζήτηση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το αναθεωρημένο κείμενό της ε, για την μεταναστευτική πολιτική. Για να προσθέσω αυτό που είπε ο Κόνη για τη χρήση του, της παράνομης τις λέξεις παράνομη ή παράτυπη. Irregular ή illegal. Ε, Μα είχαν πει ότι δεν πρέπει να λέμε παράνομη γιατί ακριβώς αυτό σημαίνει κάποια εγκληματική ενέργεια. Αυτό υπονοεί. Και ουσιαστικά Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να λέμε παράνομοι, γιατί δεν μπορεί ένας παράνομος, κάτι παράνομο να έχει βασικά δικαιώματα. Γι' αυτό δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε αυτόν τον ε, ε, όρο. Και είναι επίση πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε για ποιο λόγο κάποιο δεν έχει επίσημα έγγραφα ή είναι παράτυπο. Γιατί μπορεί να είναι για πολιτικούς λόγους, γιατί μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι και μπορεί για αυτόν τον λόγο να μην μπορεί και να επιστρέψει στη χώρα του. Πολλές φορές ε, άνθρωποι που έχουν προβλήματα με τον νομικό τους καθεστώς εργάζονται ως ε, εποχιακοί και το βασικό θέμα είναι να δούμε τη σχέση των αδειών παραμονής με τις άδειε εργασίας. Και πρέπει να περιμένουμε και τι θα γίνει με τα θεμελιώδη δικαιώματα των ε, ε, νομίμως εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που θα το γνωρίζουμε το φθινόπωρο. Πρέπει λοιπόν να δημιουργούμε συνθήκες ε, ώστε να μπορεί ο εργαζόμενος να αποφασίσει αν θα μεταναστεύσει ή όχι και επίσης όταν αποφασίζει να το κάνει να υπάρχει ίση μεταχείριση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Λεβουά. Ήταν ε, πάρα πολύ διαφωτιστικές ε, οι ομιλίες σας και οι παρεμβάσεις σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας και τώρα να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή τον κύριο Μωράες. Ευχαριστώ. Θα μιλήσει και ο κύριος Κοφεράτη γιατί θα είναι ο συνεισηγητής μου για το θέμα αυτό και ενδεχομένως και εκείνος να θέλει να πει ορισμένα πράγματα. Γι' αυτό θα είμαι σύντομο. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω κιόλα. Να ευχαριστήσω και όλους σας για τις παρεμβάσεις γιατί θα έχουμε πάρα πολύ δύσκολο έργο μπροστά μας. Υπήρξαν πολλές ακροάσεις. Η συγκεκριμένη ακρόαση που έχουμε σήμερα έχει πιο συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της ε, πρότασης. Ε. Οπότε και εγώ και ο Σέργιο θα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας για τις επόμενες εβδομάδες. Θα θέλω να ευχαριστήσω και την Ελένη Κόλος, η οποία τώρα περνάει και έρχεται προς το Προεδρείο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό να ευχαριστούμε τον κόσμο πριν διατυπώσει κάτι εγγράφος. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν μαζί μου. Σύντομα λοιπόν ήθελα να πω το εξή. Πρώτον, δεν περίμενα να δω σήμερα το επίπεδο κατανόησης του ζητήματος αυτού. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι καταλαβαίνουν πώς υπήρξε αυτή η τομεακή προσέγγιση, δηλαδή ότι υπάρχει ένα θέμα για τους επογειακούς εργαζόμενους, για τους χαμηλής ειδίκευσης και προέκυψε λόγω της κατάστασης με το Συμβούλιο και της κατάστασης με την ε, ε, μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν βλέπουμε τόσο, τόση χαρά την ε, υπομονή όλων των ομιλητών, καταλαβαίνουν ε, την ε, θέση στην οποία δεν θα θέλαμε να βρισκόμαστε βέβαια. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα πάνελ για όλους τους εργαζόμενους, γιατί αυτό είναι η συμμεταχείριση και θα έπρεπε να είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε κάποιες νόμιμες διόδους, ώστε κάποιοι άνθρωποι να την χάνουν καλής μεταχείρισης, ίσης μεταχείρισης και να υπάρχει κάποιος ρεαλισμός στην πρόταση αυτή. Ο κύριος Κοφεράτη, η κυρία Ρομέρο Λόπεθ ε, είναι μεταξύ των συναδελφών ε, που μιλούν ε, με πολύ εμπεριστατωμένο τρόπο για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, όχι μόνο ότι υπάρχει στο χαρτί. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω και ειδικότερα να ευχαριστήσω και τους ε, ομιλητές του τρίτου πάνελ. Ε, είναι πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μας είπατε. Θα τα λάβουμε υπόψη μας ε, και στη διατύπωση του εγγράφου. Έχω και εγώ δουλέψει σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και θα θέλα ειδικότερα συνεπώς να σας ευχαριστήσω και για την προοπτική σας, την οποία θα τη συμπεριλάβουμε στην έκθεση. Για την ώρα έχουμε απλώς ένα έγγραφο εργασίας, δεν έχουμε την τελική έκθεση. Να ευχαριστήσω και τους κοινωνικούς εταίρους. Ε, θα ήθελα να τους ευχαριστήσω. Έχουμε πολλές φορές συναντηθεί και οι εκπρόσωποι των συνδικάτων και οι εκπρόσωποι του εργοδότες μας έχουν συναντήσει. Και ούτω ή άλλω ε, θα είμαστε σε επαφή μέχρι να γράψουμε και την έκθεση, να διατυπώσουμε την έκθεση. Ήταν πάρα πολύ σαφή η παρατήρηση και τα σχόλιά του. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή που ξεκίνησε με την μπλε κάρτα, μετά συνέχισε με την ενιαία άδεια, με πολύ έντονο τρόπο. Παίρνουμε λοιπόν πάρα πολύ σοβαρά το, την άποψη των κοινωνικών εταίρων και ειδικότερα το άρθρο 16 για την ίση μεταχείριση. Τέλος, για, τα, για τους συναδέλφους που κατάφεραν να μείνουν και ως το τέλος, ήταν πολύ υψηλού επίπεδου η συμβολή των συναδέλφων, γιατί πρόκειται για ένα νομοθέτημα το οποίο δεν ταιριάζει πολύ καλά στις ε, έννοιες που έχουμε στο μυαλό μα για το τι θα έπρεπε να κάνουμε. Η χαμηλή συνδίκευση εργασία, η εποχιακή εργασία, είναι κάτι το καινούριο που επεξεργαζόμαστε. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να έχουμε πολλές, ε, πολύ, πολύ μεγάλη συνεισφορά. Δεν αρκεί ιδεολογία. Έχουμε συγκεκριμένες καταστάσεις να αντιμετωπίσουμε και ελπίζουμε ότι στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα προστατεύσουμε τους εποχιακούς εργαζομένους, θα έχουμε ίση μεταχείριση και θα είμαστε σε μια θέση καλύτερη ε, από ό,τι στο παρελθόν. Να μην κάνουμε κανένα κακό, αλλά να υπάρχει μια γέφυρα για την προστασία των ευάλωτων εργαζομένων και να καταλαβαίνουμε επίσης, να δείχνουμε ότι καταλαβαίνουμε την πραγματικότητα της ύπαρξης των ανθρώπων αυτών. Έχουμε ένα καθήκον συνεπώς προς τους ανθρώπους αυτούς που είναι ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τους δώσουμε μια θέση στο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λάβουμε και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν λάβουμε υπόψη τη συνεισφορά όλων. Και ελπίζω όταν θα δείτε την έκθεση να δείτε κάποιες από τις παρεμβάσεις σας να, να αντικατοπτρίζονται. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Πολύ επικοδομητικό το σημερινό πρωινό, πάρα πολύ χρήσιμη συνεδρίαση. Βγήκαμε πλουσιότεροι νομίζω σε σχέση με τις γνώσεις μας ε, για τους εποχιακούς εργαζομένους αλλά θα μάθουμε ακόμη περισσότερα και θα είμαστε ακόμη πλουσιότεροι το απόγευμα. Πριν λοιπόν ολοκληρώσουμε την πρωινή μας συνεδρία, να πω ότι το απόγευμα θα επαναλάβουμε τις εργασίες μας όχι στις 3, αλλά στις 2. Όχι όπως συνήθως στις 3, αλλά στις 2. 2 με 5 θα είναι η απογευματινή μας συνεδρίαση. Μόνο ένα σάντουιτς θα προλάβουμε να φάμε. Να δώσω και το λόγο στον κύριο Κοφεράτη που είναι εισηγητής της Επιτροπής Απασχόλησης. Εσείς θα έχετε τον τελικό λόγο. Εγώ απλά ε, θέλω να πω ότι όπως και ο συνάδελφος ο Μωράς και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους που έλαβαν μέρος σήμερα το πρωί σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και τώρα έχουμε πάρα πολύ υλικό το οποίο θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νομίζω λοιπόν όπως ελέγχθη επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της συζήτησης είναι ένα πολύ λεπτό θέμα ένα θέμα που καλούμεθα να το αντιμετωπίσουμε γιατί η όλη διαδικασία, οι μεταναστευτικές ροές τρέχουν, ξελίσσονται και συνδέονται βεβαίως με έκτακτες καταστάσεις όπως είναι παραδείγματος χάρη αυτή η κρίση στη Μεσόγειο. Ε, σήμερα μιλήσαμε για μία ψηφίδα ενός περίπλοκου ε, μοσαϊκού και καλούμεθα να ολοκληρώσουμε να τελειοποιήσουμε το μοσαϊκό. Θα αναφερθούν λοιπόν και άλλα επιχειρήματα. Και θέλω να σας πω ότι εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτόν τον τρόπο εργασίας, δηλαδή στην αντιπαράθεση. Γιατί πάρα πολύ συχνά στα έγγραφά μας ε, γράφουμε ότι είναι σημαντική η αντιπαράθεση και αφού τελικά είμαστε πεπισμένοι, γιατί να μην το κάνουμε στην πράξη, να που το κάναμε σήμερα το πρωί. Άρα δηλαδή πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο να δώσουμε συνέχεια σε αυτή την έκθεση, όπου βέβαια ο καθένας θα κάνει τη δική του τη δουλειά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και χρήσιμο πριν καταλήξουμε σε συγκεκριμένα τυπικά στοιχεία να ανταλλάσσουμε απόψεις. Να ανταλλάσσουμε απόψεις σεβόμενος ο ένας τον άλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει όσο πιο πολλά πράγματα παθαίνει κανείς τόσο πιο εύκολη γίνεται η δουλειά του. Ευχαριστώ. Και εμεί ε, σας ευχαριστούμε. Ξεκινάμε λοιπόν όπως σας είπαμε στις 2 σήμερα το απόγευμα και ε, επανερχόμεθα για το δεύτερο ε, πακέτο της μετανάστευσης, ενδοεπιχειρησιακές ε, μεταθέσεις. Ευχαριστούμε όλους που συμμετείχαν και σε αυτό και στο προηγούμενο πάνελ. Σας ευχαριστούμε όλους. Γεια σας.